Είναι η τελευταία ψηφοφορία για ένα σημαντικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τον κώδικα θεωρήσεων. Και ήφιστε πριν την ψηφοφορία στην Ορομέλεια και ενώπιον όλων των μελών να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την επικοδομητική συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους κοιόδης συζητητές στην Επιτροπή Λίμπε, τον πρόεδρο και συνάδελφο Κλοντ Μωράες. Αλλά με δεδομένο ότι αυτή είναι η τελευταία ολομέλεια του Κοινοβουλίου μας, καλό θα ήταν να, και σύνθεση είναι να εκφράσουμε δημοσία την ικανοποίησή μου που μπορέσαμε να υπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες στο σώμα αυτό, το μόνο ερετό δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα αυτής της του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να σας ευχηθώ πραγματικά εκ βάθους καρδίας ό,τι καλύτερο για όλους και να σας πω ότι είναι, ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ όλους σας συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε και εμείς κύριε Λόπες Αγγιλάρ. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πρώτη ανάγνωση ολοκληρώνεται. Έκθεση Ράο Σάντο. Και εδώ ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 82. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται. Προχωρούμε. Έκθεση Ράντεφ. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 73 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ολοκληρώνεται η διαδικασία. Ψηφοφορία για την έκθεση Ρέντα. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρούται έτσι. Έκθεση Βίρκουνεν Μαρινέσκου και Τέλιτσκα. Τροπολογία 108 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές, θα γίνει έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρόταση με ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται. Έκθεση Ντάλτον. Τελειώνουμε με αυτήν. Τροπο, πολλές τροπολογίες της, Επιτροπή, της αρμόδιας Επιτροπής ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία 31 άρχεται η ψηφοφορία. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για το 19. Ωραία. Έλεγχος για το, την τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. 19. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία 31 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Για την 59 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Με ονομαστική ψηφοφορία 63 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67 άρχεται η ψηφοφορία με νομαστική ψηφοφορία πάλι. Πέρας. Δεκτή. 82 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 87. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 105 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ονομαστική ψηφοφορία για το 163 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος για την 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 160. Με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Η 66 υπερψηφίστηκε, άρα πηγαίνουμε στην 160. Ψηφίζουμε την 160 με ονομαστική ψηφοφορία. Πάντα ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 157. Άρχεται η ψηφοφορία. 157. Πέρας. Απορρίπτεται. 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 81. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η επόμενη. 83D με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Προχωρούμε λοιπόν στην 85. Όλες οι άλλες καταπίπτουν. 85 υπέρα. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρη. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Να σηκώνετε το χέρι σας αν γίνεται. 86 γιατί όλες οι υπόλοιπες, Η 175 πέφτει. 86 δέλτα υπέρ, κατά, αποχές. Λυπάμαι αλλά δεν σηκώνονται τα χέρια σας. Θα γίνει λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 86D άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 88. Γιατί έχουν καταπέσει οι προηγούμενες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 165 Ντε, ναι, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Με ονομαστική ψηφοφορία 161. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 162. Άρχεται, πάλι με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Με ονομαστική ψηφοφορία 158. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και 156 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε Δε. υπέρ, κατά, αποχές θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 18η άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 159. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται και η διαδικασία των ψηφοφοριών. Ο κύριος Έκαουτ, ε, θα πρέπει να σταματήσετε τις συζητήσεις με τους συναδέλφους γιατί είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Α, όχι, όχι, όχι. Βεβαίως, ξεκινάμε κατευθείαν. Έχουμε λοιπόν την έκθεση Αϊκάουτ. Μέχρι να πέσουν οι τίτλοι, νομίζω ότι θα ηρεμήσουν και οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά... Α, ναι, δεν έχει έρθει όμως η Επιτροπή. Να περιμένουμε λοιπόν. Euh, Συνάλφοι, ας προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ πολύ όσοι συζητούν στους διαδρόμους ε, ή να διακόψουν ή να συνεχίσουν αλλού. Επίσης οι κλητήρες παρακαλώ να κάνουν αυτή τη δυσάρεστη δουλειά που έχουν που είναι όμως πολύ χρήσιμη. Κύριε Άικαουτ, θα σας δώσω το λόγο. Μια και είναι η σειρά της δικής σας έκθεσης. έκθεση. Ε, πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο, κύριε Άικαουτ. Uh, thank you for all the ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενδιαφέρον που δείχνετε για το διοξιδίτη του άνθρακα και τα φορτηγά, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλά κάνετε και το προσέχετε το θέμα αυτό, γιατί είναι η νομοθεσία την οποία καλούμαστε να εγκρίνουμε στην τρέχουσα θετία. Αυτό τι σημαίνει ότι πέρα από την νομοθεσία αυτή θα κληθούμε να κάνουμε πολλέ βελτιώσει, αλλά εδώ χρειάζεται να γιορτάσουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ρυθμίσει τι του άνθρακα, τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Όπω έγινε και με τα ΙΟΤΑΧΗ, ήταν ε, δύσκολο ο αγώνα. Μεγάλη αντίσταση που αντιμετωπίσαμε. Καταφέραμε, θεωρώ όμω, με καλή συνεργασία με του διάφορου κοιόδε συζητητέ από τι πολιτικέ ομάδε να ευχαριστήσω για τη συμβολή σα και τη συνεισφορά σα. Δεν συμφωνούσαμε πάντα. Αλλά νομίζω ότι σε τελική ανάλυση πετύχαμε μια συμφωνία την οποία όλοι υποστηρίζουμε. Και έχουμε την αίσθηση ότι πραγματικά αγγίζουμε το σημαντικό πυρήνα του θέματο αυτού. Και βλέπουμε λοιπόν μείωση του διοξιδίου του άνθρακα 25% μέχρι το 2025. Μέχρι το 2030 δεσμευτικό στόχο 30%. Και ιδιαίτερα αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική θα δώσει ένα σαφές μήνυμα προς τους αυτοκίνητο παραγωγούς ε, βαρέων οχημάτων ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες. Επίσης, καταφέραμε να κλείσουμε και όλα τα παραθυράκια σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά τις υπερπιστώσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τα υπερπιστωτικά όρια. Και έτσι λοιπόν σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες καύσης, σε ό,τι αφορά την επένδυση σε νέες τεχνολογίες για το μέλλον. Το μέλλον το οποίο μπορεί να αποτελεί και υδρογόνο αλλά και άλλες ε, μορφές ενέργειας. Αυτό λοιπόν είναι μια σαφή ε, καθοδήγηση προς τους παραγωγούς. Ήταν σκληρός ο αγώνας και προφανώ από πλευρά των πρασίνων θα θέλαμε να έχουμε πιο φιλοδοξού στόχου επιτάπητο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει σαφήνεια μακροπρόθεσμη πλέον για του παραγωγού, προκειμένου να ξέρουν πού οδεύουν και πού θα πρέπει να επενδύσουν. Για να εξασφαλίσουν και ότι το μέσο μεταφορών επίση καθαρίζει και κινείται προ την ε, μείωση της χρήσης του άνθρακα, γιατί όταν ρωτάμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κλάδος, να σας πω ότι είναι 6% του συνολικού ε, των συνολικών επενδύσεων, αλλά σε σχέση με τις οδικές μεταφορές μιλάμε για 25% ποσοστό. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ σημαντική κατηγορία η οποία επιπλέον αυξάνεται η σημασία της. Μέχρι το 2050 ξέρουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μειώσει και να έχουμε αφαιρέσει τον ανθρακά από την οικονομία μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή η νομοθεσία. Θα γίνουν αναθεωρήσεις μέχρι το 2022. Να σας ε, υποσχεθώ ότι μέχρι τότε θα κοιτάξουμε και τους στόχους που θα, έχουμε, θα θέσουμε αύριο και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά παραπάνω. Γιατί θα δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, όπως σας είπα αύριο. Και αλλάζει λοιπόν η αγορά. Έχουμε νέε θέσει οι οποίε θα προκύψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πραγματικά ήταν η σωστή στιγμή να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπω ε, άλλε χώρε, ε, μάλλον όπω η Ιαπωνία, η ΙΠΑ, ο Καναδά έχουν ήδη ρυθμίσει το θέμα αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα προσπαθούμε να προλάβουμε αυτές τις χώρες αυτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν την κατάργηση του άνθρακα στον τομέα του μεταφορών αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Είναι λοιπόν καλή η έκθεση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, την Επιτροπή, το Συμβούλιο που απουσιάζει για τη στενή συνεργασία και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο επίτροπο, ο κύριος Κανιέτα. Madam President, honorable members. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα για την τελευταία συζήτηση για αυτό το νομοθέτημα. Η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό επίτευγμα και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ε, φιλόδοξου ε, πλαισίου για την ε, καθαρή ενέργεια για το 2030. Αυτή η συμφωνία κατέστη δυνατή χάρη στις προσπάθειες, επικοδομητικές προσπάθειες και των δύο οργάνων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή τον κύριο Έικαρτ και όλους τους συνεισηγητέ για αυτή την επιτυχία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η συμφωνία η οποία πετεύχθη είναι ισορροπημένη και φιλόδοξη. Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι για τα νέα βαρύ επαγγελματικά οχήματα η, ο μέσος όρος των εκπομπών το 2025 θα είναι 50% χαμηλότερος σε σχέση με τις αυτές του 2019. Τα βαρέα οχήματα αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών εκπομπών των επαγγελματικών οχημάτων. Και ε, ξεκινώντας από το 2019 με τα υπερπιστωτικά μόρια ε, θα μειώσουμε στο 0 τις ε, εκπομπές. Το 2022 θα γίνει μια συνολική επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας αυτής. Αυτό το κείμενο συμπληρώνει την εικόνα. Ο τομέας των οδικών μεταφορών κινείται σαφώς προς, προς μια πιο καθαρή λειτουργία. Τα βασικά ωφέλη είναι ότι οι εκπομπές βαρέων οχημάτων θα αντιπροσωπεύουν το 25% ε, των συνολικών οδικών μεταφορών. Ε, αυτή τη στιγμή θα αυξηθούν κατά 10% το 2030 αν δεν κάνουμε τίποτα. Με τους στόχους μας όμως και με τους ε, μελλοντικού μας στόχους θα μειωθούν κατά 24% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τους ε, συνολικούς στόχους που έχουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του Παρισιού. Επίσης θα γίνουν εξοικονομήσεις ε, ε, από πλευρά των ε, ιδιοκτητών τους. Ε, Ξονομήσεις λόγω φθηνότερου καυσίμου. 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των των μεταφορών που δίνουν δουλειά σε 2 εκατομμύρια άτομα θα βοηθούν πάρα πολύ. Επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία θα ενισχύσει την καινοτομία της και τη, θα διοχετεύσει καλύτερα τις επενδύσεις της. Δίνουμε κίνητρα για, μηδενικό, για οχήματα μηδενικών εκπομπών ε, ενώ δίνουμε το μήνυμα ε, ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, υποδομές επαναφόρτισης. Τέλος, θα αυξηθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη και θα μειωθούν οι εισαγωγέ πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σα καλέσω να στηρίξετε αυτή την συμφωνία αύριο. Θα βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κατεύθυνση τη μετάβαση προ τι καθαρέ μεταφορέ. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει και δύο δηλώσει που ε, προκειμένου να στηρίξει τη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Κοινοβουλίου. Ε, θέλω να ευχαριστήσω μία ακόμα φορά όλα τα μέλη για τη στήριξή τους. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Βίρκουνεν, εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματο τη Επιτροπή Μεταφόρων και να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για το καλό παράδειγμα, ε, για το καλό αποτέλεσμα που πετύχαμε. Από πλευρά τη Επιτροπή ε, Μεταφορών ε, έχουμε να πούμε ότι και η παραγωγή ε, βαρέων οχημάτων θα πρέπει να φροντίσουν για μείωση 25% μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030. Είναι φιλόδοξο ο στόχο, αλλά πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκδίδουμε τέτοιε προδιαγραφέ εκπομπών για τέτοια φορτηγά. Και φυσικά, ω τώρα υπήρχαν κίνητρα για την ε, αποτελεσματικότητα και την αποβατικότητα των οχημάτων και για το κόστος, τη μείωση του κόστους ε, των καυσίμων των φορτηγών. Αλλά με τις διατάξεις αυτές θα προωθηθούν περαιτέρω και οι καινοτομίε στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξουν και μέθοδοι μέτρησης όλες ε, Θα πρέπει να ληφθεί επίση υπόψη η κατανάλωση ενέργεια σε όλο τον ε, κύκλο παραγωγή. Γιατί έχουμε μεγάλο περιθώριο μείωση των εκπομπών στι οδικέ μεταφορέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στι πολιτικέ ομάδε Έχουμε τον κύριο Φιέλνερ από το ΕΛΚΑ. Για δύο λεπτά ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σε... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ολοκληρώνονται πολλά χρόνια δουλειά και για μένα και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Αύριο θα εγκρίνουμε τους κανόνες. Ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Έχουμε καλύτερες μεταφορές χωρίς μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αυτή είναι η τελευταία φορά που απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για 15 πανέμορφα και εξαιρετικά χρόνια. Άρχισα να γκριζάρω νικρό μου όλα αυτά τα χρόνια εδώ και άλλοι και άλλων, αλλά ήταν τιμή μου να εκπροσωπώ τη Σουηδία και το κόμμα των συντηρητικών. Μπορέσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς όφελος του ελεύθερου εμπορίου που βγάζει τους ανθρώπους από τη φτώχεια κάνει πλουσιότερη την Ευρώπη, να βελτιώσουμε το περιβάλλον, φέρνουν τον, φέραμε τον άνθρωπο στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, αλλάξαμε την Σουηδία, αλλάξαμε τα πράγματα και για την Ευρώπη. Μπορεί να μην ήμουν πάντα ένας μετριοπαθής, αλλά πάντα προσπάθησα να προασπίσω την, το σωστό και τους ψηφοφόρους μου γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι κάτι που αξίζει να πολεμήσουμε για την ειρήνη και την κοινότητα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι αυτή είναι η βασική ελπίδα για την οποία πρέπει να δουλέψουμε. Ευχαριστώ. La parole Τζόφολη, δύο λεπτά για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Καλύτερα με το μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει μικρόφωνο κύριε Τζόφολη. Συνεχίζετε να μην έχετε μικρόφωνο. Με ακούτε τώρα. Η, ο κανονισμός που υποστηρίζουμε παρά τα προβλήματα που έχει καθι, ε, ε, ε, φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από πολλές αντιστάσεις κοινά όρια για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα για τα βαριά επαγγελματικά οχήματα που συμβάλλουν κατά 6% στις συνολικές εκπομπές τη Ένωση, εκπομπές που προβλέπεται να αυξηθούν. Πέρα των target στόχων που είναι φιλόδοξοι αλλά μπορούμε να, τα, τους πετύχουμε, έχουμε μια σειρά πρότυπων επιδόσεων στο δρόμο με εκπομπές για την κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αυτά τα πραγματικά στοιχεία συχνά απομακρύνονται από αυτά που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά των εργασιρίων και είναι αναγκαία για να αποφύγουμε στρεβλή συμπεριφορά και τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για ελέγχους, για ανεξάρτητους ελέγχους. Κατά σημαντικό είναι το αίτημα της Επιτροπής μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση ε, ε, των εκπομπών των οχημάτων αυτών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή τους. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ένα μηχανισμό κινήτρων για την διάδοση ηλεκτρονικών φορτηγών ή χαμηλής, χαμηλών εκπομπών για να εξασφαλίσουμε από το 2025 ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό των οχημάτων αυτών ε, στο ύψος του 2%. Θα δοθούν κίνητρα σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και υποδομές για, την ηλεκτρική, για τα ηλεκτρικά φορτηγά. Στην πορεία για την ε, απομάκρυνση από τον άνθρακα, που κατά 94% εξαρτάται ακόμα και τώρα από το πετρόλαιο, θα πρέπει να εξετάσουμε και το ρόλο του φυσικού αερίου. Είναι αναγκαίο ωστόσο η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ταμείο για την ε, ε, πανακατάτηση των εργαζομένων στον κλάδο για να καταστήσουν την βιώσιμη, τη μετάβαση βιώσιμη και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ο κόνισμος αυτός αποτελεί ένα επιπλέον βήμα σε μια Ευρώπη που αλλάζει προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη συμμαχία μεταξύ βιομηχανίας και περιβάλλοντος. Ο κύριος Μάκρη, λεπτό. Αύριο το μεσημέρι έχουμε την τελευταία ε, ψηφοφορία της τρέχουσας και πάλι έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε για συγκεκριμένα μέτρα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι εκπομπές του του άνθρακα για τα φορτηγά είναι ευθύνονται για 6% των συνολικών εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ένα τέταρτο των ε, οδικών μεταφορών. Και αυτές οι εκπομπές αυξάνονται ακόμα και στη δική μου χώρα, στη Φλάνδρα. Θέλουμε, αν θέλουμε λοιπόν ε, να πετύχουμε τους στόχους μας για τις δεσμεύσει μα για το κλίμα, θα πρέπει να πρασινίσουμε τον στόλο μας. Έχουμε την τεχνολογία αυτή. Είναι κρίσιμη σημασία, καταρχά να υπάρξει ένα πρότυπο μείωση του διεξιδίου του άνθρακα για τα φορτηγά και τα κίνητρα για να ενθαρρυνθούν τα φορτηγά χαμηλών εκπομπών. Είναι σημαντικό και γι' αυτό λοιπόν το κόμμα μου το ΕΝΒΑ υποστηρίζει αυτή την τελική νομοθεσία παρά το γεγονό ότι θα θέλαμε πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξία. Το πρασίνισμα λοιπόν του στόλου είναι πολύ σημαντικό για καλύτερη ποιότητα τη ατμόσφαιρα γιατί αυτή προκαλεί θανάτους πρόωρους. Τα πρότυπα αυτά φροντίζουν να υπάρχει και μείωση της, ε, του κόστου των καυσίμων. Αυτό είναι καλό για το καταναλωτή. Και τέλος, ε, η φιλόδοξη αυτή θέση προτύπων ε, χρειάζεται για να προσελκύσουμε επενδύσεις και κοινοτομία. γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο κ. για δύο λεπτά έχει το λόγο από την Άλτα. Πρόεδρε, ξεκινώ ευχαριστώντας τους συντρόφους και συναδέλφους που δούλεψαν μαζί μου αυτά τα χρόνια στις διαπραγματεύσεις. Είχα συνεργαστεί με τον κύριο Άικχαουτ και τον Κρίστο Φιέρνερ. Γκρίζαν τα μαλλιά του, είπε ο κύριος Φιέρνερ, αλλά αν δω τον Επίτροπο ή και εμένα στον καθρέφτη θα έλεγα πολύ περισσότερα γκρίζα μαλλιά έχουν άλλοι. Έχουμε μπροστά μας κάποιες σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, κατακαιρματισμός στην κατασκευαστική διάσταση. Πολλοί κατασκευαστές θα τηρήσουν τους στόχους χωρίς δυσκολία, άλλοι θα το πετύχουν πολύ πιο δύσκολα και θα δυσκολέψουν έτσι τα πράγματα. Άλλο πρόβλημα είναι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως τα λέμε. Το... Τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, αλλά με βρώμικο ηλεκτρισμό, δεν είναι και πολύ καθαρά. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σημαντικούς στόχους, ε, όπως αυτούς που συζητήσαμε χτες με την Κρέτα Τούμπεργκ αν θέλουμε θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι ο δρόμος μπροστά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια γέφυρα για το μέλλον με εναλλακτικά καύσιμα, εξασφαλίζοντας ότι οι εκπομπές, ε, τα όρια των εκπομπών είναι χαμηλότερα από αυτά του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούμε σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση προς τα εμπρός έχει να κάνει με αυτό που είπε στο ξεκίνημα της παρέμβαση, του ΟΜΠΑΣ, την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής τα επόμενα έτη. Μιλάμε τώρα για το επόμενο κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει έτοιμη δουλειά, εξασφαλίζοντας ότι η πρόταση αυτή θα φτάσει στην, ε, τον προορισμό που έχει και ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι θα γίνονται τα σωστά πράγματα. Ο Μπάς και άλλοι που μπορεί να είναι εδώ θα μπορέσουμε αν θέλουμε να βοηθήσουμε την υλοποίηση αυτής της, ε, ε αυτής της κάποιος ε, ζητάνε να δέξει να απαντήσετε μια μπλε κάρτα. Πάντα με χαρά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συναδελφό, τον κύριο Τόρβαλτζη, γιατί το διοξείδιο του ανθρακά προφανώ και αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Και γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δούμε και το κύκλο, σε όλο τον ε, κύκλο παραγωγής των φορτηγών. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και τι γίνεται με τα χρησιμοποιημένα φορτηγά. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα διαρκές ε, τέτοιο ζήτημα στις ε, πόλεις και αυτά θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο το οποίο χρειάζεται δεν είναι τόσο τα ευφύ οχήματα, αλλά κυρίω οι ευφύ οδηγοί. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρει φυσικά ο κύριο Ρούμπι ευφύ οδηγού. Αλλά αυτό χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να μας ε, εκπαιδεύσουν στην οδήγηση. Χρειαζόμαστε τα τεχνικά εργαλεία για να έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο και να μην φοβόμαστε την τεχνολογία και όλες τις ευκαιρίες που παρέχει. Αν δεν φοβόμαστε, θεωρώ ότι μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Εκ. 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Συχνά άσκησα κριτική στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τις αποφάσεις προς όφελος των μεγάλων ομίλων και προς ε, εις βάρος ε, της, του ανθρώπου, των, των ζώων και του περιβάλλοντος. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που πέτυχε ο εισηγητής, ο κύριος Αικχάουτ. Αύριο θα ψηφίσουμε για τον πρώτο κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα φορτηγά. Παρά της μεγάλης αντίδρασης της, του οικονομικού κλάδου και πολλών κυβερνήσεων και κυρίω τη γερμανική κυβέρνηση, αυτή η πρόταση ξεπερνά κατά πολύ την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντο. Δεν επαρκεί, ασφαλώ. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά να κάνουμε σε πολλού τομεί. Σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία αυτή εδώ στην Ολομέλεια. Δεν πρόκειται να είμαι βουλευτή στην επόμενη θετία. Θα σα καλέσω λοιπόν να τηρήσουμε το άρθρο 13 της Συνθήκης Λισαβόνα και να λάβουμε υπόψη την ευημερία των ε, δισεκατομμυρίων ζώων τα οποία τη χάνουν και ε, τα θανατώνουμε, να κάνετε πολιτική με την καρδιά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσετε φυσικά και το κουμπί της λογικής. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πολιτικά παράδειγματα να μην κοιτάμε μόνο την οικονομική ανάπτυξη, να μην είναι μόνο αυτό ο απότερο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ευημερία, η ευτυχία όλων των ε, ζώων, των οργανισμών και των ζώων. Αυτό αναμένουν οι πολίτε από εσά. Αυτό προσδοκούν οι πολίτε από εσά. Σα ευχαριστώ. Να είστε καλά και να έχετε το χέρι στην καρδιά στι μελλοντικέ πολιτικέ αποφάσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Ο κύριος Λίζε, ευχαριστώ πάρα πολύ αξιότιμη κυρία συνάδελφε, κυρία Έξ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον προσωπικά. Έχω μία ερώτηση όμως να σας κάνω παρόλα αυτά. Αυτές τις πληροφορίες, από πού τις έχετε πάρει ότι αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας ξεπερνούν κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ζήτησε και η γερμανική κυβέρνηση 15% και 30%. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχος ο στόχο και δεν ξεπερνά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Σέκα. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι σε κάποια σημεία στις διαπραγματεύσει πετύχαμε στόχους οι οποίοι ξεπερνούν ε, σίγουρα κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το οφείλουμε κυρίως στον πολύ καλό συνάδελφό μα, τον εξαιρετικό συνάδελφό μα τον κύριο Έκα, ο οποίο ε, πολέμησε με νύχια και με δόντια προκειμένου να είναι φιλόδοξη η έκθεση και γι' αυτό θα ήθελα προσωπικά να του απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, Ντέλη, η κυρία Ντέλη έχει το λόγο. Παρακαλώ, Καρύμα. Συνάδελφοι, αυτή την εβδομάδα δεχθήκαμε στο Κοινοβουλίο την Γκρέτα Τούμπεργκ που ήρθε να μας πει αναλάβετε δράση, κάντε κάτι, κάντε κάτι τώρα. Φροντίστε ότι εσείς που αποφασίζετε να επιτρέψετε να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ζήσουν ευτυχισμένες σε έναν φιλόξενο κόσμο. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη και την υγεία μας, θα πρέπει να, και να μειώσουμε την ρήπανση, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να υποχρεώσουμε τον κλάδο των μεταφορών να συμβάλλει όπως οι άλλοι. Στους δρόμους της Ευρώπης 5% ε, είναι μόνο τα φορτηγά μεταξύ των οχημάτων που παράγουν ωστόσο το 27% το 1 τέταρτο δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των οδικών μεταφορών στην Ένωση. Αν θέλουμε μια μέρα να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του COP21 να σώσουμε για να σώσουμε το κλίμα και τον πλανήτη είναι καιρός να σταματήσουμε με αυτή την ανισορροπία. Με το κείμενο που υποβάλλεται ψηφίζουμε και κάνουμε τα πρώτα βήματα για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, λιγότερα ε, ε, αέρια μέχρι το 2000, με μείον 15% για τα φορτηγά. Ο κανονισμός πάει παραπέρα από την πρόταση επιτροπή και για πρώτη φορά δεσμεύει την Ευρώπη να μειώσει την ε, ρήπανση των μεγάλων φορτηγών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι νικήσαμε. Τι δείχνει αυτή η νίκη. Δείχνει ότι όταν εμείς οι ψηφοφόροι Ακούμε τα αιτήματα, ιδίως της νεολαίας, που κάθε εβδομάδα κάνει απεργία για να σώσει το κλίμα. Όταν εγκρίνουμε, ε, όταν περνάμε από τα ωραία λόγια σε συγκεκριμένες δράσεις, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Προσοχή ωστόσο. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την ε, δυνατότητα τα παιδιά μας να ανασάνουν, να ζήσουν ελεύθερα, να χαρούν αυτόν τον ωραίο πλανήτη, θα πρέπει αύριο να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό, γιατί ψηφίζοντας το κείμενο ψηφίζουμε για το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για την Ευρώπη των Εθνών και Ελευθεριών. Λαντσίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κλάδος της κίνησης είναι θεμελιώδης και για την οικονομία και για την κοινωνία των κρατών μελών. Ωστόσο εδώ συνεχώς ξεχνάμε αυτή τη διάσταση και δεν ακούμε τα αιτήματα των επιχειρηματιών και εργαζομένων. Τα μέτρα που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων αναχρονιστικά ή, ή ε, παράλογα. Μιλάμε για μια βιώσιμη μετακίνηση προς την κινητικότητα χωρίς κατανάλωση, χωρίς όμως να κάνει μια αξιολόγηση των αντικτύπων των μέτρων που προτείνονται. Το μέτρο μιλά, υποχρεώνει να στραφούμε στα ηλεκτρικά, εξαφανίζοντας και αγνώντας τις άλλες εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν στην αγορά. Θα έπρεπε εξ αρχής να προβλέπεται η χρήση μείγματος τεχνολογιών και μεγαλύτερες προθεσμίες για να διευκολυθούν οι επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών εκπομπών ε, μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα, ιδίως ό,τι αφορά τα ε, μεγάλα τα φωτιγά. Ο κλάδος θα πληγεί εις βάρος της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και των κρατών μελών. Η Ευρώπη θα γίνεται εξ, ακόμα περισσότερο ε, εξαρτημένη από τρίτες χώρες για την απακτήση ε, μπαταριών. Και Επιπλέον, όπως αναφέρει ο τύπος και παράδοξα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο ε, νέες στήλε για ε, ηλεκτρική ενέργεια που όμως τροφοδοτούνται από ε, δίζελ. Η, ο κλάδος της, ε, της, της οδικής κίνησης θα μπορούσε να χάσει ε, μόνο στη Γερμανία μεταξύ 75.000 και 210.000 ε, μονάδων μέσα στο 2030. Σκεφτούμε καλύτερα την πρόταση αυτή που όπως διατυπώνεται αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι ακατανόητη και με αποτελέσματα αντίθετα από αυτά που έχει ως θέση ως Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σόσνιετς. Ένα λεπτό. Ε, στα έγγραφα μιλάμε συνεχώς για μηδενικές εκπομπές, αλλά μηδενικές εκπομπές δεν υπάρχουν ούτε θα υπάρξουν. Είναι ένα εργαλείο marketing που χρησιμοποιείτε εσείς ή αυτοκινητοβιομηχανίες. Μεταφορές μηδενικών εκπομπών δεν είναι δυνατές. Κάποιο ε, ε, κάποιος θα εκπέμπει αν δεν εκπέμπουν τα οχήματα, θα εκπέμπουν οι βιομηχανίε οι οποίε θα παράγουν την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα οχήματα. Οπότε πολύ ωραία να δράσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές. Κάπου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θα χρειαστεί να μεταφερθεί. Μηδενικές εκπομπές δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν η έκθεση αυτή είναι ανεύθυνη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λίζα. μισή λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και είναι πολύ καλό το γεγονό ότι αύριο για πρώτη φορά ορίζουμε όρια για τι εκπομπέ των βραιών οχημάτων. Γιατί όλοι τα μίστα πρέπει να συμβάλλουν αυτό που του αναλογεί στη μείωση των εκπομπών. Είναι φιλόδοξο αλλά εφικτό το σχέδιο που έχουμε μπροστά μα και είναι καλό που έχουμε που δεν υποκύψαμε στις υπερβολικές ε, ε, απαιτήσει των πράσινων στο κείμενο αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπάσα για την ε, ρεαλισμό που έδωσε, γιατί ήθελε πολλά παραπάνω αρχικά, αλλά επικεντρώθηκε στα ουσιαστικά και αυτό ήθελε και το ΕΛΚ, αυτό ήθελε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν ευφυέ αυτό. Να ευχαριστώ και τον Κρίσταφερ Φιέρνερ για την δέσμευσή του, όχι μόνο για το θέμα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Αλλά θα ήθελα να πράξω την ευκαιρία όλο ιδιαίτερος για να ευχαριστήσω και τον Επιτρόπο κύριο Κανιέτα, γιατί στην ακρόαση, ακρόαση του αντιμετώπισε τα πειρά της κριτικής και τότε ακόμα και αυτοί που τον επέκριναν τότε θα πρέπει σήμερα να ομολογήσουν ότι πετύχαμε πολλά μαζί για την προστασία του κλίματος στην Ευρώπη και είναι η τελευταία νομοθεσία που θα περάσει το Κοινοβούλιο αυτό. Γι' αυτό να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Επιτροπό, τον κύριο Κανιέτε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και ένα θέμα νομίζω που θα χαρακτηρίσει την επόμενη περίοδο είναι η ενίσχυση των συντροδρόμων. Καλό είναι να ρυθμίσουμε και τα φορτηγά, αλλά θα πρέπει όλο και πιο πολλά εμπορεύματα και ε, επιβάτες να μεταφερθούν στο συντροδρόμο και να δούμε ότι σε ό,τι αφορά την ε, μείωση των εκπομπών είναι πολύ πιο επιβαρημένος ο συντροδρόμος από ότι οι άλλοι τομεί μεταφορών. Και εδώ θα πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Και κύριε Λίζε, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σόσνη, έτσι. Την αποδέχεστε βεβαίω. Με χαρά. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρο. Πολλά πατήχαμε. Πετύχαμε σε ό,τι το κλίμα σε ό,τι αφορά κάποια στερεότυπα τα οποία πέρασαν στο κλίμα. Τι θα σημαίνουν όμως όλα αυτά συγκεκριμένα για το κλίμα, ο κύριος Λίζε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά όταν ε, μου κάνετε την ερώτηση αυτή να σας το πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει τις στόχο της για το 2030 και αποφασίσαμε λοιπόν για μια νομοθεσία και αύριο θα αποφασίσουμε το τελευταίο τμήμα της νομοθεσίας αυτής, όπου νομοθετικός πώς δημιουργούμε τους όρους για να εκπληρώσουμε και με το παραπάνω τους στόχους μας για το 2040. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Ευρώπη να αποτελέσει πρότυπο και για τις άλλες επίρρους και παράλληλα έχουμε και κανόνες που δεν θα διώξουν τη βιομηχανία από την Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλή ισορροπία και όταν έχουμε τα βέλη τη κριτική και από τι δύο πλευρέ του πολιτικού φάσματο, αυτό είναι καλό δείγμα ότι είναι ισορροπημένη η νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντάλη για 1,5 λεπτό. Μυρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή μα, τον κύριο Άικχαουτ, για τη δουλειά που έκανε και το συμβιβασμό που πέτυχε, γιατί ξέρω δεν ήταν εύκολο ο φάκελο αυτό. Ήταν πάρα πολύ φοιτικό το γεγονό ότι έχουμε πλέον άλλη μία πολιτική για τη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα όπου δεν είχαμε πρότυπα για τα ε, βαρέα οχήματα. Παρά το γεγονό ότι γνωρίζαμε την μεγάλη επίπτωση που έχουν τα φορτηγά αυτά στην ε, παγκόσμια αύξηση του τη θερμοκρασία. Και αυτή αναμένεται να αυξηθεί. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να εγκρίνει δεσμευτικά πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών. Ήταν λοιπόν δύσκολο το έργο αυτό. Η διαπραγμάτευση για το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο για την θέση των benchmarks ήταν πραγματικά μεγάλο επιτεύγμα. Το ξέρω αυτό από προσωπική εμπειρία να ευχαριστήσω και τον εισηγητή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ε, τον κύριο Τσόφολη, για την μεγάλη του δέσμευση και τον ρόλο που έπαιξε για να πετύχουμε συμβιβασμό. Η θέση του Κοινοβουλίου θέτει το σωστό επίπεδο φιλοδοξίας. Αυτό χρειάζεται για να ε, καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας για το κλίμα και πιστεύω ότι το μέλλον των καθαρών οχημάτων και των φορτηγών θα καθοριστεί από την κρατομία μόνο με ισχυρά κίνητρα για την παραγωγή οχημάτων χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών τελικά θα περάσει την αλλαγή αυτή. Αυτό αποτελεί το σκόπο μας και το στόχο μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με τη δουλειά μας και προσβλέπω και τις μελλοντικές μας προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο λόγος στην συνάδελφο εγώ Νταλόντα για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Επιτέλους ε, καθορίζονται ε, στόχοι μείωσης ε, εκπομπών για τα, βόρεια, για τα βαριά οχήματα. Ε, Τέτοιου είδου στόχου και πολύ πιο φιλόδοξου είχαμε στηρίξει εμεί στην Επιτροπή Μεταφορών. Όμω η Γερμανία και άλλε χώρε πιεσμένες από την αυτοκινητοβιομηχανία τους μείωσαν τους ε, στόχους. Παρ' όλα αυτά, οι εκπομπέ διοξείδου του άνθρακα συνεχώ αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στι οδικές μεταφορέ. Αντίθετο, η αναθεώρηση του 2022 θα είναι πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου να προσαρμόσουμε την νομοθεσία και ενδεχομένω να καλύψουμε περισσότερου τύπου οχημάτων και ενδεχομένω να ξαναδούμε του στόχου μα. Παρόλο ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλης από τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα οδικό χάρτη υποχρεωτικό. Ο κανονισμό αυτός είναι ένα βήμα για να καταπολεμήσουμε την ατμοσφαιρική μόλυνση και να σεβαστούμε τους κλιματικούς στόχους, ιδιαίτερα του Παρισιού, που θα περιορίσουν την αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό προ όφελο των επόμενων γενιών. Η Ευρώπη δρά με συγκεκριμένο τρόπο κατά της μόλυνσης και τελευταία μου αυτή ομιλία στην Ολομέλεια, θέλω, θέλω να υπογραμμίσει ακριβώς αυτή την πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κάτσε διάει. Δύο αιτήματα έχουν ε, γίνει δεκτές, έχουν υποβληθεί. Φάρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Εκχάουτ και όλους τους συναδέλφους ε, που βοήθησαν να θέσουμε τέτοιους φιλόδοξους στόχους για τα βαρέα οχήματα. Επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας για διαφορετικά χαρτοφυλάκια, διαφορετικά φακέλους ε, που έχουν σχέση με τους στόχους του Παρισιού, την κυρία Ντάλη πιο συγκεκριμένα. Είχαμε κάνει πρόταση για πιο φιλόδοξους στόχους και ελπίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις, ε, οι προτάσεις του ΕΛΚ ε, βοήθησαν. Προφανώς η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας και να μειώσουμε την τοξικότητα της ανθρώπινης δράσης στον πίνακα. Οι επιστήμονες ε, στέλνουν σήμα κινδύνου στην κοινωνία αλλά ε, υπάρχει κάτι το οποίο κάνουμε, ε, δεν κάνουμε σωστά. Δεν προχωράει αρκετά γρήγορα η μείωση της χρήσης του ε, άνθρακα. Κέλλη, Σον, e έχεις το λόγο. Ασχολούμαι θέματα κλιματικά καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Και χαίρομαι για την πρόοδο που κάναμε στο Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια στον Επίτροπο Κανιέτε. Και τον κύριο Eichhout, που αποτέλεσε ατμόμηχανή μηχανή σε αυτό το τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως είπε η Μύρια Μτάλη, ε, έχουμε πλέον μια πολιτική για τα βαρέα οχήματα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές. Όσο βελτιώνεται η οικονομία, ε, εγώ πηγαίνω από το, από το, το σπίτι μου στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και από το Στρασβούργο στη Φραγκφούρτη και βλέπω όλο και περισσότερα βαρύ οχήματα στους δρόμους. Η μείωση αυτή που προβλέπουμε δεν σημαίνει ότι θα, μειώσει, θα μειωθούν οι μεταφορές. Απλά θα τις κάνει πιο α, ενεργειακά αποδοτικές. Οπότε μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Είναι μια λογική πρόοδος, προοδευτική, σταδιακή και νομίζω με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε το περιβάλλον μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Thank Ολοκληρώνει τη διαδικασία του Κατσδιάη. Το λόγο τώρα για την Επιτροπή ο Επίτροπος Άρια Κανιέται. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές, για τη συζήτηση αυτή. Να απαντήσω σε μια απευθεία ερώτηση που μου έφεσε ο κ. Σόσνιεκ. Ρώτησε, τι έκανε αυτό το κοινοβούλιο για την αργή του κλίματος. Η απάντηση μου είναι πολλά. Τι έκανε, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αργή του κλίματος. Όχι πολλά. Πριν το 2020 θέσαμε στόχους μείωσης των εκπομπών και το 2017 μειώσαμε τις εκπομπές κατά 17% σε σχέση με το 1990. Μειώσαμε τις εκπομπές, αναπτύξαμε, αναπτύξαμε τα ανανεώσιμα, κάναμε καλύτερη ε, λειτουργία των επιδόσεων, αλλά το κοινοβούλιο αυτό διπλασίασε το πλαίσιο για την ενέργεια. Ήμουν στην πολιτική, είμαι στην πολιτική 38 χρόνια. Έχω έχω, έχω υπηρετήσει σε εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Ποτέ δεν είδα τόσο έντονη νομοθετική διαδικασία ε, δραστηριότητα όσο εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους των επιτροπών, την κυρία Βάλη, τον κύριο Μπούσεκ, τον, τον Τζοβάνι Λαβία, όλους τους εισηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Άικχαουτ, που έκανε εξαιρετική δουλειά που ήταν και δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις όπως στα ανανεώσιμα. Και αυτό που κάναμε είναι ότι υιοθετήσαμε πολλά νομοθετικά κείμενα που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών το 2011 κατά 45% και αν αλλάξουν και θα αλλάξουν το 2030 θα έχουν 60% μειώσεις των εκπομπών, με μεγάλο πακέτο. Και ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο μέσος, το μέσο ποσοστό πολιτικών, πολιτικής υποστήριξης προτάσεις αυτές. Στο πακέτο ενέργειας 80% των ψηφοφοριών ήταν υπέρ. Στο κλίμα 76%. Σημαντική λοιπόν πολιτική υποστήριξη για την νομοθεσία που υιοθετήσαμε το 2030 που σημαίνει ότι είχαμε έναν διάλογο, υπήρχε αμοιβαία κατανόηση, υπήρχαν διαπραγματεύσεις και όπως σας είπα ήταν μια απίθανη ευκαιρία. Μετήσχα σε 71 τριμερείς διαλόγους. Δύσκολους που πάνω από 350 ώρες της ζωής μου. Αλλά ήταν εξαιρετικές ευκαιρίες για να μάθω και να σας ευχαριστήσω όλους γιατί η δουλειά αυτή ήταν μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την δική σας εμπλοκή. Εσείς πιέζετε και εμείς ε, απαντάμε. Αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος του καθενός. Το βασικό στοιχείο είναι ότι περνάμε ένα κείμενο που θα εφαρμοστεί για την επόμενη 20 ετία, αλλά έχουμε τη δυνατότητα αναθεώρησης καθοδών για, με αύξηση των στόχων. Στις 77% των πιθανών ψηφοφόρων για τις ευρωεκλογέ ανέφεραν σε μία σφιγμομέτρηση την περασμένη εβδομάδα ότι το περιβάλλον ήταν ο βασικός λόγος να πάνε να ψηφίσουν τις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένας βασικός παράγοντας για να συζητηθεί στις Ευρωεκλογές. Σα παροτρύνω να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, να εξηγήσετε στους πολίτες της Ευρώπης τι κάναμε αυτά τα πέντε χρόνια. Και επίσης, να πείτε τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο στις κάλπες και θα μπορέσει το Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία να βοηθήσει την ολοκλήρωση του πακέτου, την περαιτέρω πρόοδο και την συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να μπορέσει η Ένωση να γίνει το 2020 η πρώτη μεγάλη οικονομία που θα είναι ε, ε ενεργειακά ουδέτερη. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα ο κ. Σάικα, ο εισηγητής. Μπάς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και καταρχά, μια και βρισκόμαστε σε τέτοια κλίμα ευγνωμοσύνη, να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο, τον Επίτροπο Μαρία Κανιέτα, για τη δουλειά που έκανε. Και προφανώ και είχαμε στιγμέ ε, όπου διαφωνήσαμε και κάποιε από τι ώρε αυτέ τι ε, περάσαμε μαζί. Να πω ότι Ανά πάσα στιγμή ο διάλογο ήταν καλό. Δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά υπήρχε πάντα αμοιβαίο σεβασμό και αυτό είναι απαραίτητο για το μέλλον. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πετύχαμε πολλά. Πετύχαμε πολλά για το κλίμα, για την ενέργεια, για την κινητικότητα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει όμω το έργο μα. Και αυτό, όπω είπατε, δεν έχουμε ακόμα ε, μπει στη σωστή τροχιά για την ε, ε, οικονομία τυφλική προς το κλίμα. Και αυτό θα το τονίσουμε και αύριο. Και είναι ένας από τους λόγους αυτούς για του οποίου αύριο και στις ευρωεκλογέ. Το θέμα θα είναι το κλίμα, θα είναι οι εκλογές του κλίματος. Και να σας πω, δυστυχώς να δώσω και ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναήλθατε, γιατί μπορώ να σας απαντήσω για το που εμείς ως Κοινοβούλιο κάναμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο φιλόδοξη. Καταρχάς, ο, ο στόχος για το 2030 πλέον είναι νομικά δεσμευτικός. Αυτό δεν ήταν στην αρχική πρόταση. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαφές μήνυμα για το που οδεύουμε. Δεύτερον, κλείσαμε πολλά παραθυράκια στις προτάσεις και κυρίως αυτά για τις ε, για τα υπερπιστωτικά μόρια σε ό,τι αφορά τα ε, οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και τρίτων ε, σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα για τα οχήματα στον δρόμο, τα βελτιώσαμε για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι αυτά που συμφωνούμε θεωρητικά θα εφαρμοστούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τον Dieselgate. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τόσο απαραίτητα και τόσο κρίσιμα πέρα από τι τεχνικέ βελτιώσει και τι ρήτρε αναθεώρηση και το καθεξή. Και αυτά τα τρία στοιχεία είναι τόσο σημαντικά λοιπόν που στέλνουν ένα μήνυμα προ του επενδυτέ, του κατασκευαστέ ότι το μέλλον θα είναι μηδενικέ χαμηλέ εκπομπέ στα οχήματα και ότι αν συνεχίσουν όπως ε, σήμερα δεν θα πάνε μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαστικά λοιπόν καταλαβαίνω σας έδωσα τις απαντήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία να δούμε τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και μετά εν ώψη και τη Συνόδου στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, γιατί περιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τις ε, εθνικές της ε, συνδρομές βλέπω να προσεύχεται και ο Επίτροπος να ευχηθώ και εγώ για αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Πέρα τη συνδρίαση. Και θα γίνει αύριο η ψηφοφορία. Βάσει τη ημερήσια διάταξη, προχωρούμε τώρα στην ε, έκθεση Γκαζίμπ για την πρόθεση καθαρών και ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Δίνω αμέσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Γκαζίμπ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε, κυρία Επίτροπε. Πρόκειται για μια οδηγία που θα στηρίξει τα οχήματα, ε, τα ενεργειακώς πιο αποδοτικά οχήματα. Το 60% ορισμένοι λένε 65-66% της μόλυνσης ε, στις πόλεις λέγεται ότι οφείλεται στον τομέα των μεταφορών. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα οχήματά μας, ε, τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, αλλά υπάρχουν εκπομπές και από αλλού. Και αυτό το βλέπουμε στους, στις κρατικές προμήθειες και στους δημόσιους διαγωνισμούς. Αν εγκρίνουμε αυτό το κείμενο θα εγκρίνουμε πολύ φιλόδοξου στόχους και πρέπει αυτοί οι στόχοι να είναι εφαρμόσιμοι στην πράξη. από τις δημόσιες διοικήσεις. Οπότε είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να στηριχθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη και τις δυνατότητες των διαφορετικών κρατών μελών. Ελπίζουμε να μπορούν να υλοποιηθούν και τα κράτη-μέλη να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο. Προφανώς δεν μιλάμε για το 100% των αγορών γιατί υπάρχουν παραδοσιακές τεχνολογίες, σημαντικές τεχνολογίες που δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Οι τοπικές αρχές μας είπαν, ε, για παράδειγμα, ότι τα υβριδικά οχήματα είναι μια καλή βοήθεια για να μειωθούν οι εκπομπές και να προχωρήσουμε προς μηδενικές εκπομπές. Υπάρχει μια τεχνογνωσία που ήδη είναι γνωστή για αυτά τα οχήματα. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσουμε μια ελαστικότητα μέσω της ε, οδηγίας για τα εναλλακτικά καύσιμα. Για παράδειγμα, πρόκειται για κείμενα τα οποία ήδη υπάρχουν. Το κείμενο αυτό αφορά και τα βαρέ και τα ελαφρά οχήματα και θα επηρεάσει και τα λεωφορεία στις δημόσιες μεταφορές. Οι περισσότερες αγορές γίνονται μέσω κρατικών διαγωνισμών, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Η, τα αυτοκίνητα είναι ο βασικός στόχος αυτής της οδηγίας, μπορώ να πω και οι κατασκευαστές των λεωφορείων έχουν πλέον τεχνολογία την οποία θα πρέπει να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο και να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου τα νέα λεωφορεία να μπορούν να ανταγωνιστούν στις παγκόσμιες αγορές, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, η, ε, εταιρεία Solaris στην Πολωνία έχει λεωφορεία με μηδενικές εκπομπές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι η τεχνολογία ε, χαμηλών εκπομπών η οποία αναπτύσσεται με τη χρήση βιομεθανίου για παράδειγμα θα επιτρέψει να μειωθούν οι εκπομπές ε, στις ε, δημόσιες μεταφορές. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επωφεληθούμε καλύτερα από το βιοαέριο, τα βιοκάψιμα Κάτι το οποίο θα είναι πολύ θετικό για το περιβάλλον μας. Το βλέπετε αυτό στην πρότασή μου. Στο μέλλον θα κατασκευάζονται οχήματα μηδενικών εκπομπών. Αυτό το ξέρουμε. Και οι τεχνολογίες βελτιώνονται. Όμως θα πρέπει να δούμε τις τεχνολογίες αυτές στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, μπαταρίες και συσσωρευτές. Και αυτοί επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον, το βλάπτουν. Οπότε θα πρέπει να γίνει η, μείωση να γίνει ε, οριζοντίως. Ε, πρέπει να μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και από τις μπαταρίες να μπορούν να ανακυκλωθούν κλπ. Επίσης, να μπορούν να χρησιμοποιούν οι μπαταρίες λιγότερους ε, μολυσματικούς παράγοντες. Θα πρέπει να δώσουμε αυτόν τον τρόπο μια όθηση στις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες για βελτιωμένες απόδοσης μπαταρίες και πιο καθαρές μπαταρίες. Η αυτοκινητοβιομηχανία με την κατάλληλη έρευνα και καινοτομία θα παράγει αυτοκίνητα, οχήματα τα οποία πραγματικά θα είναι πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο χρήσιμα. Ε, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες τους συνεισηγητές και οδησηγητές Είχαμε μερικά προβληματάκια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν που στις δύσκολες στιγμές μας βοήθησε να βρούμε συμβιβασμούς. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρουμανική Προεδρία που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή, η Επίτροπος. Πούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλωσορίζουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με τη, μαζί σας την έκθεση Γκοζίμπ. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Και εσείς και οι συνηγικαίοι και οι όχι μόνο τώρα, αλλά σε όλη τη διαδικασία. Όπως είπατε, η συνεργασία δεν ήταν πάντα εύκολα, ήταν ανοιχτή, με αφοσίωση και με αποτελέσματα. Χάρη στην δέσμευση και την αποφασιστικότητα όλων των τριών εμπλεκόμενων στην νομοθεσία οργάνων είχαμε σωστό, καλό αποτέλεσμα. Ένα καθαρό πακέτο κινητικότητας. Ο, ο δημόσιος τομέας έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της απομάκρυνσης από τον άνθρακα στις μεταφορές. Η λεωφορία, τα λεωφορεία κυρίως όπου οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 70% της αγοράς χρησιμοποιώντας ε, την, ε, τις δημόσιες συμβάσεις για την επιτάχυνση των καθαρών οχημάτων, η οδηγία επιτρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για, την για τη συγκινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Κατά την άποψή μα, το κείμενο που συζητήθηκε στον τριμερή διάλογο στις 11 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεύει μια καλή συμβαστική λύση μεταξύ των διαφόρων θέσεων και ε, ετοιμάτων. Δείχνει ότι υπάρχει επαρκή φιλοδοξία, αφήνοντα ε, αρκετή ευελιξία για την υλοποίηση, ούτως ώστε οι στόχοι της οδηγίας να μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς μεγάλο διοικητικό βάρος για τις δημόσιες αρχές. Με την, με την έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας δίνουμε ορισμό ότι είναι καθαρό όχημα και θέτουμε σαφείς στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίω ειδικού στόχους για λεωφορεία μηδενικών εκπομπών. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι η συμφωνία που επιτεύχθη στον τριμερή διάλογο θέτει επαρκή, επαρκώς σαφή ορισμό και επαρκώς φιλόδοξους εθνικούς στόχους. Το κείμενο επίσης δίνει μεγάλη ευελιξία για το πώς οι προσπάθειες ε, επιμερίζονται μεταξύ κρατών μελών, επιτρέποντας μία κοστοποτελεσματική εφαρμογή που δεν θα δημιουργήσει σημαντική επιβάρυνση στις αρχές των κρατών μελών πολλές πόλεις μας, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, ε, η Βαρσοβία, το η Βαρκελόνη, το Μιλάνο, η Λουμπλιάνα, το Μόναχο και πολλές άλλες ήδη έχουν αναλάβει εθελούσιες δεσμεύσεις ξεπερνώντας αυτό που απαιτεί η οδηγία. Θα βοηθήσουμε και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το παραδείγμα τους. Η αναθεώρηση θα επεκτείνει και το πεδίο εφαρμογής οδηγίες για να καλύπτονται δημόσιες ε, προμήθειες μέσω πρακτικών όπως ε, ε, ενοικίαση πώληση και σύντομη ενοικίαση. Αυτό θα αντικατοπτρίζει και τις καλύτερες πρακτικές των κρατικών προμηθειών, μειώνοντας τον αντίκτυπο στην αγορά. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα παράσχουν σαφή μηνύματα προς την αγορά επιτρέποντας τις αρχές, τους κατασκευαστές και τους επενδυτές να προγραμματίσουν καλύτερα την μετάβασή μας μέχρι τα μέσα του αιώνα στην κινητικότητα μηδενικής ε, εκπομπής, βελτιώνοντας την μείωση της συμμετοχής του άνθρακα στην κινητικότητά μας και την επίτευξη του μηδενικού στόχου το 2050. E Ευχαριστώ Επίτροπε. Για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Δέλη Έχει το λόγο που δεν είναι εδώ όμως. Αργότερα. Πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε από το ΕΛΚ. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των επιζήμιων ουσιών αριθμίζεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, αποδοτικότητα, την ενεργεία και τη μείωση των εκπομπών. Και έτσι λοιπόν εργαζόμαστε καλύτερα στον οικολογικό σχεδιασμό, στη ενεργειακή επισήμανση και σε πολλά άλλα θέματα συνεργαζόμαστε ευρωπαϊκά. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει τέτοια εγγύηση Είμαστε υπέρ των ευρωπαϊκών διατάξεων. Δεν θα πρέπει όμως να επισέλθουμε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομερίας και κυρίως όχι στους δήμους και στις κοινότητες να μπούμε να κάνουμε κομμάτι με τις διατάξεις αυτές ε, κυρίες και κύριε θεωρώ ότι ε, ανοίγουμε ένα μεγάλο πλήγμα στον κόλπο των ε, δήμων και κοινωνιτήτων γιατί απέχουμε πολύ από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις για τα ηλεκτρικά ε, λεωφορεία. Κάνουν τις μεταφορές πολύ ακριβές και το πώς ε, ρυθμίζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να τα αφήνουμε στο ε, επίπεδο των τοπικό. Όχι να υπάρχουν ε, γενικές διατάξεις από τις Βρεξέλλες και στην πατρίδα μου θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση και δικαίως για την υπερβολική ανάμειξη των Βρυξελών και μεγάλο τμήμα του ΕΛΚ θα απορρίψει την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Και το λόγο λοιπόν τώρα έχει από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ο κύριος Ντάνς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Της ευχαριστίας μου στον εισηγητή, τον κύριο Γκριπ και την Κομισιόν. Το Συμβούλιο Κρίμα δεν είναι εδώ. Εξαιρετική δουλειά που έχουμε κάνει. Κύριε Κρύπ, είσαστε πολύ δίκαιος ως συγητής, πολύ αμερόληπτος. Ε, διεξάγατε τι διαπραγματεύσει μεταξύ των διαφορετικών ομάδων με εξαιρετικό τρόπο. Συγχαρητήρια. Ο φάκελο αυτός είναι πολύ καλό παράδειγμα για το λόγο για τον οποίο έχουμε εκλεγεί εδώ και το ρόλο μας. Πρέπει να γίνουμε πιο δραστήριοι στον καθαρισμό των οχημάτων, στο να κάνουμε τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους πιο καθαρά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, α, αλλά και γιατί ε, η ποιότητα γενικότερα του αέρα της πόλης είναι πολύ κακή. Οι κρατικές προμήθειες αντιπροσωπεύουν το 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 45% των ε, λεωφορείων που κυκλοφορούν. Είναι λοιπόν πολύ σωστό και πολύ επίκαιρο που θα χρηματοδοτήσουμε τα πιο φτηνά, ε, πιο συγγνώμη, καθαρά οχήματα ε, μέσω των κρατών μελών. Το 2030 το 60% των λεωφορείων θα πρέπει να πληρούν τους όρους οδηγίας. Η Κομισιόν βέβαια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές αρχές θα έχουν τα κατάλληλα μέσα και επαρκείς πόρους. Απαντώντας στους συναδέλφους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω το εξής. Χρειαζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μας και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα από μόνα τους κάπως θα κινηθούν. Πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις σήμερα. Σε όλα τα κράτη-μέλη βλέπουμε νέου να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται και όχι μόνο νέου, γενικότερα ευαισθητοποιημένου πολίτε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Και είμαι περήφανο που το κάνουμε. Το Κοινοβούλιο και οι πόλεις είναι αυτέ που ζητούν πάντοτε περισσότερα, ενώ τα, οι κυβερνήσει, οι κεντρικέ κυβερνήσει είναι αυτέ που κρατάνε τα χαλινάρια. Αυτή είναι η εμπειρία μου τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στο κοινοβούλιο αυτό ω Βρετανό. Αν όμω αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε εδώ για να κάνετε το ορθό. Έμαθα πολλά από εσά και ελπίζω θα επιστρέψω για να μάθω περισσότερα. Thank you very much, dear colleague, and good luck. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Καλή τύχη σας εύχομαι. Και τώρα το λόγο έχει από το ECR ο κύριος Ντεμέσμακερ για 1,5 λεπτό. Μάρκα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπή, συνάδελφοι. Πριν από λίγο συζητήσαμε για τις πρώτες μειώσεις των διοξιδίτων ανθρακά για τα βαρέα οχήματα. Και τώρα έχουμε ένα φάκελο για τα καθαρά και ενεργειακώς αποβατικά οχήματα και πώς θα μπορούμε να τα προωθήσουμε. Είναι καλό το αποτέλεσμα και νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ως μήνυμα για την τελευταία ε, ολομέλεια αύριο, την ψηφοφορία δηλαδή, τη τρέχουσα θητεία, θα έχουμε δύο φορέ την ευκαιρία να επιλέξουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Στην ε, καταπολέμηση τη ρήπανση τη ατμόσφαιρα, οι δημόσιε συμβάσει αποτελούν όντω ένα σημαντικό κίνητρο για την μετάβαση σε μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών οι αρχές θα πρέπει να δράσουν ε, υποδειγματικά. Και η δική μου κυβέρνηση, η φλαμανδική ε, κυβέρνηση, είναι υπέρ μια τέτοιας βιώσιμης πολιτικής. Χρειάζεται λοιπόν η μετάβαση αυτή για την ε, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στις πόλεις μας και στις κοινότητε μας και κυρίως στη χώρα μου. Για την, το κόμμα μου, για το NVA, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν στην συμφωνία τεχνολογικά ουδέτερες λύσεις, όχι μόνο α, οχήματα με μπαταρίες και ηλεκτρικά, αλλά υβριδικά με ε, υγροποιημένο αέριο κτλ. Χρειαζόμαστε όλες τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να κινηθούμε πραγματικά προς μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα από την Άλτε το λόγο έχει ο, η κυρία Μιλμπάου Μαραντίκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Αυτή η πρόταση πρέπει να δώσει δύο βασικά χαρακτηριστικά στον κοινό μας στόχο της μείωσης των εκπομπών στις μεταφορές κατά 20% μέχρι το 2025. Ε, δύο βασικά χαρακτηριστικά, ρεαλισμό και σαφήνεια. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για να... Ε, σχετικοποιήσουμε τα όσα λέγονται για τον δίζελ. Γιατί μας, ε, το δίζελ μας εμποδίζει να μειώσουμε ε, το, τις εκπομπές, περιμένοντας τις μηδενικές εκπομπές και ε, δημιουργεί μεγάλο κοινωνικό κόστος, διότι ήδη βλέπουμε μείωση στις, στην απασχόληση εξαιτία της κρίσης του δίζελ. Και υπάρχουν εναλλακτικέ που είναι πολύ πιο καθαρές από τον δίζελ. θα πρέπει η μετάβαση να γίνει σταδιακά προς τις μηδενικές εκπομπές. Ε, θα πρέπει να μπορούμε με ρεαλισμό να καθορίσουμε σαφείς στόχους για το μέλλον. Άλλες ε, χώρες, στους οποίες πουλούν οι δικοί μας κατασκευαστές, το έχουν ήδη κάνει. Προβλεψιμότητα και ρεαλισμός ε, θα πρέπει να βοηθήσουν και τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να ε, διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους με τρόπο έτσι ώστε να αποδώσουν στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο αυτό το κείμενο πέραν το ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κρίσης της πωλήση, θα βοηθήσει, θα ενθαρρύνει μια βιομηχανική πολιτική προς τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Επίσης, ε, θα επιτρέψει σε κάθε τύπο μεταφοράς να προσφέρει ό,τι μπορεί σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, την κοινωνική αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η εμφάνιση νέων τύπων πρόσβαση στα οχήματα. Για παράδειγμα, σε ορισμένε ε, χώρε, όπω τη δικιά μου, ο μέσο όρο ηλικία των αυτοκινήτων από 8 έτη το 2007 πέρασε στα 12,4 το 2017. Το 62% μάλιστα έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών. Και θα φτάσει και μερικέ φορέ στα βαν, στα μικρά επαγγελματικά οχήματα φτάνει τα 13 έτη. Το να μπλοκάρουμε την ανανέωση του στόλου περιμένοντα τα οχήματα μηδενικών εκπομπών είναι πολύ κακό, θα ήταν πολύ κακή είδηση και για το περιβάλλον και για την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά ο κύριος, η κυρία Κονέτσινα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ποιο είναι πραγματικά το αποτέλεσμα αυτό. Υπερβολικές απαιτήσει στους παραγωγούς για τη μείωση των εκπομπών και τίποτα άλλο. Το κείμενο της οδηγίας για την πρόθεση των ε, αποδοτικών οχημάτων ε, θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια αγορά ελεύθερων, ε, καθαρών οχημάτων, αλλά έχει φτάσει πάρα πολύ αργά και περιλαμβάνει πολλά παραθυράκια. Οι, οι αυτοκινητοβιομηχανίε θα πρέπει να δαπανίσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες, αλλά ποιος θα τις αγοράσει. Ο κρατικός τομέας ε, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Τα κράτη-μέλη μεταθέτουν το φορτίο και το κόστος στους κατασκευαστές. Στην πραγματικότητα δεν θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών. Τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς επίσης δεν ήταν ικανοποιητικά. Η, η περίοδος μεταγραφής είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ικανοποιητική. Το Κοινοβούλιο πούλησε το θέμα αυτό πολύ φτηνά. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, είναι η τελευταία φορά, θα σας πω, που προεδρεύω στην Ολομέλη αυτή, τη θητεία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την δυνατότητα που μου δώσατε εσείς οι πολλοί και οι λίγοι εδώ σήμερα να είμαι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της ιδέας μου προσπάθησα να τιμήσω την θέση αυτή με συμμετοχή, δέσμευση και βούληση να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει όταν ε, προσπάθησα να επαναφέρω τον πλουραλισμό μέσα στο Προεδρείο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας κβάθους καρδίας και ε, καλή επιτυχία σε όλους όσοι κατεβαίνουν στις εκλογές για να βελτιώσουν την Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Για τους ε, πράσινους, ο κύριος Μαρτσελέζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως έλεγε χθε η Γκρέτα Τόμπεργκ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σπίτι, το σπίτι μας ε, ε, καταραίει. Αυτό έχουμε μπροστά μας μια κλιματική κρίση και χρειάζεται σήμερα, χτες μια λύση. Ο, ο, κλάδος των οδικών μεταφορών είναι από τους πιο ρηπογόνους. συμφωνούμε σήμερα να βελτιώσουμε την κατάσταση ζητώντας από όλα τα κράτη-μέλη ε, να αντιμετωπίσουν πείσουν το 20% των οχημάτων με, με καθαρότερο τρόπο. Αυτό σίγουρα είναι βελτίωση. Ωστόσο, όπως θύμισε χτες η Γκρέτα Τόμπεργκ, μπροστά στην κρίση δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά ό,τι είναι δυνατό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πραγματική επανάσταση στον κλάδο των μεταφορών και της κινητικότητας, μια, μια, μετα, μια επανάσταση στην υγεία και το κλίμα. Για παράδειγμα, στις πόλεις της Ισπανίας, ε, Βαλένθια, Μαδρίτη, γίνεται μία μετάβαση σε μία βιώσιμη μετακίνηση χωρίς καύσιμα, χωρίς ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας, ε, ένας στόλ, θα έχουμε ένα στόλο ε, λεωφορείων καθαρά 100% ε, χωρίς, χωρίς ε, ορυκτά καύσιμα του χρόνου. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβολικανιά. Ένα λεπτό από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μεταφορές στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουν πιο καθαρές και θα χρειαζόμαστε πιο φιλικές προς το περιβάλλον όδους μεταφοράς. Και νομίζω ότι είναι σωστό το γεγονός ότι με την οδηγία αυτή θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι οι δημόσιες προμήθειες θα δώσουν το καλό παράδειγμα. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, γιατί οι δημόσιες μεταφορές αποτελούν 75% των, ε, οι δημόσιες μάλλον αγορές ε, το από πλευρά των κρατών αποτελούν των ε, συνολικών και έτσι Στη Γερμανία έχουμε πολλά καλά παραδείγματα. Ε, το Βερολίνο μέχρι το 2030 θέλει να είναι χωρίς εκπομπές ε, μέχρι το 2030 και ήδη στην πατρίδα μου έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία, πιο πολύ από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Γερμανία. Όλα αυτά είναι εφικτά λοιπόν και γι' αυτό είναι σημαντικό και τα λεωφορεία με βιοαέριο να αναγνωριστούν για ε, τα λεωφορεία αστικά λεωφορεία που καλύπτουν μεγαλύτερε αποστάσει. Και νομίζω λοιπόν ότι κάνουμε ένα πολύ καλό και σημαντικό βήμα με την τρέχουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Σάλντεμούζα είναι η επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε πολλά κλιματικά προβλήματα και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Όλοι όσοι παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Και χθες αυτό μας είπε και η Γκρέτα Τούνμπερκ. Έχουμε λοιπόν ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά και τις πολιτικές και σε ό,τι αφορά την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας που είναι πολύ φτωχή ποιότητα. Ε, τα καθαρά οχήματα είναι τμήμα τη λύση, θεωρώ, και πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε θέσει του στόχου σε πιο υψηλό επίπεδο, να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, κάτι κάνουμε τουλάχιστον τώρα θέτουμε δεσμευτικού στόχου για του Δήμου και τι κοινότητε σε ό,τι αφορά την πολιτική των δημοσίων συμβάσεων, τι αγορέ, τι δημόσιε των οχημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν επιλύει το πρόβλημα τη ρήπανση τη ατμόσφαιρα, δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω, ελπίζω το επόμενο κοινοβούλιο να δείξει πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξία από ότι και εμεί. Καλωσορίζουμε παρόλα αυτά το γεγονό ότι γίνεται μία βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπούλτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι που παρατηρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει ε, αυτή την πρόταση. Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον εισηγητή και τους και εισηγητές για τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις που μας επέτρεψαν να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή έγκαιρα πριν διακόψει το Κοινοβούλιο μαζί με, άλλα, μαζί με τα άλλα στοιχεία των πακετων κινητικότητας κινητικότητα 1-2-3, η αναθεωρημένη οδηγία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να μα βοηθήσει να πετύχουμε σημαντικέ μειώσει εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, που είναι απαραίτητες προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας με τη Συμφωνία COP29 του Παρισιού. Η υιοθέτησή της θα αποτελέσει έγκυρη, έγκαιρη συγγνώμη, συνεισφορά στην επίτευξη αυτών των στόχων μέχρι το 2025. Πριν κλείσω, θα ήθελα όμως να κάνω ένα-δύο σχόλια στα όσα είπατε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας μας. Πράγματι, αυτό το πακέτο, αυτή η πρόταση, είναι φιλόδοξη. Αλλά αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ακριβώς αυτό. Ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστική και συνάδει με τις προβλέψεις για την αγορά. Να υπογραμμίσουμε ότι η πώληση γύρω τη σημαντικά δίκτυα δηλαδή πόλεων, ε, τοπικές, ε, η Local Governance for Sustainability, το Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων έχουν ε, εκφράσει και στο Κοινοβουλίο και στην Ρωμανική Προεδρία την πλήρη στήριξή του στην πρόταση της Κομισιόν. Οπότε ναι, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές είναι έτοιμες. Τα οχήματα με μηδενικές εκπομπέ αυτή τη στιγμή στηρίζονται σε... Ε, ε, είναι, έχουν ψηλή τιμή, αλλά αν το κόστος αυτό διαιρεθεί με το χρόνο ζωής τους, μειώνεται και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο μέχρι ε, να εφαρμοστεί η Οδηγεί αυτή, πολύ δε περισσότερο, που οι οικονομίες κλίμακος θα ρίξουν ακόμα περισσότερο το κόστος. Η οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε και υπάρχοντα ε, ε χρηματοδοτικά όργανα όπως το Connecting Europe, Facility, ε, το EFSI κλπ. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα κονδύλιο ακόμα και για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από πολλές ε, ευρωπαϊκές πόλεις. Οπότε είναι σημαντική η σαφής στόχη για τις κρατικές προμήθειες και θα διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Ένα σχόλιο τώρα σε ό,τι αφορά μάλλον κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τον Ιούνιο 2018 μια ομάδα μεγάλων αυτοκινητοβιο... αυτοκινητοβιομηχανιών, Solaris, Skoda, ε, Volkswagen, Ursus κλπ. έστειλαν μια ανοιχτή επιστολή στο Συμβούλιο και ζητούσαν περισσότερα φιλόδοξους στόχους από αυτούς που πρότεινε η Κομισιόν και επιβεβαίωναν ότι είναι έτοιμες να ανταποκριθούν. Οπότε ενθαρρυνόμαστε σε αυτή μας την, ε, σε αυτήν την κατεύθυνση που κινούμαστε και από τις δύο πλευρές. Και από τους αγοραστές και από τους πολιτές. Επίσης να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε. Πολλές μεγάλες πόλεις ήδη έχουν ξεπεράσει τους στόχους σε ό,τι αφορά στις, ε, ε, στις ε, δεσμεύσεις τους. Ο στόχος της οδηγίας είναι να ενθαρρύνει και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν αυτό το καλό παράδειγμα, αναγνωρίζοντας ότι Πολλέ μικρέ και μεσαίε πόλεις ενδεχομένω δεν είναι ακόμα έτοιμε, δεν έχουν επαρκή τεχνογνωσία ή πόρου όπω το Άμστερνταμ ή το Παρίσι. Είμαστε όμω έτοιμοι να τι βοηθήσουμε για να διαπραγματευτούν από κοινού καλύτερε τιμέ με την αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε αναμένω να υιοθετηθεί η έκθεση ε, του κύριου Ξύπ αύριο. Αυτό το θέμα, αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουμε τη σαφή ανάγκη και ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Yes, Madam Ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σας λόγια. Οπότε τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Τσίπα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ηλεκτρισμός ως πηγή ενέργειας είναι πράγματι πολύ αποτελεσματική πηγή για τα αυτοκίνητα. Είναι βέβαια ακριβώς, ακριβή πηγή. Επίσης γνωρίζουμε ότι στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα αυτού, δηλαδή των καθαρών οχημάτων, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και στην ε, παραγωγή, στην κατασκευή ε, οχημάτων. Πώς θα πείσουμε λοιπόν τον κόσμο εφόσον θα έχουμε πιο καθαρό αέρα, ατμόσφαιρα. Τα καθαρά οχήματα βοηθούν να έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, άρα αυτό ακριβώς που θέλει ο κόσμος και ζητά. Και έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει ένας καθηγητής σε μια πολωνική πόλη που του αρέσει να τρέχει. Και μετά από πολλά χρόνια που έτρεχε είπε «Ξέρω ότι έχω κάνει κάτι στραβό, κάτι λάθος, γιατί τώρα έχω πρόβλημα με τα πνευμόνια μου». Αυτό δείχνει πόσο πολλοί είναι οι πολίτες που τελικά έχουν προβλήματα στην αναπνοή, πεθαίνουν πρόωρα εξαιτίας της ρήπανσης της ατμόσφαιρας. Όλο περισσότερες πόλεις βλέπουν τις αρχές τους να αποφασίζουν να περιορίζουν την πρόσβαση των οχημάτων στο κέντρο των πόλεων αυτών. Και τα μόνα οχήματα τα οποία επιτρέπονται είναι τα ηλεκτρικά. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε κάποιος νωρίτερα εδώ, ότι Σίγουρα επιβάλλονται περιορισμοί από τις χώρες μέλη, από τις τοπικές αρχές, σε μερικές περιπτώσεις, αλλά ε, δεδομένων των επαφών που έχω με την τοπική αυτοδιοίκηση σε περιφέρειες, πόλεις, δήμους κτλ. Πρώτα γίνονται διαβουλεύσεις και μετά λαμβάνονται αποφάσεις. Και βλέπω ότι ο κόσμος τελικά ε, θέλει να δεχτεί τον ευρύτερο ορισμό για οχήματα μηδενικών εκπομπών, καθαρά οχήματα που κυκλοφορούν με μεθάνιο, με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να προσαρμόσουμε επίσης τα οχήματα που ήδη βρίσκονται στην αγορά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε αναπτύξει στις διαβουλεύσεις που έχουμε τους κοινωνικούς εταίρους και με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, κυρίως τις τοπικές αρχές, γιατί μας λένε τι περιμένουν να περιλαμβάνει η νομοθεσία αυτή προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Εννοείται ότι πρόκειται για ένα συμβιβασμό μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων του Κοινοβουλίου, ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θέλω να εκφράσω εδώ τις ευχαριστίες μου σε όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτού του κειμένου. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετά το 2020 θα στηρίξουν τους στόχους της οδηγίας. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο για εκείνους που θέλουν να εμπλακούν στην υλοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συνεργασία σας, όλους σας, για τη συνεργασία σας όχι μόνο στην οδηγία αυτή ε, και σας, γιατί όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε κάτι. Δεν συμφωνούμε πάντα όλοι σε όλα, αλλά πιστεύουμε όλοι ότι κάνουμε κάτι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα λάβει χώρα αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπούλς για την παρουσία της εδώ. Καλό σας βράδυ. Και καλωσορίζω εδώ την κυρία Γιούροβα, την Επίτροπο Γιούροβα και θα συζητήσουμε τώρα μαζί της την έκθεση του κυρίου Ταντέου Σβιεύκα. Πρόκειται για την χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Η έκθεση του κ. Ζιέφκα. Έχετε το λόγο κ. Ζιέφκα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσά, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, βλέπουμε ότι η θητεία ολοκληρώνεται, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία και πρέπει να εγκρίνουμε. Η ευρωπαϊκή αγορά, οι επιχειρήσει στην Ευρώπη περιμένουν και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή ε, να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα, ε, Επίσης, να ευχαριστήσω την ομάδα της γιατί ε, έκαναν ε, πάρα πολύ καλή δουλειά, ε, κατέθεσαν μια θαυμάσια πρόταση και έτσι περιόρισαν και το χρονικό διάστημα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τέστη λοιπόν δυνατόν να διεξάγουμε τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο με απόλυτη ηρεμία και ησυχία. Ευχαριστώ τους και τις εισηγήτριες, τους συναδέλφους μάλλον, που ήταν σκιώδη εισηγητές. Περί πρόκειται, πρόκειται για το εταιρικό δίκαιο που είναι πολύ σημαντικό για την κοινή αγορά. Και πρόκειται κατ' ουσίαν και για ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία, την ψηφιοποίηση. Η νέα οδηγία δίνει νέες δυνατότητες για την καταχώρηση των επιχειρήσεων, όπου ε, μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τις ε, ψηφιακές ε, τεχνολογίες, συγκεκριμένα το διαδίκτυο. Είναι βέβαια λίγο περίεργο το ότι μόνο στο τέλος της θητείας συζητάμε για την ψηφιοποίηση σε σχέση με τα δικά μας τα θέματα για την κοινωνία της πληροφορίας. Μιλάμε αρκετό καιρό, αλλά τώρα αυτό που ενδιαφέρει είναι το τι προσδοκούν οι εταιρείε από εμάς. Κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ο στόχος που έχουμε είναι η βελτίωση, η διευκόλυνση της ζωής των εταιριών σε αυτό το θέμα της καταχώρησής τους. Πρόκειται για έγγραφα, παραστατικά, το πώς ε, διαβιβάζονται, ε, το πώς γίνεται ο συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, βέβαια υπάρχουν ήδη αυτές οι δυνατότητες, αλλά η όλη διαδικασία ήταν χρονοβόρα και δαπανηρή. Και υπάρχει και μια ανασφάλεια σχετικά με το πώς γίνεται η καταχώρηση σε ένα άλλο κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν πρόκυψε το εξής. Οι δυνατότητες στην αγορά εξαφανίστηκαν ή εξαφανίζονται πριν καν δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία. Μια εταιρεία ή δεν υφίστατο καθόλου ή ήταν αναγκασμένη να παραιτηθεί από συμβάσεις γιατί ο χρόνος για καταχώρηση ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα λοιπόν με αυτή την πρόταση περιορίζουμε το χρόνο καταχώρησης. Η ψηφιακή καταχώρηση πρέπει να, μπορεί να γίνεται από 5 μέχρι το πολύ 10 ημέρες. Βεβαίως ε, πρέπει να εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις, ε, ε, πρέπει να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαίως στην οδηγία εκφράσαμε κάποιες επιφυλάξεις για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου απάτης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, πολύ συγκεκριμένα, για ποιες επιχειρήσεις πρόκειται, έχω στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες στην Ευρώπη και περίπου το 80% εξ αυτών είναι κεφαλαιακές εταιρείες και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 não estava garantido à partida. Porquê? Para nós, Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ισχύουν αυστηρέ προδιαγραφέ κατά των απατών, όταν δηλαδή τα κράτη δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείε να συστήνονται με ένα απλό πάτημα του ποντικού. Εμεί δεν θέλουμε να υπάρχουν εικονικέ εταιρείε, ούτε να προάγουμε επιχειρηματικά μοντέλα που ορίζονται ω το Delaware τη Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Συγητή, την κυρία Επίτροπο, συγχαρητήρια στην διαπραγματευτική ομάδα, στην Σκιώδη Συγήτρια. Το αποτέλεσμα προβλέπει το εξή. Ο δεσμευτικό έλεγχο τη ταυτότητα των ανθρώπων που θέλουν να συστήσουν την εταιρεία ε, τα κράτη-μέλη παρά την πλήρη ψηφιοποίηση για λόγους δημοσίου δικαίου μπορούν να καλέσουν αυτά τα άτομα να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε η επιγραμμική καταχώρηση να μην γίνει ένα εργαλείο για εικονικές εταιρείε. Νέε λοιπόν προϋποθέσεις, καλύτερη πληροφόρηση, αυτά θα πρέπει να φαίνονται από τα μελλοντικά λογιστικά στοιχεία για να μπορεί να λειτουργεί και το σύστημα BRIS. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι στο μέλλον σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες έτσι ώστε να αποκλείονται κάποια στελέχη από τις εταιρείε οι απαταιώνες δεν θα πρέπει να μπορούν να εξαπατούν ε, άλλα κράτη-μέλη. Οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται την ψηφιοποίηση, αλλά η Ευρώπη δεν θα μπορεί να γίνει ένα σούπερ μάρκετ ε, ψηφιοποίηση με τις αυστηρές προδιαγραφές και με τον έλεγχο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Τα κράτη-μέλη θα μεριμνούν έτσι ώστε να μην προκύπτει κατάχρηση του εταιρικού δικαίου. Συγχαρητήρια λοιπόν για το σπριντάρισμα. Θα το χαρακτηρίσω αν μου επιτρέπετε, το οποίο κατορθώσαμε έστω και στο τέλος της θητείας αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Επόμενος πακέτ εκ μέρου του ECR. Έχετε το λόγο. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Φλάνδρα οι μικρομεσές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν και τη σποδηλική στήλη της οικονομίας. Ε, ζούνε χιλιάδες και χιλιάδες οικογένειες από αυτές. Τώρα μιλάμε για την ψηφοποίησή τους. Και μιλάμε και για το δίκαιο που όντως πρέπει να συνοδεύει αυτή την ε, ψηφιοποίηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και για να συμβεί αυτό πρέπει οι χώρες μέλη να φροντίσουν η ψηφιοποίηση αυτή να γίνει όσο γίνεται πιο απλά. Οι δυνατότητες μιας επιχειρίας να οργανωθεί ψηφιακά δεν πρέπει να επιτρέπει κανένα περιθώριο απάτης. δεν θα πρέπει να υπάρχουν παραθυράκια ώστε να μπορεί να γίνεται νομιμοποίηση, για παράδειγμα, παράνομου χρήματος. Πρέπει να βρεθούν τα μέσα εκείνα τα οποία θα εγγυηθούν για την ασφάλεια, μέσα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή οτιδήποτε άλλο για την καταχώρηση στο Μητρό. Όντως, για τις επιχειρήσεις τα πράγματα πρέπει να γίνονται πιο εύκολα, πιο απλά. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι εξοικονομούν χρήματα αλλά και γιατί θα μπορέσουν να δημιουργηθούν και περισσότερες επιχειρήσεις. Και αυτό σίγουρα θα είναι θετικό εφόσον θα γίνεται ηλεκτρονικά η καταχώρησή τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σφιεύσκα για να κλείσει τη συζήτηση, προηγουμένως η Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας όλους και πράγματι σας ενθαρρύνω να υπερψηφίσετε το κείμενο αυτό, αυτή την πρόταση. Με την νομοθετική αυτή πρόταση, όντως, καλούμε τις μικρομεσαίες και γενικά τις επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, μπορούμε τώρα να επικεντρώσουμε και τις προσπάθειές μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση θα γίνει εφικτή και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις τελευταίες του σκέψεις από αυτού και συγχαρητήρια και για το έργο σας έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο και όλους τους συναδέρφους για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται έτσι μια μεγάλη διαδικασία συνεργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Για μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συνομοθέτης, είναι προφανές ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούνται από ανθρώπου με κυριότητα, οι οποίοι δεν θα προβούν σε απάτες. Προτείνουμε λοιπόν καλές λύσεις για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους. Η καθημερινότητα είναι ψηφιακή έτσι καλλιώς σήμερα. Απάτες πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Και στην κλασική καταχώρηση δεν βλέπω γιατί τώρα να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για απάτες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις εργασίες μας και συνεισέφεραν επενδύοντας χρόνο και έργο για να ετοιμαστεί αυτή η νομοθετική πρόταση. Και προς το Συμβούλιο θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αργήσουμε να εφαρμόσουμε την οδηγία αυτή. Οι πολίτες μας περιμένουν ανυπόμονα αυτό το νομικό μέσο που είναι τόσο σύγχρονο και ελπίζω αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση. Αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Στη συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι, στην μερική διάταξη έχουμε την έκθεση τη κυρία Εύελιν Ρέγκνερ για συνοριακέ μετατροπέ, συγχωνεύσει και διασπάσει. Καταρχήν, θα ακούσουμε την εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο καταφέραμε εδώ είναι ένα ορόσημο. Η οδηγία είναι περίπλοκη, είναι πολύ διευρυμένη, έχει σχέση και μπορεί να συγκριθεί με την οδηγία περί προστασίας δεδομένων, παραδείγματο χάρη, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να συνδυάσουμε την εντολή των δύο θεσμών και να επεξεργαστούμε ένα κοινό κείμενο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, την Επιτροπή, ε, την Επίτροπο, τους και οδησηγητές, αλλά και το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν ένα νέο ε, νόμο ο οποίος ε, προβλέπει και ρυθμίζει την κινητικότητα των επιχειρήσεων και εισάγει μια ενιαία διαδικασία για τις ε, συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις των εταιριών. Ναι, πράγματι όλες οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα να μετεγκαθίστανται σε μια άλλη χώρα. Εγώ Προέρχομαι από τα συνδικάτα και θεωρώ ότι τα οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που αυτό το δικαίωμα ποτέ δεν απέτυχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, ισχύει η νομολογία, αλλά η νομολογία ήταν πέρα από τους νόμους και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο να δημιουργηθούν εικονικές εταιρείε. Γι' αυτό εμένα αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Οι εταιρείε μπορούν να ασκούν ε, το δικαίωμά τους, αλλά όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να είναι σωστά προστατευόμενοι. Μπορέσαμε να βρούμε έναν καλό κοινό παρονομαστή. Οι βασικέ προποθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμφανίζονται σε αυτή τη νέα οδηγία, καλύτερη προστασία των εργαζομένων όταν τα κράτη-μέλη μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Και επίσης ε, και μια δεσμευτική ρήτρα κατά των καταχρήσεων ε, για να μπορούμε ακριβώς να αποφύγουμε αυτές τις εικονικές εταιρείε. Ε, το θέμα του προσωπικού με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εισακούνται, να ενημερώνονται όταν πρόκειται για την ύπαρξή τους και για, και για την εργασία τους. Η σωστή ενημέρωση των εργαζομένων επιτρέπει στο μέλλον να είναι δικαίωμα η ενημέρωση των εργαζομένων για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Να υπάρχει δεσμευτική, υποχρεωτική, να υπάρχουν υποχρεωτικά διαβουλεύσεις και επιπλέον εισάγονται και νέα ε, δικαιώματα για τους εργαζόμενους ε, όταν μια χώρα μετεγκαθίσταται. Ε, οι εργαζόμενοι στο μέλλον θα έχουν μια εκτενή έκθεση στα χέρια τους για το μέλλον των θέσεων απασχόλησής τους. Θα ερωτώνται για τη μετεγκατάσταση, θα μπορούν έγκαιρα να τοποθετούνται και για πρώτη φορά αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν αιτιολογημένη άποψη από την διοίκηση. Επίσης, καθίσατε σαφές ότι οι εθνικοί κανόνες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ε, τις, ε, τους ενωσιακούς ε, κανόνες και επίσης το ότι τα εργοστασιακά συμβούλια θα πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους για να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Το θέμα του συναποφασίζει, βελτιώνεται με την πρόταση της Επιτροπής και εδώ προβλέπεται προστασία τεσσάρων ετών και αυτό ισχύει για ε, ορισμένα, για όλα τα κρατημέλη, κάτω βέβαια από ορισμένε προποθέσει. Ο δεύτερο τομέα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ απορρέει από την εργασία που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ε, φορολογικά σκάνδαλα, τα LuxLeaks, ε, τα Panama Papers και πολλά συναφή όσον αφορά την απόσποση των εργαζομένων, κυρίω στον τομέα των μεταφορών. Εκεί υπάρχουν πολύ συχνά καταχρήσει μέσω των εικονικών εταιριών. Το εταιρικό δίκαιο συστηματικά είναι αντικείμενο καταχρήσεων για να βρουν ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι τις καλύτερες συνθήκες ε, συνήθως εις βάρος στην πλάτη των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ υπερήφανη για μια δεσμευτική ρήτρα κατά των καταχρήσεων που προβλέπεται πλέον η αρμόδια υπηρεσία στην οποία το δικαστήριο πρέπει να απευθυνθεί εάν η αρμόδια υπηρεσία υποπτεύεται ότι υπάρχει κατάχρηση πρέπει να εξετάσει στις τρεις υποχρεωτικές διαδικασίες ε, κατά πόσον πράγματι τηρήθηκαν τα εθνικά και τα ε, ενωσιακά δικαιώματα, μήπως έγιναν κάποιες προσπάθειες παράκαμψή τους ή μήπως υπάρχουν άλλοι εγκληματικοί στόχοι. Εάν διαπιστωθεί ότι ισχύει κάτι από όλα αυτά, τότε δεν θα δίδεται η άδεια σε μια εταιρεία. Εάν λοιπόν μια εταιρεία τελήσει, να παρακάμψει δικαιώματα ή να συστήσει παράνομα εικονικές εταιρείες, τότε η μετεγκατάσταση απαγορεύεται. εικονικες είναι λοιπόν η ρήτρα που ισχύει και για συγχωνεύσεις και για διαιρέσεις εταιριών, αυτή η συγκεκριμένη ε, οδηγία παίρνει σάρκα και οστά. Εάν μετά την αναδιάρθρωση προκύψουν ε, ύποπτες εξελίξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. Με την κινητικότητα των εταιριών δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πλέον καταχρήσεις και εικονικές εταιρείε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα εκτεταμένο πακέτο, μία δέσμη μέτρων που μου επιτρέπει να ευχαριστήσω όλους τους και τον κύριο Ντεγκράντε και τον Πασκάλ Ντιγόν, οι οποίοι όλοι προσπάθησαν αυτή την ε, εκτεταμένη δέσμη μέτρων επιτέλους να την ε, καταστήσουν σε κάτι το απόλυτα συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με συγκίνηση, γιατί είναι η τελευταία ολομέλεια για μένα στη θητή αυτή. Συμμετείχα σε τόσε πολλέ ε, την τελευταία πενταετία και πρέπει να πω ότι εργαστήκαμε για πάρα πολλά θέματα και με την κυρία Ρέγνερ και με τον κύριο Ντεγκράντες και πάντοτε αισθανόμουν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συνέργεια πολιτικής βούλησης, ε, λογικής ε, και κατανόησης. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτό το πακέτο εταιρικού δικαίου, ε, που είναι πολύ πολύπλοκο, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και πολλοί δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε να το ολοκληρώσουμε. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος μιας πολύ δύσκολης αλλά επιτυχούς διαδικασίας. Η ευρωπαϊκή αγορά προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις εταιρείε ε, να αναπτυχθούν. Όμω, πολύ συχνά οι εταιρείε ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ωφέλη στην πράξη. Η πρόταση τη Κομισιόν απάντησε ε, σε αίτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα συνδικάτα και τι οργανώσει των επιχειρήσεων για νέου κανόνε στον τομέα αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια, την κυρία Ρέγνερ ε, και τι αντίστοιχε προεδρίε του Συμβουλίου για την υποκριτική του προσέγγιση και την αποτελεσματική του δουλειά σε αυτή την ιδιαίτερα πολύπλοκη και σημαντική σημαντική πρόταση. Χαίρομαι πολύ που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκαν ένα ρεαλιστικό και καλό συμβιβασμό που θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους υπαλλήλους. Η οδηγία θα βοηθήσει τις εταιρείες ε, να μετακατασταθούν ε, και να οργανωθούν στην ενιαία αγορά, ενώ θα παρέχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για τους ε, ενδιαφερομένους και τους υπαλλήλους. Η Κομισιόν καλωσορίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων κατά της κατάχρησης. Ήταν ένα σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Κομισιόν καλωσορίζει επίσης τις διατάξεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπου περιλαμβάνονται πολλά από τα θέματα που τέθηκαν στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κατόφλι των τεσσάρων πέτων για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, και Στι ε, τρει διασυνοριακές πράξεις. Ο υποχρεωτικό χαρακτήρας αυτών των διαπραγματεύσεων και οι διατάξει προστασία τη διαπραγματευόμενης λύση ε, ε, αν υπάρχουν και μετέπειτα πράξεις, παρέχουν ένα πλήρες πακέτο ασφαλιστικών δικλείδων. Επιπρόσθετα, το νέο άρθρο για την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών και τη διαβούλευση τονίζει και τα δικαιώματα των υπαλλήλων να έχουν λόγο σε μια διασυνοριακή διαδικασία. Και αυτό ήταν ουσιαστικό για το Κοινοβούλιο. Ε, θυμόμαστε τι αποκλίνουσε θέσει που υπήρχαν όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει. Και η Κομισιόν θα ήθελε να συγχαρεί του συνομοθέτε για τι λύσει ε, που βρέθηκαν ε, για ε, τον συμβιβασμό που αποτελεί ένα καλό βήμα προς τα μπρος σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Παρέχει εύρωστους και δίκαιους κανόνες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, που συμμετέχουν στις συνοριακές διαδικασίες, ενώ δεν είναι πολύ βαριά διαδικασία στην πράξη. Επομένως, η Κομισιόν μπορεί να υποστηρίξει πλήρως το συμβιβασμό και ανυπομονή για την αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΚΟΝ, ο κύριος Λούντβικσον, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήμουν συντάκτης γνωμοδότησης από πλευράς της Οικονομικής Επιτροπής και ετοίμασα την γνωμοδότησή μου που λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφαλείς κανόνες οι οποίοι να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις που εργάζονται σοβαρά. Συγχρόνως όμως χρειαζόμαστε και κανόνες που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε το dumping ε, στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Πρέπει να αποφύγουμε απλώς και μόνο ε, ο στόχος της μετακόμισης να είναι να αποφεύγονται οι κοινωνικοί κανόνες, δηλαδή να μην σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Ρέγνερ και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και όσους γνωμοδότησαν για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας και με το Συμβούλιο. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τώρα περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως οι νέοι κανόνες προσφέρουν και μία ενισχυμένη ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους μετόχους των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αύριο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και είναι επίσης σημαντικό να έχουμε ασφαλείς κανόνες όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως όμως να αποφύγουμε κάθε κατάχρηση, κάθε απάτη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς θα υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Μέσα από το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε περισσότερη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά. Είναι μια δικαιοσύνη η οποία θα επιτευχθεί εάν πάψουν να υπάρχουν εικονικές επιχειρήσεις. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ξεκινάμε με τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ πρώτα απ' όλα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Γιούροβα. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Συμβούλιο για το έργο του. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και φίλη μου, αν και ο αντίπαλος πολλές φορές, την κυρία Ρέγνερ. Εμείς στο ΕΛΚ στηρίξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την οδηγία, γιατί το κύριο στόχος είναι να διευκολύνεται η ζωή των επιχειρήσεων, των μικρομισών κυρίω και να μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο περίπλοκο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους, τους μετόχους κλπ. Και γι' αυτό οι νέες εναρμονημένες διαδικασίες περιλαμβάνουν και τις ρήτρε ασφάλειας για να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα όλων αυτών. Κυρίε και κύριοι, έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ελευθερία εγκατάστασης βάσει του άρθρου 49 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πάντα υποστηρίζαμε ότι οι επιχειρήσει οι οποίε εγκαθίστανται σε μια χώρα μέρο έχουν το δικαίωμα και την ελευθερία να μπορούν να μεταφέρουν την έδρα του σε άλλη χωρί να χάνουν τη νομική του προσωπικότητα. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί Μερικέ φορέ, ακόμα και χωρί οικονομική δραστηριότητα στη νέα χώρα. Θεωρούμε όμω σημαντικό, όπω και η Συγκίτροπος και το Συμβούλιο, να βάλουμε και μία ρήτρα κατά των καταχρήσεων όταν γίνονται τέτοιες διασυνοριακές μετακινήσεις πρέπει να αποφεύγουμε απάτες και κατεχρήσεις του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά, όπως ξέρει και η συγγήτρια, υπογράμμισα πάρα πολύ ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δικαιολογούνται. Δηλαδή, αν έχουν πάρει ε, κρατικές επιδοτήσεις, αν έχουν οικονομική ενίσχυση, δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα, να υποφελούνται δηλαδή από το σύστημα και να αφήνουν ξεκρέμα και τους εργαζόμενους. Αυτό θέλουμε και στην Ισπανία. Εμείς επίσης θέλουμε εξ έλεγχο της μετακίνησης για να επαληθεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία πάτη και να επικυρώνεται η δραστηριότητα αυτή μόνο εφόσον υπάρχει κατάλληλη εγγύηση για όλους. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι θετικό. Υπάρχει ελευθερία μετακίνηση που ήταν πάντα η προτεραιότητά μα, γιατί πιστεύουμε σε μια Ενωμένη Ευρώπη χωρί σύνορα. Αυτό είναι η προτεραιότητά μα και αυτή είναι και η ευθύνη μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τεγκράντες Πασκουάλ. Τώρα ε, για τους σοσιαλιστές ο Μικαέλ Ντέτζεν. Δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Κύριε Επίτροπε, με την αυρινή ψηφοφορία ε, δίνουμε τέλος σε μια παράδεκτη κατάσταση όπου οι εταιρείε θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα χωρίς να τηρούν τους κανόνες. Χωρίς κανόνες λοιπόν ήταν δυνατόν να αναζητήσει κανείς ε, βραχυπρόθεσμα κέρδος και να εγκασταθεί στη χώρα με τους ε, χαμηλότερους μισθούς και τους λιγότερους φόρους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κανόνες οι οποίοι θα προστατεύουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Η προστασία προστασία στα δικαιώματα ενημέρωση και διαβουλεύσεων. Η προστασία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στη συνάδελφό μου την κυρία Ρίγνα ε, για την επιτυχία που σημείωσε παρά τις δυσκολίες. Η πρώτη επιτυχία τη είναι ότι πλέον από μια χαόδη κατάσταση περνάμε σε μια ρυθμιζόμενη η ε, διοίκηση για πρώτη φορά είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στο προσωπικό ένα, μια λεπτομερή έκθεση ε, σχετικά με την αναδιάρθρωση της εταιρεία ε, μία ρήτρα κατά των καταχρήσεων θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν τα αίτια της αναδιάρθρωσης. Καλό και αυτό. Έτσι λοιπόν η ε, ε, εξελίξει αυτές και τα φαινόμενα των εικονικών εταιριών μπορούν να αποφευθούν τα κράτη-μέλη βέβαια δεν ήθελαν να κάνουν άλλο ένα μεγαλύτερο βήμα, έχασαν αυτή την ευκαιρία. Αλλά δεν ήταν η Ευρώπη, δεν ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών που είχαν παρεμποδίσει, που παρεμπόδισαν την καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Ε, το Κοινοβούλιο βρήκε ε, καλές συμβαστικέ προτάσει. Ε, οι προτάσει αυτέ δείχνουν το πώ μπορούμε να προχωρήσουμε και στο θέμα τη συναπόφαση. Βλέπουμε υπάρχει μια πλήρης αντίφαση ανάμεσα στα συνδικαλιστικές ελευθερίες και στα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Το κείμενο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι η καλή αρχή για ένα σύστημα κανόνων. Εγώ θα υπερψηφίσω το κείμενο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι επιγόντως απαραίτητο να υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο για τη συναπόφαση στην Ευρώπη. Επειδή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και τους συναδέλφους μου για το ότι μου τη δυνατότητα να εργαστώ και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τέτσελ και καλή τύχη. Ο κύριος Σίτερβαν τώρα για την ΚΟΕ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους εισηγητές που αγωνίστηκαν ε, κατά της φοροδιαφυγής ε, και υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά διαπιστώνω ότι ένα πολύ καλό κείμενο του Κοινοβουλίου νοθεύτηκε στον τριμερή διάλογο. Αυτό το οφείλουμε στο Συμβούλιο που δεν είναι παρόν. Υπάρχουν νέοι κανόνες ε, για το δικαίωμα εγκατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους νέους κανόνες δυσχεραίνεται η ε, άσκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ε, εμείς θέλαμε να αποφύγουμε τις εικονικές εταιρείε, ε, να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωτικότητα, καλό αυτό, όμως ε, χάνονται τα δικαιώματα των πολιτών, γίνεται κοινωνικό ντάμπινγκ, γι' αυτό λοιπόν εμείς ως αριστεροί, όπως και ο συνάδελφος, ζητάμε μια οδηγία πλαίσιο για τη συναπόφαση, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ο κύριος Βόμποντα απουσιάζει, επομένως το λόγο έχει ο κύριος Ράντεφ. Έχετε μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σήμερα συζητάμε αυτό το νομοθετική πράξη που αποτελεί μέρος του εταιρικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ρέγνερ αλλά και την Κομισιόν γιατί άκουσε την εκκλησή μας για διασυνοριακή εναρμόνιση σε περίπτωση των μετατροπών συμφωνήσεων και διασπάσεων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο κύριος σκοπός είναι να διευκολύνουμε τις ε, εταιρείε και κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν προβαίνουν σε μετατροπές, ε, συγχωνεύσεις και διασπάσεις διασυνοριακά. Η οδηγία αυτή θα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό. Ο έλεγχος καταλληλότητας, πιστεύω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υποχρεωτικά μέτρα κατά της κατάχρησης θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να σταματήσουν ε, κάποιες τέτοιες πράξεις όταν ε, έχουν ε, απατηλό σκοπό. Εδώ έχουμε διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα των πιστωτών, των μετόχων και των εργαζομένων. Οι εργαζομένοι θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τις συνέπειες των διαδικασιών αυτών και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφία και όσων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου θα προστατεύονται. Ταυτόχρονα οι πιστωτές θα έχουν ε, ξεκάθαρες ε, και αξιόπιστες εγγύησεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ράντεφ. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών δεν υπάρχει κάποιο ομιλητή για τη διαδικασια the Επομένω, Επομένως, θα δώσω τον Επίτροπο στην κυρία Γιούροβα. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρεμβάσεις σας, για τα θετικά σας σχόλια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς όσους ε, τονίσατε ότι χρειάζονται κανόνες για την καλύτερη κινητικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείε. Πράγματι αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έχουμε αυτή την ε, νομοθεσία διευκόλυνσης η οποία θα ε, παρέχει και ασφαλιστικέ δικλείδε κατά της κατάχρηση, ασφαλιστικέ δικλείδε που θα εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων των μετόχων ε, και των εργαζομένων, που θα εγγυώνται ότι δεν ε, θα έχουμε φοροποφυγή, φοροδιαφυγή ή τη δημιουργία εταιριών προπετασμάτων, εταιριών γραμματοκιβωτίου. Ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη αυτή η νομοθεσία, χρειάστηκε πολύ εμπειρογνωμοσύνη και όπως είπα και στην αρχή, χρειάστηκε και μεγάλη πολιτική βούληση. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι συνεργαστήκαμε σε ένα πνεύμα συμβιβασμού και βέβαια μας πίζει και ο χρόνος ε, στο τέλος. Είμαστε στο τέλος της θητείας μας, αλλά τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεργασία Πιστεύω ότι από κοινού παρουσιάζομαι μια καλή και ισορροπημένη πρόταση και ελπίζω ότι αύριο θα υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιούροβα. Η Ευελίν Ρέκνε τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε όποιος ε, έχει ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο ε, πρέπει να είναι μαραθωνοδρόμος με ε, ικανότητες ταχείας με ικανότητες πρινταρίσματος όπως τα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο εμείς ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια για να επιτύχουμε καλές προδιαγραφές στην Ευρώπη. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιότητα και μέχρι και το τέλος, μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας αγωνιστήκαμε για να περάσει η δέσμη μέτρων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο, ε, τους ε, διαπραγματευτές από τη Ρουμανική Προεδρία, την Καμπριέλα συγκεκριμένα, να ευχαριστήσω ε, τους ε, σκιώδης ηγητές και κυρίως και τους συνεργάτες μας. Θα ήθελα αυτό το τελευταίο λεπτό να το εκμεταλλευτώ για να πω ότι ναι πράγματι έχουμε τώρα επιτύχει πάρα πολλά και σημαντικά αλλά το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η οδηγία πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα οριζόντιο εργαλείο για τους ε, εργαζόμενους έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε και το περίφημο escalator έτσι ώστε να μπορεί να γίνει, να υπάρξει προσαρμογή ανάλογα με τις ε, καταστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε ε, και σας εισηγήτρια και την Επίτροπο έκλεισε η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Και συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη και φτάνουμε τώρα στην ε, έκθεση του κύριου Στίσλαβ Κρασνοντεύσκη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή πρώτα. Παρακαλώ. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Γιατί μετά από τρεις τριμερείς διαλόγους και ώρες διαπραγματεύσεων, καταφέραμε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια μερική συμφωνία που θα ψηφιστεί αύριο. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Εκφράστηκαν πολλοί φόβοι για το ταμείο αυτό. Φόβοι που εμένα μου φαίνεται ότι δεν έχουν καμία βάση. Αυτοί οι φόβοι, αυτές οι διαφωνίες, οι αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα κάτι το οποίο μένα με εκπλήσει. Εγώ προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, όλων των συναδέρφων του κύριου Μπούτικοφερ, για παράδειγμα, του κύριου Μαρτά, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τα επιχειρήματά τους και είχα την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι αυτοί ήταν λίγο πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θέτουν υπομφισβήτηση το κείμενο αυτό και βασίζονται ε, στα εξή δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι ηθικής και το άλλο έχει να κάνει με τη φύση της κατεξοδότησης πράξης. Το ζήτημα ήταν, όσον αφορά την ηθική πτυχή, το μήπως το Ταμείο αυτό αμφισβητεί τις σχέσεις μας με την Ατλαντική Συμμαχία, με το ΝΑΤΟ, που αποτελεί και την δομή που μα εγγυάται την ασφάλειά μας. Αυτό ερχόταν μάλλον από το αριστερό τμήμα του ημικυκλίου. Ακόμα και αν υπήρχαν ε, τέτοιες φωνές που ακούστηκαν και από το κέντρο και από τη δεξιά πτέρυγα του ημικυκλίου. Αυτά τα επιχειρήματα δεν έχουν βάση. Ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε πιστεύω ότι αναγκάζει το Συμβούλιο να σέβεται απόλυτα τόσο όσα διαπραγματευτήκαμε. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι η Επιτροπή, η Επίτροπος, είναι ικανοποιημένη και αυτή από τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Επιτρέψτε μου τώρα να παριθμίσω κάπως γρήγορα τι πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλο ότι το Ταμείο αυτό θα το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, ότι η τεχνολογία θα διακρίνεται ότι το επιπλέον κόστος δεν θα περιορίζεται, ότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις προτιμησιακές στη συμμετοχή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και εκείνες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επίσης ότι θα υπάρχουν απαιτήσει ηθικής πάρα πολύ αυστηρές για οποιαδήποτε δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο αυτό. Συνεπώς, πετύχαμε πολλά από το Συμβούλιο. Αν συγκρίνουμε, δηλαδή, ότι προβλέπεται για το Ταμείο από το ΕΔΙΤΠ αυτό που είναι, ας πούμε, για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πετύχουμε ότι επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος, αν υπάρχουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλείονται από την χρηματοδότηση. Επίσης, πετύχαμε ότι η αναφορά για στήριξη από το Ταμείο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα, για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δείχνουμε ότι το Ταμείο δεν θέλει να στρατιωτικοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να προωθήσει τις εξαγωγές όπλων. Όχι. Θέλουμε να στηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των εξοπλισμών. Και είμαι πεπισμένος ότι το Ταμείο αυτό θα επιτρέψει να δημιουργήσουμε νέα τεχνολογία και άμυνα υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που δεν καταφέραμε όμως να πετύχουμε από την άλλη μεριά εννοείται είναι μέσα στη φύση του Ταμείου, είναι η κατεξιοδότηση πράξη. Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί το Ταμείο από την αρχή του 2021. Ίσως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να αναφέρει κανείς, αλλά εγώ αυτά ήθελα να πω μέχρι τώρα. Διατηρήσαμε τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά επιχειρήματα αυτά της αριστεράς δεν στέκουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαρι... πολύ. Επόμενος ε, ε, εκ μέρους ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο πρόεδρος ο κ. Μακάλιστερ. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο κάνουμε ένα μεγάλο βήμα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα κοινά στοιχεία στην ε, έρευνα και στον, ε, στην αγορά ε, στρατιωτικών εξοπλισμών. Έτσι για να μπορούμε να οργανώσουμε την άμυνά μας. Ως εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό, ένα πράγμα κρίνω ιδιαίτερα σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θέτει τα θεμέλια για καλύτερη συνεργασία και πάνω σε αυτό ε, μπορούμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω σε θέματα ασφάλειας, ε, πολιτικής ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση των ε, εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη στρατιωτική ικανότητα και σε τελική ανάλυση μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους φόρους. Με το αμυντικό ταμείο βελτιώνουμε την αμυντική μας ικανότητα και ως εκ τούτου και την προστασία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους συναδέλφους αύριο το μεσημέρι να υπερψηφίσουν αυτόν τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, ε, κύριε Μακάλιστερ. Τώρα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Πιενκόφσκα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, για άλλη μια φορά χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία ή που μας δίνετε ευκαιρία να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Δεν υπάρχει συνεργασία για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Η πρόταση της Επιτροπής, από τότε που υπήρξε αυτή η πρόταση, είχαμε πολύ ουσιαστική δουλειά. Ε, σήμερα έχουμε μία ψηφωνία για την οποία ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αύριο τα βασικά στοιχεία του Ταμείου αποτελούν ορόσημο για την Αμυντική Ένωση. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να ευχαριστήσω την ε, διαπραγματευτική ομάδα της Ήτρε. Όλοι σας ε, είσαστε πολύ αφοσιωμένοι. Ο εισηγητή, η κυρία Γκροστέ, το κύριο Ρικέ, Μαρτάν Κόφερ και βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάω και τον κύριο Μακάλιστε. Σα ευχαριστώ όλου σα θερμά. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θα ενισχύσει την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, θα βελτιώσει την αμυντική της ικανότητα και από την άλλη ε, θα βελτιωθεί η χρήση των ε, δημόσιων κονδυλίων. Με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευαισθητοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά και να επιφέρουμε καινοτομίε ε, βελτιώνοντας ε, την τεχνολογική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος κάνοντας την Ευρώπη μια πηγή ασφάλειας, ε, όχι ε, σε αντίφαση με τον ΝΑΤΟ, αλλά συμπληρώνοντάς του. Θα περιλαμβάνονται πάρα πολλά στοιχεία Γι' αυτά αγωνίστηκε σκληρά το Κοινοβούλιο. Θα αναφέρω λίγα εξ αυτών. Τα ανέφερε ο εισηγητή, αλλά θα τα πω και εγώ από την προοπτική τη Επιτροπή. Πρώτον, οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωσης θα ισχύουν με βάση τον κανονισμό και την ενωσιακή ε, διακυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Ε, το ε, Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτό το Ταμείο. Δεύτερον, θα τεθεί το θέμα της ε, επιλεξιμότητας σε σχέση με το Ταμείο. Εδώ οι κανόνες είναι σαφείς. Μόνο οι ενωσιακές ε, εταιρείε, οι οποίες ε, σέβονται θέματα ασφάλειας στον εφοδιασμό και σε πολλούς άλλους τομείς, μόνο αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανένα, απλά ορίζουμε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή για να διασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές εταιρείε όταν ασχολούνται με έρευνα και ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. Τρίτο θέμα, συνεργασία. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του Ταμείου. Εμείς δίνουμε κίνητρα με συγκεκριμένους κανόνες, προκαλώντας και την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους αμυντικούς ομίλους, αλλά και μικρούς παίκτες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς ελπίζουμε να ανοίξουμε την αλυσίδα εφοδιασμού, την αμυντική. Τέταρτον, στο νομικό κείμενο καθίσατε σαφές ότι οι πράξεις θα πρέπει να είναι συμβατές ε, με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, όπως επίσης και με ηθικές αρχές που περιλαμβάνουν τα δίκαια αυτά. Το Κοινοβούλιο ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ε, εκφραστεί επί των θεμάτων της δεοντολογίας και επί των εμπειρογνωμόνων. Επίσης το Ταμείο αποκλεί δράσεις ε, για την ανάπτυξη θανατηφόρων όπλων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Εξάλλου, εμείς θα στηρίξουμε τις καινοτομίες το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό ε, βρίσκονται στην ίδια θέση, κυρίως αναφορά τις αποκαλούμενες disruptive τεχνολογίες. Αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Σιγητή ότι ε, θα έχουμε τις ε, εφαρμοστικές πράξεις Έχουμε ένα κατάλογο που εισήχθη για να οριστεί το πλαίσιο του προγράμματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη και πρόθυμη να έρχεται κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο για να συζητιέται το πρόγραμμα. Αυτή η προσέγγιση δεν αφορά μόνο θέματα άμυνας. Υπάρχουν και άλλα ε, προγράμματα και άλλες προτάσεις χρηματοδότησης που καταφεύγουν σε εφαρμοστικές πράξεις και που γίνονται δεκτά από το Κοινοβούλιο και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Μπιενκόφσκα. Στην ε, συνέχεια, από την Επίτροπη Προϋπολογισμών, ο κύριος Λαμασούρ. Για ένα λεπτό, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι εξ ονόματος Επιτροπής Περιπολογισμών, ε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους ε, όσους πέτυχαν αυτή την μερική συμφωνία και ιδίως την ομάδα του Κοινοβουλίου η κυρία Επιτροπό ανέφερε τα μέλη τη για την Επιτροπή Προπολογισμών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο ενωτόμα ε, έργα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια προκειμένου η άμυνα να μπορεί να αποφεληθεί από κονδύλια της Ένωσης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η συμφωνία αυτή δίνει στο πρόγραμμα όλα τα μέσα για να πετύχει τις φιλοδοξίες του και μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα μέσα του InvestEU και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αύριο θα το επιβεβαιώσει η Ολομέλη. Επίσης, χαίρομαι για το πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα που στέλνει αυτό το πρόγραμμα σε ένα τομέα που βρίσκεται στην καρδιά της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό το ταμείο μας δείχνει ότι η μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων δραστηριοτήτων στη Ένωση θα επιτρέπει να έχουμε περισσότερη ασφάλεια για να έχουμε και μικρότερο συνολικό κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμασούρ. Στη συνέχεια, εκ μέρου του ΕΛ και η κυρία Γκροστέτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο κύκλο αυτό μετά από 20 ετή παρουσία και είμαι ικανοποιημένη που μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμήνας απόψε γιατί ελπίζω ότι θα είναι ένα επιπλέον εργαλείο Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μέσω τη ανάπτυξη τη συνεργασία. Πρόκειται για ιστορική στιγμή και αποφαλούμε να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κρασμοντεύσκη και την Επίτροπο, την κυρία Μπιάνκοφσκα, που μας επέτρεψαν να πετύχουμε μια ταχεία συμφωνία ε, βέβαια, κάποιοι προσπάθησαν να κάποιοι να μπλοκάρουν ε, τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε πραγματική βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμενος και κάτι που κανείς δεν φανταζόταν δυνατό το πετύχαμε. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις και στο επόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει τον προπολογισμό των 13 δισεκατομμυρίων την περίοδο 2021-2027. Θα πρέπει να προσελκύσουμε τα καλύτερα προγράμματα και τα πιο καινοτόμα από την πλευρά των κρατών μελών και τη βιομηχανία. Αυτό το Ταμείο απαντά στις ανησυχίες των πολιτών μας για την ηθική, για την απαγόρευση των θανατηφόρων οπλικών συστημάτων. Έχουμε επιχειρήματα απέναντι σε κάποιες ειρηνικές ε, ιδεολογίες που ε, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Αυτό το Ταμείο θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ενισχύσει την αυτονομία της σε στρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μία ανεξάρτητη ικανότητα με χρηματοδότηση προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυτή η αρχή τη στρατηγική αυτονομία, είναι ζωτική σε πολλού άλλου τομεί, στο διάστημα, στην υγεία, την ενέργεια, τα τρόφιμα και βεβαίω στην ασφάλεια και στην άμυνα. Γιατί σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο θα πρέπει να βασιζόμαστε στην ένωση με τι δικέ μα δυνάμει. Έτσι θα έχουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτρέψει να προστατεύσει καλύτερα την ασφάλεια των κρατών μας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκροστέτ, και σας ευχόμαστε ότι καλύτερο στο μέλλον. Είπατε μετά από 25 χρόνια είναι η τελευταία σας παρέμβαση αυτή. Ωραία. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Εντουάρ Μαρτά, παρακαλώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως και καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο κατάφεραν να φτάσουν σε αυτήν την συμφωνία και χαίρονται, αυτό θέλανε και δεν υπάρχει κατεξουσιοδότηση πράξη. Κάτι που μπορεί να φαίνεται ένα τεχνικό στοιχείο για πολλού, αλλά όχι, γιατί είναι θέμα ελέγχου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα των πολιτών για ένα πρόγραμμα 13 δισεκατομμυρίων και για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Φυσικά και στηρίζω τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε αύριο και ιδιαίτερα το άρθρο για την απαγόρευση κάποιων όπλων, το άρθρο 11 επίσης, γιατί πράγματι δεν είναι δυνατόν απλώς να αναφερόμαστε στο διεθνές δίκαιο, γιατί υπάρχει εμφυσιμία εδώ. Για παράδειγμα, ο λευκός φόσφορος, η χρήση του για πυρομαχικά επιτρέπεται. Αν όμως χρησιμοποιηθεί χωρίς ε, διακρίσεις εμπριστικά, αυτό το καταδικάζει η ίδια σύμβαση της Γενέβης. Και έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις που έχει καταδικάσει ε, στην Γάζα, για παράδειγμα. Έπειτα, το απεμπλουτισμένο ουράνιο και εδώ, σαν όπλο, απαγορεύεται στο Βέλγιο. Δεν ρυθμίζεται όμως αλλού και ούτε αναφέρεται στο διεθνέ δίκαιο. Εφόσον λοιπόν ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται, θα έπρεπε να έχουμε ένα κατάλογο με συγκεκριμένον εξοπλισμό για τον οποίο δεν πρέπει να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, για τι εξαγωγέ όπλων. Δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυρώνει την προσέγγιση που θέλει το Συμβούλιο να είναι όλα στην διακριτική ευχέρεια των χωρών μελών. Είναι θέμα ερμηνεία. Πού είναι τα 8 κριτήρια του 2008 και η συμφωνία για την εμπορία των όπλων που έχουν επικυρώσει όλε οι χώρε. Αυτά μπορεί εσά να σα φαίνονται λεπτομέρειε, για μένα έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτά. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντέψκι, για την υπομονή του και για τη δουλειά του. Επανέρχομαι και στην ηθική αυτή τη πρόταση, τα ανέφεραν και η Επίτροπο και ο εισηγητή, αλλά πολιτικά θέλω να πω ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία θα το θυμάται αυτό. Από το 54, το 1954 προσπαθούμε και όμως δεν καταφέραμε να έχουμε την κοινότητα άμυνας και τώρα το 2019 επανερχόμαστε και προσπαθούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις αυτής της κοινότητας που απέτυχε. Τώρα λοιπόν Όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν εμπιστοσύνη, δείχνουν αλληλεγγύη. Να μην υπάρχει επικάλυψη σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης στην άμυνα, μείωση του κόστους, η οικονομία κλίμακος. Το γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο όλο και περισσότερο αβέβαιο, με μεγάλη αστάθεια, καλό είναι να μπορούμε να διασφαλίζουμε την προστασία μας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Ταμείο αυτό θα μας επιτρέψει καλύτερη ενσωμάτωση των εργαλείων των αμυντικών θα μας βοηθήσει να κάνουμε οικονομίες και θα υπάρξει και μία παρετέρω ολοκλήρωση. Κρίμα που υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες σαν στόχο έχουν να εμποδίσουν τη συμφωνία σε τριμερή διάλογο. Κι όμως είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και μας εκπλήσει που ένα τόσο σημαντικό θέμα τελικά το χειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη, σε μια περισσότερο δυνατή Ευρώπη. Ας φροντίσουμε να έχουμε μια πιο δυνατή Ευρώπη που να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους πολίτες της. Να έχουμε αυτό το αμυντικό ταμείο, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την δικιά μας την κυριαρχία, την βιομηχανική και την αμυντική και συγχρόνως να διασφαλίσουμε και την προστασία των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Στη συνέχεια, εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, έχουμε τη Μαρίσα Ματία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα και μπορείτε να μιλάτε για χρηματοδότηση, αλλά να δώσουμε 13 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα σημαίνει ότι αφαιρούμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα σημαίνει ότι θα ανταλλάξουμε την ελληνική, τη συνοχή, τα μέτρα που προστατεύουν την ποιότητα ζωή των Ευρωπαϊκών πολιτών για να επενδύσουμε σε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Οι τεχνικέ λύσει ε, δεν αποτελούν παρά ε, ουσιαστικά μια πρόφαση για την πώληση όπλων. Χρειάζονται ασφαλή Ευρωπαίοι, όμως στην απασχόληση, στις δημόσιες υπηρεσίες, σε ένα βιώσιμο μέλλον. Τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στον τομέα της άμυνας. Με τον ίδιο τρόπο, τίποτα δεν αιτιολογεί να δημιουργηθεί ε, μια νέα γραμμή του προπολογισμού ε, που ούτε καν σέβεται τα όσα εγγράφονται στη συνθήκη είναι μια πολύ ακριβή επιλογή και πολύ πιο ακριβή από τα 13 δισεκατομμύρια που έχουν εγγραφεί εδώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ματίας. Στη συνέχεια για τους πράσινους ο κύριος Μπουτικόφερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός ότι στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την κοινή ασφάλεια. Αυτό είναι το σημείο κίνησης της επιχειρηματολογίας μου. Γι' αυτό λοιπόν ένα αμυντικό ταμείο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίξει ε, θετικό ρόλο. Όμως σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις δεν πετύχαμε το εφικτό. Η επικάλυψη, η ανεπάρκεια θα εξακολουθούν να υπάρχουν στην ε, αγορά των εξοπλισμών το γεγονός ότι σπαταλήσαμε την ευκαιρία που μας προσφέρθηκε. Αυτό ε, δεν οφείλεται στον εισηγητή ε, που θέλω να τον επενέσω γιατί πραγματικά ε, είναι πνεύμα αντιλογίας, πρέπει να το πω αυτό και μερικές φορές μου έκανε και κέφι το να διαπληκτίζουμε μαζί του για το θέμα της πραγματικότητας και του ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων, από τον ε, κύριο Ρουκέ και από την κυρία Γκροστέτ ε, άκουσα ξεκάθαρα του είδα να εκπροσωπούν την, τα γαλλικά λόμπι εξοπλισμών και την ε, στρατιωτικοποίηση, της σχετική ιδεολογία. Αυτό λοιπόν που έχουμε τώρα είναι ένα αμυντικό ταμείο ε, του οποίου η δεοντολογία και οι αρχές περιοντολογίες είναι απλά μία βιτρίνα. Ένα αμυντικό ταμείο που πολύ σωστά είπε ο κύριος Μαρτά, ε, ένα ταμείο σε 7 χρόνια θα διαθέσει 13 δις. Ένα αμυντικό ταμείο που θα οδηγήσει τελικά ε, στο να έχουμε περισσότερες εξαγωγές εξοπλισμών. Ένας τέτοιος ευνουχισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι όνειδος. Αλλά παρόλα αυτά σημειώθηκε μια καλή ουσιαστική επιτυχία ότι δεν θα δοθούν χρήματα για τους, ε, για τα ρομπότ δολοφόνους. Δεν αρκεί όμως αυτό. Και γι' αυτό εμείς ε, θα καταψηφίσουμε. Κατά τα άλλα, να σας προειδοποιήσω για άλλη μια φορά όσον αφορά την ιδεολογία της ε, στρατηγικής αυτονομίας. Όποιος προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, είναι απλά εθεροβάμων. Ευχαριστώ κύριε Μπουτικόφερ. Στη συνέχεια, ο κύριος Μπουλόκ για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Πρόεδρε, προκειμένου να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή Γιούνκερ θέλει να χρηματοδοτήσει έργα άμυνος που θα κοστίζουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ τεχνολογία για τετρών, επικοινωνίες με δορυφόρους, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, εποπτεία στη θάλασσα. Συνεχίζει να εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια ολοκληρωτική ένωση και τελικά προς μια στρατιωτική. Η Κομισιόν προσπαθεί να παρουσιάσει αυτή την εξέλιξη που μια ειρηνευτική διαδικασία, όμω είναι σαφόφωνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποστηρικτέ τη έχουν έναν στρατό κατά νου. Ο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ε, ενθάρρυνε τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Στρατού πρόσφατα για την υπεράσπιση τη Ευρώπη. Πώ μπορεί κάποιο να δημιουργήσει ένα ομοσπονδιακό στρατιωτικό ε, έργο που θα συμμετέχουν 27 ε, κράτη και 24 γλώσσε, ε, όπω συνήθισε να λέει η Μάργαρετ Θάτσερ, δεν έχει χρήματα παρά τα χρήματα που κερδίζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή που, τη στιγμή που είναι σε κρίση το ευρώ και γίνονται περικοπές για την ανάπτυξη, ε, τώρα, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας τη ε, βιομηχανία ανησυχεί του πολίτε όπως και διαιρεί άνθρακα. Ένα πανευρωπαϊκός στρατός ε, θα είναι η τελευταία ευρωπαϊκή καταστροφή σε αντίθεση με τη Ρωσία ή τη ΕΠΑ. Δεν είναι ένας νέο παράγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε και την ψηφοφορία για το Brexit ε, και ε, την ε, κυβέρνηση της Ιταλίας που θα αποθαρρύνουν την περαιτέρω ομοσπονδιοποίηση. Εδώ έχουμε ένα σύνολο γραφειοκρατών που λαμβάνουν αποφάσεις για την άμυνα, για τον πόλεμο και την ειρήνη. Εμεί είμαστε κατά της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού στρατού και ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα συνειδητοποιήσουν ότι να δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Κομισιόν είναι λάθος και είναι η τελευταία μου ομιλία σε αυτό το κοινοβούλιο και ε, απευθύνω έκκληση να απομακρυνθείτε από ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος και δεν θα υπάρξει κανένα καλό από τη δημιουργία στρατού και ελπίζω ότι οι εκλογές για το νέο κοινοβούλιο θα ανατρέψουν αυτή την τάση και θα προωθήσουν το σεβασμό του έθνους κράτους και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπουλοκ Και Καλή επιτυχία για το μέλλον. Να σας ευχηθώ. Στη συνέχεια περνάμε στον κύριο Μπούζεκ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον αμυντικό πυλώνα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι η βιομηχανία άμυνας δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά είναι και η ανάπτυξη της βιομηχανίας γενικότερα στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είμαι ικανοποιημένο όχι μόνο λοιπόν για την ανάπτυξη της άμυνας, αλλά και της βιομηχανίας άμυνας. Περί τίνος πρόκειται. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για την συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεύτερον, πρόκειται για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης και πρόκειται και για ενθάρρυνση των χωρών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους σε σχέση με τις παραγγελίες και τις προσφορές. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα στην δικιά μου την περιφέρεια. Έτσι θα μπορέσουμε, πιστεύω, σύντομα να κάνουμε τους Ευρωπαίους να υποφεληθούν από τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα έχουν δημιουργηθεί από τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις της δικιάς μου περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντεύσκη, ο οποίος πάρα πολύ καλά βοήθησε στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συνεισηγητές, όπως επίσης και την κυρία Γκροστέτ, η οποία ήταν προηγουμένως η συγγήτρια της δικιάς μας έκθεσης για το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πούσεκ, ο επόμενος, ο Βίκτορ Μποστινάρου. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. κυρία Επίτροπε, να ξεκινήσω από εσά. Σα ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τον εξαιρετικό τρόπο που διαπραγματευτήκατε σε ένα κόσμο που έχουμε αστάθεια και πολλές ευρυδικές και νέες απειλές. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παγιώσει το ρόλο της ως παγκόσμιο παίκτη που θα ασκεί επιρροή. Σήμερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για όλους τους πολίτες μας και ε, ε, γι' αυτό βρήκε απήχηση. Η ανάπτυξη της ε, κοινή πολιτικής άμυνας είναι μία από τις κύριες συνεισφορές στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκόπος της νομοθετικής πρότασης που έτυχε διαπραγμάτευσης με το Συμβουλίο είναι να ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας στα πλαίσια του πολιετου δημοσιονομικου δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, έτσι ώστε να απαντήσει στις αυξανόμενε προτεραιότητες της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να να αρχίσουμε να ε, απαντάμε στον κατακαιρματισμό του τομέα της άμυνας και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, να ενθαρρύνουμε την συνεργασία ε, και την κοινή απόκτηση εξοπλισμών. Επίσης, όπως ε, ανακοινώθηκε, είχαμε κύριες προτεραιότητες κλειδί της δικής μου πολιτικής ομάδας για το τομείο αυτό. Εμείς αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αμυντική βιομηχανία και στην πρόθεση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ε, για ε, τα μέσα άμυνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι να υπογραμμίσω την ανάγκη να συνεχίσουμε τη διαδικασία της ε, προώθησης μιας παγκόσμιας τάξης βάσει κανόνων, έτσι όπως αναφέρεται στην Χάρτα 1 και να παγιώσουμε τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, καθώς αυτό αποτελεί τη μόνη εγγύηση ασφάλειας στην Ήπειρό μας είχα την, ε, το προνόμιο να εργαστώ στο φάκελο αυτό τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να σας συστήσω να υπερψηφίσετε αύριο και καθώς αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο κοινοβόλιο, επιτρέψτε μου να πω σε όλους σας ευχαριστώ καρδίας για αυτά τα 12 χρόνια τα οποία εργαστήκαμε για το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Κυρία Γκροστέτ, ας ε, παραμείνουμε ειρηνικοί αλλά ποτέ αγαθοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 13 δισεκατομμύρια ευρώ τόσα ε, θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ε, μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων σε 7 χρόνια. Αυτά αφαιρούνται από τις επενδύσεις στην καταπολέμηση στόχια, την πρόθεση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Είναι πόροι που θα προωθήσουν τώρα τον πόλεμο, θα χρηματοδοτήσουν την εξοπλιστική βιομηχανία, τροφοδοτώντας μια κούρσα στρατιωτικοποίησης. Ε, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ανοίγεται και την πότρη του προγράμματος έρευνας ε, για, όχι αποκλειστικά για ε, και μη στρατιωτικούς σκοπούς και ε, θα χρησιμοποιήσετε τα δίκτυα μεταφορών για τη στρατιωτική κινητικότητα. Όποιο προωθεί τον πόλεμο και τροφοδοτεί αυτή τη βιομηχανία δεν μπορεί να πετύχει την ειρήνη. Έτσι λοιπόν αυτή η νομοθεσία δεν σέβεται ε, τους λαούς. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο συνεργασίας που να έγκυται στις ε, αξίες της Ειρηνή. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φεραίρα. Και τώρα ο κύριος Κοφέρ έχει θέσει μια μπλε κάρτα. Δέχεστε παρακαλώ. Κύριε Φερέιρα, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Σας μιλώ φιλανδικά. Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερέιρα, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι στραφήκατε κατά της ε, στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε ότι η δική σας η πολιτική ομάδα, η ΓΚΟΕ, σε όλες αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις των πολλών μηνών δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά ένας έστω ευρωβουλευτής για να συζητήσει. Και ε, δεν καταλαβαίνω πώς τολμάτε να στρέφεστε κατά του μιλιταρισμού και δεν έχετε κάνει τα μαθήματά σας. Κύριε φέρα αύριο θα επιβεβαιώσετε ότι δεν θα είναι με την υποστήριξη αυτή τη ομάδα που αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα που θέλει να διαθέσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στην εξοπλιστική μηχανία θα εγκριθεί. σω ε, με κάποιε ψήφου από τη δική σα πλευρά, δεν ξέρω, θα δούμε. Σίγουρα με τι ψήφου τη Σοσιαλδημοκρατία και όλη δεξιά. Και φυσικά δεν αγνοώ τη σύνθεση αυτού του οίκου, όπω και εσεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι θέσει μα είναι μη ψηφικέ ακόμη. Και λέω ακόμη γιατί νωρίτερα ή αργότερα νωρίτερα και μάλλον νωρίτερα θα είναι πλειοψηφικέ ε, απόψει ε, και εμεί θα ανατρέψουμε αυτή την κούρσα εξοπλισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι εσεί κάπω έχετε ανεχθεί στο παρελθόν αυτέ τι ε, στρατιωτικέ περιπέτειε. Yeah. sitten edustaja Inrik Taran saa puheenvuoron, niin hänellä on minuutti. Olkaa hyvä, edustaja Taran. Ο κύριος Ταράν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον ε, συνάδελφό μου, κύριο Μπίτι Κόφα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι παρότι άσκησε κριτική κατά αυτής τη πρόταση και σωστά έπραξε, φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι το Ευρωπαϊκό Αμαντικό Ταμείο έρχεται ε, πολύ καθυστερημένα και είναι και πολύ λίγο γιατί δεν κατορθώσαμε να νομοθετήσουμε για να υπάρχει μια, ε, ε, ένας ευρωπαϊκός στρατός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα υποστηρίζω την έκθεση όσον αφορά την αίρεσιμότητα, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Ε, προς τον κύριο Μπούλοκ ε, θα ήθελα να πω ότι ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Στρατός ε, θα υπάρξει, θα μιλάει αγγλικά. Δυστυχώς λόγω αυτής της περιπέτειας του Brexit δεν θα υπάρξει Βρετανός διοικητής, αλλά θα υπάρξει αυτός ο στρατός. Και προς τον κύριο φαρέρη, θέλω να πω ότι τα τρία δις είναι τίποτα, ψίχουλα. Ακόμα και ο προπολογισμό ε, της ε, Λετωνία είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία αύριο για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο έρχεται στο τέλο μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που μα οδήγησαν μέχρι εδώ. Εγώ ήμουν και ο εισηγητή, αλλά θέλω να ζητήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ελέγχει ε, την ε, εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου. Αύριο δεν είναι το τέλο, αλλά είναι η αρχή μια ε, νέα αμυντική πολιτική. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να είναι παίκτη και όχι παρατηρητής. Εγώ ήμουν υπέρ και γενικά η δική μας ομάδα ήταν υπέρ των ε, κατεξοδότηση πράξεων. Ορισμένες τροπολογίες ε, πέρασαν το, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να υψώνει τη φωνή του για να υπάρχει ένα ε, όραμα πραγματικά ευρωπαϊκό που θα επιτρέπει τρία στάδια με πνεύμα του ανταγωνισμού θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, τεχνολογίες μας. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να μην υπάρχουν ε, άμεσες απευθείας αναθέσεις. Ε, εμείς έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις για κάποια κριτήρια, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν χωρίς τιμωρητική διάθεση. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρηματοδοτεί λάθους δεν θέλουμε να υπάρχει συνεργασία με άλλους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά την παραγωγή και την έρευνα. Δεν θέλουμε ε, να διαταράσσεται η αλυσίδα παραγωγής ε, με το να αποκλείονται κάποιες χώρες. Ε, επίσης δεν θέλουμε σε τελική ανάλυση αυτό το ταμείο να ε, χρηματοδοτεί θανατηφόρα όπλα χωρίς ελεγχό η πρόεδρο διακόπτη. Ο κύριος Καστάντο μιλάει με ένα ρυθμό απίστευτα γρήγορο. Πάση περιπτώσει, θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα για έναν ευρωπαϊκό στρατό, ακόμα και εάν ε, ε, αναφέρονται οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου στις συνθήκες. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αυτό το ταμείο, ένα ταμείο το οποίο θα διευκολύνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα διευκολύνει την άμυνα και την ε, ασφάλεια, ένα ταμείο το οποίο δεν θα στρέφεται κατά άλλων, αλλά ούτε θα θέλει να προστατεύει ιδιαίτερα κάποιους, ένα ταμείο το οποίο θα είναι ανοιχτό για άλλες συνέργειες. Τέλος, το ταμείο αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα κενά, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι τελικοί χρήστες ε, θα είναι οι δικοί μας οι άντρες ε, και οι γυναίκες ε, και όλοι εκείνοι που βρίσκονται και σε καθεστώς πολέμου. Πρόεδρος, κοιτάξτε, οι διερμηνείς πραγματικά τώρα εξεπέρασαν τον εαυτό τους, γιατί δεν υπάρχει και όριο στην ταχύτητα. Μιλάτε τόσο πολύ γρήγορα. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο, πιο αργό ρυθμό, λέει η πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκάλερ. Παρακαλώ κύριε Γκάλερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά έτσι ώστε οι πολίτες μας να προστατεύονται από εξωτερικές απειλές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό το ταμείο ε, για να μπορεί να αξιολογηθεί η ασφάλεια και να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το βρίσκω πάρα πολύ λυπηρό το ότι κάποιοι από αριστερά αλλά και μέχρι δεξιά ε, δεν θέλουν να προσφέρουν αυτή την καλύτερη προστασία στους πολίτες μας. Αυτό είναι ολιγορία. Ολιγορία κατά των πολιτών μας που τους αξίζει καλύτερη άμυνα ολιγορία και έναντι των στρατιωτών μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη στο Μαλί, ε, στη Σομαλία, στη Μεσόγειο υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας. Έχουν το δικαίωμα να έχουν τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίζουν υγιείς στις πατρίδες τους. Τέλος, αναφέρομαι στο Συμβούλιο και στα μεμονωμένα και στην Επιτροπή. Στο μέλλον εσείς θα κληθείτε να αποδείξετε δείξετε ότι τα 13 δις που προβλέπονται για τον αμυντικό αυτό προπολογισμό θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού για αγορές, ε, για εξοπλισμούς, ε, για βελτίωση τη ικανότητας. Τώρα πρέπει να αποδείξετε ότι ε, τα 210 δις ευρώ στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται καλύτερα οι πρωτεύουσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και όχι να θέλουν να καταφύγουν σε προγράμματα όπως το ΕΦΚΑΣ ή τα τεθωρακισμένα μάχης. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες μας τελικά τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Από το σύνθημα στρατηγική αυτονομία θα πρέπει να περάσετε σε μια συνεπή αμυντική πολιτική, πολιτική εξοπλισμών, έτσι ώστε οι πολίτες μας και η βιομηχανία μας να κατανοούν περί πρόκειται. Ε, το ταμείο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι το, μόνο το πρώτο βήμα και κατά τα άλλα θα χαιρόμουν πάρα πολύ ε, το πώς θα, να δω πώς θα ψηφίσω ο κύριος Μπούλμαν από τον πρόεδρο ε, μια τόσο μεγάλη πολιτική ομάδα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, μπορεί κανεί να περιμένει και μια προσωπική τοποθέτηση. Ο κύριος Ροζάτης στη συνέχεια για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα συζητάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ασφάλεια της Ευρώπης, ε, μια αγορά δημόσιων κονδυλίων ε, για την απόκτηση αμυντικών μέσων. Αυτό είναι κατακαιρματισμένο ε, στην Ευρώπη. Μόλις το 16% αυτών των ε, δημόσιων διαγωνισμών υλοποιούνται από δύο ή περισσότερα κρατημέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επίπεδο συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο. και φυσικά ε, η ασφάλεια αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας και υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις ε, όπως η επιθετική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ο μουσουλμανικός ε, εξτρεμισμός και απαιτούν να ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ακριβώς αποτελεί ένα μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία στο βιομηχανικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη του κλάδου στα κράτη-μέλη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει 13 δισεκατομμυρία ευρώ. Ένα ποσό που θα επιτρέψει την ενίσχυση των ικανοτήτων ε, στην έρευνα και στην κοινοτομία στον αμυντικό κλάδο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην κατανομή των κορτιλίων ε, για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε το δυναμικό όλων των χωρών και αναφέρομαι και στις μεγάλες χώρες αλλά και στη χώρα μου στην Πολωνία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωσάτη. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Κατσδιάη. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Πόσπεσιλ πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσωπικά όλη τη συζήτηση και θα την στηρίξω. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Αυτές οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό γενικότερα για την οικονομία. Τέτοια προγράμματα δεν είναι δυνατόν βέβαια να απειλούν τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να αποτελούν μια εναλλακτική λύση διαφορετική από το ΝΑΤΟ. Εμείς στην Τσεχία πιστεύουμε ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασίας. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση, αλλά η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ να ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Πρώτα, ευχαριστούμε κύριε Πόσπισιλ. Ο κύριος Μαριάς τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 13 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, την εκπαίδευση, την κατάρτιση την αντιμετώπιση της φτώχειας. θεωρώ ότι αυτό το ποσό επί της ουσίας θα μπει στην υπηρεσία των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών της ευρωπαϊκής ένωσης που ως γνωστόν πουλάνε όπλα ακόμη και στην τουρκία ακόμη και στη σαουδική αραβία. στην πράξη τι γίνεται; ζήτησε ο τραμπ να βάλει η ευρωπαϊκή ένωση το χέρι στην τσέπη για τα θέματα της άμυνας. αυτό είναι όλο το θέμα. και πλέον ερχόμαστε να υπηρετήσουμε αυτή την πολιτική μετατρέποντας σε όλο και πιο στρατιωτικοποιημένη την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση και γι' αυτό αυτό που θα συμβεί στην πράξη είναι να γίνονται όλο και πιο πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης στον τρίτο κόσμο. θεωρώ ότι τα κονδύλια αυτά πρέπει να πάνε κυρίως για τη στήριξη της ίδιας της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Παρακαλώ. Κύριε Σόσνιερτς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε αυτά που είπε ο καθηγητής Κρασνοντεύσκη, ότι πρόκειται για ένα παραπάνω βήμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας. Και αρκεί να ακούσουμε την κυρία Κροστέτ για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία σε βάθος ολοκλήρωση. Καταλαβαίνω ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να πετύχουν περισσότερα. Χάσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε τώρα βρίσκονται στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και δρούν ανάλογα. Πώς όμως θα υποφεληθεί η Πολωνία. Ουσιαστικά καταστρέφουμε την ανεξαρτησία μας. Χάνουμε τον έλεγχο του δικού μας ε, στρατού. Η έρευνα και ανάπτυξη που μπαίνουν ε, σε κοινό πλαίσιο σημαίνει ότι χάνουμε τον έλεγχο της δικιάς μας έρευνας και ανάπτυξης. Τι θα γίνει στις χώρες οι οποίες τελικά δεν θα έχουν το δικό τους στρατό. Φτιάχνουμε ένα τέταρτο ράιχ της Γερμανίας. Πρόεδρος, τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, εξότιμοι ευρωβουλευτές, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τίποτα δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή, δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους που με τόση αφοσίωση προσπαθήσετε να ε, καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Σε δύο πτυχές θα αναφερθώ μόνο. Πρώτον, για τη συνεργασία, γιατί πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο ποσό, στα χρήματα. Θέλω να σας πω και πάλι ότι η έλλειψη συνεργασίας στον τομέα της άμυνας κοστίζει και το κόστος αυτό είναι ανάμεσα στα 25 με τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, επειδή δεν υπάρχει συνεργασία στον αμυντικό βιομηχανικό τομέα. Έπειτα, για την εξαγωγή όπλων, επειδή κάποιοι από εσά το έθεσαν. Και εδώ είναι σαφές το θέμα. Έχουμε συζητήσει πολύ γι' αυτό. Είναι καθαρά αρμοδιότητα των χωρών μελών. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα με τον κανονισμό. Δεν αυξάνουμε την εξαγωγή όπλων. Αυτό που θέλουμε και αυτή που είναι η πρόθεσή μας είναι να μειωθεί η εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Η τεχνολογία μας να μην εξαρτάται από τρίτες χώρες. Η συνεργασία θα βοηθήσει σε αυτό. Η μείωση της τεχνολογικής μας εξάρτησης είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου αυτού και είμαι σίγουρη ότι η άμυνα θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μιλάμε ακόμα για την ε, αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαίρεται για την συμφωνία ε, στην οποία καταλήξαμε μετά τους τριμερείς διαλόγους και ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί η πρόταση αυτή. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους, τον εισηγητή, τους σκιώδες εισηγητέ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, τον κύριο Μπούτσεκ, γιατί είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή δουλειά. Δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία είναι ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο ε, και τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία κατέδειξε ότι δεν ε, συμπίπτουν οι απόψεις μας. Στους σοσιαλδημοκράτες ε, εκφράστηκαν από πλευράς τους διαφορετικές απόψεις ε, και στο επίπεδο των, στο μέτωπο των πρασίνων και εκεί διαφορετικές απόψεις. Ε, υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Υπάρχουν κράτη όπου δεν υπήρξαν εισβολές, ε, ούτε κατοχή εδαφών. Από την άλλη όμως υπάρχουν κράτη όπως οι χώρες της ε, Βαλτικής ε, και χώρες ε, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που εξακολουθούν να αισθάνονται υπό απειλή. Ναι, καλά τα κοινωνικά προγράμματα, αλλά αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία, τότε προφανώς και κινδυνεύει η κοινωνική μας ευημερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αυστριακή και τη Ρουμανική Προεδρία γιατί δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και ε, επέδειξαν ε, ιδιαίτερη τεχνογνωσία και όσοι φοβούνται το θέμα των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ, να τους πω το εξής. Κοιτάξτε, στη δική μας την περιοχή ξέρουμε πολύ καλά τι είπατε. Είμαστε υπέρ αυτού του ταμείου, αλλά είμαστε και υπέρ του ότι το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφαλειά μας είναι ο εγγυητής της ασφαλείας μας. Επ' αυτού δεν αλλάζει τίποτα. Και θα θέλαμε άλλες χώρες, η Γαλλία Παραδείγματο χάρη, να δραστηριοποιηθεί για την προστασία της ε, ανατολικής πτέρυγας ε, του ΝΑΤΟ. Ε, Τέθηνε ερώτημα από τι ή πώς θα ωφεληθεί η Πολωνία. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε αν συνεργαστούμε να εξυγχρονίσουμε τον, ε, τους εξοπλισμούς, τη βιομηχανία εξοπλισμών ε, και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω ε, τα κονδύλια αυτού του ταμείου να διατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπερψηφίσετε το κείμενο όπως ακριβώς ε, το διαπραγματευτήκαμε. Παρακαλώ να απορρίψετε όλες τις τροπολογίες υπέρ του 31CP και υπέρ όλων των ε, τροπολογιών της ε, Ολομέλειας, γιατί αλλιώς θα καταπέσει η συμφωνία μας. Αυτή είναι η θερμή μου παράκληση προς όλους σας. Το γεγονός αυτό, όπως σας είπα, το έχω ενστερνιστεί, γιατί αποτελεί ευκαιρία για την αμυντική βιομηχανία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και για την βελτίωση των αμυντικών μας ικανοτήτων που είναι πολύ σημαντικές. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να επερασπιστούμε τον τρόπο ζωής μας και τον πολιτισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, συγχαίρω και ευχαριστώ τον ομιλητή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Τώρα προχωράμε. Κοινή συζήτηση για τα καλυμμένα ομόλογα. Έκθεση του κυρίου Μπέρντ Λούκε και θα ακολουθήσει και μία άλλη συζήτηση για τα καλυμμένα ομόλογα και τα η δημόσια εποπτεία. Είναι δύο εκθέσεις του κύριου Λούκε. Κύριε Λούκε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για κάθε κεφαλαία αγορά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ασφαλή, ασφαλείς κινητές αξίες. Γνωρίζουμε δυστυχώς βέβαια ότι αυτό σπανίζει. Γνωρίζουμε ότι οι τιτλοποιήσεις δεν προσφέρουν επαρκή κάλυψη. Αυτό το γνωρίζουμε το αργότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι και τα κρατικά ομόλογα δεν προσφέρουν επαρκή προστασία. Ούτε και αυτά της Ευρωζώνης. Δεν είναι ικανοποιητικά ασφαλή. Όπως σας είπα, το συνειδητοποίησαμε και με την κρίση του ευρώ και του δημόσιου χρέους. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν ε, τα καλυμμένα ομόλογα, ότι αυτά είναι ασφαλή τα καλυμμένα ομόλογα υπάρχουν εδώ και πάνω από 250 χρόνια και μέχρι τώρα ε, δεν έχουν καταρρέψει. Πρόκειται για μια κινητή αξία που την χρειαζόμαστε στην Ευρωζώνη και στην κεφαλαγορά. Γι' αυτό λοιπόν εκπλήσει το γεγονός ότι τα καλυμμένα ομόλογα δεν έχουν εξελιχθεί επαρκώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχει μόνο μία μικρή ομάδα κρατών που έχουν αυτή την παράδοση των καλυμμένων ομολόγων και την χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν σχεδόν καθόλου εμπειρία από καλυμμένα ομόλογα και δεν έχουν και σχεδόν καθόλου νομοθεσία για αυτά. Αυτό προσπαθούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε εκδίδοντας ή ε, θεσπίζοντας, ψηφίζοντας οδηγία και κανονισμό για τα καλυμμένα ομόλογα. Η οδηγία είναι παράλληλα και το οδηγό νήμα για τις εξελισσόμενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τα καλυμμένα ομόλογα επιτυγχάνουν και αποκτούν ένα αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν να μεταφέρουν στην νομοθεσία τους αυτό που έχει αποδειχθεί σωστό εδώ και πολύ καιρό και που είναι μια πρακτική, δοκιμασμένη πρακτική στο θέμα των καλυμμένων ομολόγων. Όσον αφορά την νομοθεσία, πραγματικά προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά που αναφέρουμε, που πιστεύουμε για τις κινητές αξίες, όλα αυτά ε, για τα οποία διαπραγματευτήκαμε και νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα έχει τώρα λάβει τέτοια μορφή έτσι ώστε να έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες καλυμμένων ομολόγων. Αφενός εκείνα τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία ορίζονται στον κανονισμό ε, περί επάρκειας κεφαλαίων ομόλογα τα οποία προσέλκυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι είναι τα καλυμμένα ομόλογα υπό εξέλιξη, εκείνα που θα προσφέρουν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, θα εξετάσουν νέες δυνατότητες εξασφαλίσεων. Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ καλές συνθήκες πλαίσιο, έτσι ώστε τα καλυμμένα ομόλογα να επικρατήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ικανοποιητικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο και αυτές οι κινητές αξίες να γίνονται αποδεκτές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε να θέσουμε πρότυπα σε διεθνές επίπεδο για αυτό το χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την εμπιστοσύνη των ε, ε, πιστωτών και των ομολογιούχων. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και το ενδιαφέρον των οντοτήτων ε, των εκδότριων οντοτήτων έτσι ώστε να ανοίξει η αγορά μας και να μην κλείσει έναντι εκείνων οι οποίοι επίσης ενδεχομένως ενδιαφέρονται για τη χρήση αυτού του εργαλείου. Νομίζω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σήμερα προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία και βεβαίω θέλω να ελπίζω ότι αυτό το εργαλείο θα γίνει ευρέω αποδεκτό στην Κεφαλαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μπιερκόφσκα, παρακαλώ. Μικρόφωνα παρακαλούμε. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μια σταθερή πηγή και αποτελεσματική προ το κόστο πηγή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια τη κρίση. Ανταποκριθήκαν καλά είναι πάρα πολύ δημοφιλή σε κάποια κράτη-μέλη, ενώ σε κάποια είναι κάτι καινούριο. Η πρόταση Κομισιόν προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω αυτή την αγορά, βασιζόμενη στα υψηλά πρότυπα και τι καλέ πρακτικέ των εθνικών συστημάτων. Ε, πρόκειται για ε, ένα βασικό ε, στοιχείο τη αγορά κεφαλογορών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πανευρωπαϊκή αγορά ομολόγων που θα υποστηρίζει το δανεισμό στην πραγματική οικονομία, χωρί να ενοχλεί ήδη τι εθνικέ σε αγορές που λειτουργούν καλά θα υπάρξει όθηση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων στα κράτη-μέλη όπου είναι λιγότερο αναπτυγμένες αυτές οι αγορές. Οι κανόνες αυτές ε, θα σημαίνει ότι ε, θα υπάρχουν ασφαλή εργαλεία για τις τράπεζες που θα επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουν τις εταιρείε και τα νοικοκυριά. Εκτιμούμε ότι η πιθανή εξοικονόμηση για τους δανειστές θα είναι περίπου 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, θέλει η Ένωση να εναρμονίσει τους κανόνες προληπτικής εποπτείας ε, προκειμένου να συνεισφέρει Φέρουμε στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο πυλώνε. Καταρχήν σε μια οδηγία που παρέχει ένα κοινό ορισμό των καλυμμένων ομολόγων, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των μέσων και εντοπίζει ε, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλή ποιότητα που μπορούν να επιλεχθούν για να καλυφθούν από καλυμμένα ομόλογα. Επίση, έχουμε και την οδηγία για την εποπτεία ε, και θέτει του κανόνε για τις ε, ετικέτε. Και ο δεύτερο νομοθέτημα, ο ενισχύει του κανόνε για πρώτα μισή μεταχείριση που θα, θα καλύπτουν τα ομόλογα που αγοράζονται από τράπεζε. Όπω ε, είδαμε στου τριμμέ διαλόγους και έχουμε και στη δήλωση τη ε, Κομισιόν, η Κομισιόν θέλει να τροποποιήσει την ε, αναλογία για την κάλυψη ρευστότητα για να ρυθμίσει τα καλυμμένα ομόλογα. Αυτό θα, καλύψει, θα αντιμετωπίσει συγγνώμη, την επικάλυψη μεταξύ του ε, του αποθέματος ρευστότητας ε, αποθέματος αλλιές ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία. Ε, θα στείλουμε αυτά τα στοιχεία στο Κοινοβούλιο πριν από την ευρενή ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την επιτυχή για το επιτυχές αποτέλεσμα και κυρίως τον εισηγητή και όλους τους κοιόδες εισηγητές. Ο στόχος της πρότασης της Κομισιόν ε, διατηρούεται χάρη στην επικοτομητική προσέγγιση της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου και της καλής συνεργασίας με το Συμβούλιο. Η μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο και εφαρμογή των νέων κανόνων για τα καλυμμένα ονόλογα θα πρέπει τώρα να προχωρήσει γρήγορα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχουμε μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη προωθώντας τις ε, θέσεις εργασίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ροζάτη. Παρακαλώ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εργαζόμαστε πάνω σε δύο έγγραφα, τα οποία ε, δημιουργούν νέες αρχές λειτουργίας για τα καλυμμένα ομόλογα. Πρόκειται για εγγυημένα ομόλογα και είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο δημιουργεί μια κεφαλιακή ένωση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. Αυτά τα εγγυημένα ομόλογα ορίζονται δίνεται ορισμό του στο έγγραφο αυτό. Και τι είναι, είναι μια εγγύηση. Επίσης έχουμε δύο κατηγορίες εγγύσεων. Έχουμε τις ευρωπαϊκές που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και έχουμε τις premium, οι οποίες επιπλέον καλύπτουν και τις απαιτήσει του κανονισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, του CRR. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί από μόνη της να αποφασίσει για το πούλο του ενεργητικού και για το ρευστό. Καταλήξαμε σε ένα συμβασμό το 8% εγγύσεων για την ποιότητα των πιστώσεων. Επίσης υπάρχουν οι τραπεζικές εγγύσεις που γίνεται ένα έγγραφο υψηλής ποιότητας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον βουλευτή, τον Ευρωβουλευτή Λούκε για την εξαιρετική αυτή έκθεση, αλλά επίσης και για την καλή συνεργασία που είχαμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική της συμμετοχή. Ζητώ από όλους τους Ευρωβουλευτές να υπερψηφίσουν χωρίς τροπολογίες αυτή την έκθεση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Σαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς για τα καλυμμένα ομόλογα, όπως ονομάζονται. Η διαδικασία ξεκίνησε εδώ το 2017 με μια έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία θέσε και τις βάσεις του έργου μας για το νομοθετικό πακέτο που σήμερα έχουμε μπροστά μας. Δεν ήταν εύκολο, γιατί στην κάθε χώρα τα καλυμμένα ομόλογα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Αποτελούν ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του κατά τους αιώνες έχουν βέβαια αναπτυχθεί διαφορετικά στις διάφορες εθνικές αγορές, αλλά έχουν νόημα. Και σε κάποιες αγορές όπως στη Δανία και τη Γερμανία τα καλυμμένα ομόλογα θεωρούνται ένα μέσο επενδυτικό πάρα πολύ συνηθισμένο. Σε άλλες χώρες όπως τη δικιά μου τη Μάλτα δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχει εδώ λοιπόν μια πολιτική πρόκληση μπροστά μας για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην ε, αγορά, ε, την, ε, μάλλον την ένωση της κεφαλαϊκής αγοράς. Ε, θα έπρεπε όμως να αποφασίζονται όλα από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ή θα έπρεπε να δεχτούμε τις διευθετήσεις που έχουν γίνει στις εθνικές αγορές μέχρι τώρα και που έχουν αποδείξει την αξία τους. Εγώ θα συμφωνούσα με το δεύτερο. Ε, δεν πρέπει να αλλάξουμε πράγματα τα οποία έχουν λειτουργήσει για δεκαετίες, για αιώνες ε, ικανοποιητικά. Βέβαια, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να δημιουργηθεί με στόχο την προδευτική σύγκληση προς παρόμοιους κανόνες και πρακτικές. Το σεβαστικό κείμενο που έχουμε μπροστά μας ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την πρόκληση. Περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής ΕΚΟΝ του 2018 και διορθώνει διάφορες πτυχές που θα ήταν μια ανησυχία για την ομάδα μου. Το κείμενο λοιπόν προωθεί την αναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενισχύει την διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, ενώ συγχρόνω αποφεύγει τον κίνδυνο ανατροπή των επιτυχημένων εθνικών συστημάτων καλυμμένων ομολόγων. Χαίρομαι που αυτέ οι προτεραιότητε αντικατοπτρίζονται στο κείμενο και κάνω έκκληση στο Σώμα να εγκρίνει αυτήν την πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Πόση ώρα έχω κύριε Πρόεδρε. How much time I have, Mr. Chairman? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 30 seconds. Thank you. Και 30 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για αυτού του είδους τα ομόλογα όταν φυσικά έχουν δει όλοι ότι ακόμη και κρατικά ομόλογα έχουν καταρρεύσει. Ιδίως στην πατρίδα μου όπου τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τα οποία εμπιστεύτηκαν οι έλληνες πολίτες πάρα πολλοί μικρομεσαίοι συνταξιούχοι επένδυσαν τις, ε, τους κόπους μιας ζωής στα ελληνικά ομόλογα και ήρθε μετά το περίφημο psi με απόφαση του eurogroup και κουρεύτηκαν τα ομόλογα αυτά κατά 53%. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι στην Ελλάδα που είχαν εμπιστευτεί τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που δεν έχουν πλέον χρήματα να πληρώσουν τα φάρμακα να μπορέσουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουν καταρρεύσει τα κρατικά ομόλογα υπάρχει δυσπιστία απέναντι σε αυτή τη μορφή ομολόγου και φυσικά όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο κύριος λούκε κάνει προσπάθεια η εισήγηση αλλά βεβαίως και ο κανονισμός να υπάρξουν οι μέγιστες εγγυήσεις ούτως ώστε αυτά τα ομόλογα να θεωρηθούν ασφαλή να έχουν φυσικά και πολλούς επενδυτές και έτσι να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο το οποίο θα διαμορφώσει μια συνολική αγορά και ταυτόχρονα θα πάρει κοντά του και αρκετούς επενδυτές. όμως θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα γίνουν αυτές οι διασφαλίσεις ούτως ώστε πραγματικά να μην φτάσουμε σε σημείο να καταρρεύσουν ακόμα και αυτά τα ομόλογα. όλα φυσικά κρίνονται από το πώς θα λειτουργήσει η αγορά. αν υπάρχει μεγάλη κρίση τότε πολλοί διερωτώνται αν και αυτά τα ομόλογα θα αντέξουν. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ναχτεγάλ τώρα. Η κυρία Ναχτεγάλ δεν είναι εδώ όμως. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρολτ. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή που βρήκε με ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση. Η συμφωνία για τους κανόνες σε ό,τι αφορά τα καλυμμένα ομόλογα εντάσσονται σε μια λογική που θέλει να ενισχύσει την Ένωση Κεφαλαγορών. Είναι ουσιαστικό να μην χάσουμε το στόχο έσχατος σκοπός του νόμου που υθετούμε Στη συγκεκριμένη περίπτωση ουσιαστικά πρόκειται για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας. Βεβαίως προσπαθούμε να φέρουμε στις τράπεζες μια πηγή χρηματοδότησης ε, μακροπρόθεσμη για να ελοπιθεί ο στόχος αυτός. Τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην αποδυναμώσουμε το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών. Καταρχήν, χωρίς αυτό να ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει βελτίωση της χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις ε, και τους πολίτες. Και δεύτερον, αν αυτό ενέχει κινδύνους που ε, ουσιαστικά διακυβεύουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι αξιοσημείωτο, γιατί θα επιτρέψει στις χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμη αγορές αυτές να ευνοήσουν τη δημιουργία ενός εργαλείου που ε, φαίνεται να είναι σταθερό ακόμη και σε περίοδους κρίση και να φέρθηκε ο συγητή. Άλλα εργαλεία όπως ε, παραδείγματος χάρη ε, μιας ευρωπαϊκής εγγύησης θα συζητηθούν περαιτέρω. Και καθώς τελευταία φορά παίρνω το λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία και θα ήθελα να σας, να σας ευχηθώ. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια η κυρία Μπέρες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το πλαίσιο της ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών καθεστώτων που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πρόσδεκτο. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα χρήσιμο εργαλείο επαναχρηματοδότησης και θα συνεισφέρει στην εμβάθυνση των κεφαλαίων θα πρέπει να θυμηθούμε όμως ε, ότι ε, τα ομόλογα αυτά έχουν επιτρέψει στις τράπεζες λειτουργήσουν σε δύσκολες συνδικές στην αγορά το 2008 παραδείγματος χάρη όταν είχαμε ε, το, το πόγιο της κρίσης. αυτά παίρνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε εθνική αγοράς. Στη Γαλλία υπάρχει δυνατότητα να ε, έχουμε διαφορετικά στοιχεία κάλυψης. Ε, ε χάρη να έχουμε ε, και ε, δάνεια σε κίνητα αλλά και σε άλλες χώρες Δανία, Σουηδία, Ισπανία ε, και γι' αυτό έχουν εμπνευστεί από τις καλύτερες ε, πρακτικές με την δυνατότητα να έχουμε και αυτή την ευρωπαϊκή ετικέτα. Επίσης επιτρέπει στους πρωταγωνιστές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ετικέτα διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο και μπορούν να ευνοηθούν και οι επενδυτές ακόμη και σε περιόδους ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι τράπεζες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανένα το λόγο για το ΚΑΤΣΔΙΑΙ, έτσι λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για τις ε, παρεμβάσεις σας, ε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία για αυτά τα καλυμμένα ομόλογα. Οι επενδυτέ εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ότι αυτά τα χρηματοψηφιακά εργαλεία που αποκαλούνται ευρωπαϊκά καλυμμένα ομόλογα ή premium καλυμμένα ομόλογα, αυτά υπάγονται σε ειδική εποπτεία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση, να είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν οι βασικές διατάξεις. Ε, βεβαίως, εμείς θέλουμε να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε τα καλυμμένα ομόλογα να γίνουν ακόμα πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρο. Ε, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο για άλλη μια φορά στον συνάδελφο κύριο Λούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, αγαπητοί στάλφοι. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδης ηγητές, κυρίως και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα ήδη ελέγχθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δύο μόνο παρατηρήσεις θα κάνω. Το πρώτο είναι ένα σύντομο σχόλιο ε, απευθυνόμενος προς τον κύριο Μαριά στον συνάδελφό μου. Βεβαίω και πρέπει κανεί πάντα να εξασφαλίζει ότι τα ομόλογα θα πληρώνονται πίσω. Παράδειγμα, τα κρατικά ελληνικά ομόλογα, παράδειγμα που μερικά δεν αποπληρώνονται. Εδώ όμω μιλάμε για άλλο πράγμα, μιλάμε για ομόλογα τραπεζών. Άρα δηλαδή υπάρχουν εξασφαλίσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πουλ κάλυψης ε, το οποίο είναι προστατευμένο από παρεμβάσεις άλλων ομολογιούχων. Εγώ θα πρότεινα η ελληνική κυβέρνηση στο μέλλον να καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία και τα κρατικά της ομόλογα να τα εξασφαλίζει μέσα από πραγματικές αξίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα έτσι ώστε να βελτιωθεί και η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την δυνατότητα δανειοληψίας. Μετά, αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, σχετικά ότι δεν είναι καλό να διαταράσει κανείς τις εύρυθμα λειτουργούσες αγορές. Ε, σωστό αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, γιατί αν δεν θέλει κανείς να διαταράξει καμία αγορά, ε, τότε θα πρέπει να επιτρέπει όλες τις πρακτικές και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει και τις χειρότερες πρακτικές. Αυτό όμως δεν είναι ο στόχος της εναρμόνισης που επιδιώξαμε. Νομίζω τα καταφέραμε καλά να αποφύγουμε αυτόν, τον παραπλανητικό δρόμο. Με πώς με το να προβάλλουμε την ποιότητα της νομοθεσίας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και με τον τρόπο αυτό ασκούμε πίεση σε άλλα κράτη-μέλη να θελήσουν να προσαρμοστούν. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται γενικά η νομοθεσία για τα καλυμμένα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό ανοίγουμε ένα πολύ καλό δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πέντε λεπτά παρακαλώ στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να αρχίσω λέγοντα ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για προφορική ερώτηση τώρα στο τέλο τη θητείας, αλλά για ένα παράπονο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώ προ την Επιτροπή και το Συμβούλιο, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει θεμητή συνεργασία, ότι δεν υπάρχει θεσμική συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σοβαρό. Πρώτα απ' όλα θέλω να επενθυμίσω τα γεγονότα. Ήδη το άρθρο 226 της συνθήκης της Λισαβόνας επέτρεψε ήδη από το 2009 όταν εγκρίθηκε η συνθήκη αυτή, επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νομοθετική πρωτοβουλία για να ρυθμίζει τις εξουσίες των ερευνητικών επιτροπών. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου σε δύο θέματα, στον εκλογικό ευρωπαϊκό νόμο και στην ρύθμιση ακριβώς των ε, επιτροπών εξέτασης πραγμάτων. Το 2012, τρία χρόνια μετά, από τον David Μάρτεν που ήταν τότε εισηγητή, αρχίσαν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ήδη από την προηγούμενη θητεία δεν υπήρξε συμφωνία και το 2014 σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε το κείμενο αυτό. Εντάξει, χωρί συμφωνία τη Επιτροπή και του Συμβουλίου. Όταν εγώ ορίστηκα εισηγητή στην αρχή αυτή τη θητεία, το 2015, άρχισα να προσπαθώ να κάνω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για πάνω σε ένα κείμενο το οποίο είχε εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα. Και εδώ είναι που αρχίζει το πολιτικό μου παράπονο, γιατί δεν καταφέραμε να πετύχουμε το Συμβούλιο και η Επιτροπή να συνεδριάσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα θεσμικό τριμερή διάλογο, σε έναν λογικό πολιτικό διάλογο, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο να μα επιτρέπει έναν κανονισμό που να ρυθμίζει τι αρμοδιότητε του σώματο σε θέματα εξέταση των πραγμάτων. Πολλές ε, προσπάθειες κάναμε εμείς με ευελιξία που επιδείξαμε προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είπαμε, ετοιμάς, μας είπατε μάλλον ότι είμαστε νέο κείμενο και το κάναμε μετά από εννέα μήνες συνεδριάσεων με τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελικά καταλήξαμε σε ένα νέο κείμενο που το ονομάσαμε non-paper. Το παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο και μας απάντησε με επιστολή, όπως κάνει συνήθως, με ενστάσεις νομικές, ε, αντιρρήσεις, ανησυχίες. Επί της ουσίας η απάντηση ήταν πάντα επί της διαδικασίας. Κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Μία αποδοχή της διαπραγμάτευσης. Και εξού το παράπονό μας ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν συνεργάστηκαν μαζί μας, δεν θέλησαν να έχουν διάλογο μαζί μας. Και μας ε, ταπεινώσατε κυρίες και κύριοι. Έτσι αισθάνομαι, ειλικρινά και μεγάλη απογοήτευση έχοντας δουλέψει τέσσερα χρόνια με την Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, με την κυρία Χούμπνερ, για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση που δεν κατέστη εφικτή. Δεν είναι μόνο διαδικαστικό το ζήτημα, κυρίε και κύριοι. Γι' αυτό και έρχεται εδώ το πολιτικό μας παράπονο. Γιατί το πρόβλημα ουσίας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν δέχονται να υπάρχουν επιτροπές με δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων. Όλες αυτές οι εξεταστικές επιτροπές ενοχλούν τους επιτρόπους, ε, τις κυβερνήσεις κλπ. κλπ, κλπ. Επί της ουσίας λοιπόν αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι φοβόσαστε. Μήπως κληθούν μάρτυρες, επίτροποι, ε, μέλη κυβερνήσεων. Και αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα. Δεν θέλετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει μια εξουσία που είναι τόσο σοβαρή όσο είναι οι εξεταστικές επιτροπές, που είναι κάτι απαραίτητο στον κοινοβουλευτισμό του 21ου αιώνα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αρνείστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια δυνατότητα που του έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας και στον 21ο αιώνα που υπάρχουν τόσα θέματα κακοδίκησης ή που πλήττουν το κράτος δικαίου να μην μπορεί να τα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπούμε απευθείας τους πολίτες για να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν αύριο θα εγκρίνουμε κυρίες και κύριοι ένα ψήφισμα που είναι σκληρό αλλά και δίκαιο. Είναι ένα ψήφισμα ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά είναι κάτι αναγκαίο κυρίε και κύριοι. Αυτά θέλω να σα πω. Θα μεταφέρουμε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και θα του ζητήσουμε στη συνεδρία του με το Συμβούλιο να το πει. Θα το στείλουμε στου πίτσεν καντιντάτε από τι διάφορε πολιτικέ οικογένειε να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πολιτικό παράπονο. Και να συζητηθεί αυτό το θέμα και με τους επόμενους. Είναι αναγκαίο προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ένα κοινοβούλιο που να εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Τεχματικών Επιθέσεων, η κυρία Χουμπνερ, το ε, κύριο όπλο είναι αυτό για ένα σύγχρονο κοινοβούλιο. Αν ε, σκεφτούμε το Dieselgate, το Panama Papers και άλλα σκάνδαλα, κατανοούμε ότι είναι θεμελιώδες ε, το Κοινοβούλιο να έχει δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων εύρωστο. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συστηματικά αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι για να κάνουν πραγματική συζήτηση για το περιεχόμενο τη πρόταση του Κοινοβουλίου. Το επιχείρημα ήταν ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου δεν λάμβανε υπόψη τι θεμελιώδει ανησυχίε. Όμω αυτό σημαίνει ότι αγνοείται την ε, ε, ειδική νομοθετική διαδικασία που έχει θεσπιστεί με το άρθρο 226 της ε, συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση συμβιβασμού αποδεκτή από όλους. Το Συμβούλιο ζήτησε το αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει ήδη να συμπεριλαμβάνει ένα κείμενο αποδεκτό από το Συμβούλιο. Όμως δεν λειτουργεί έτσι η διαδικασία. Πώς το Συμβούλιο η Κομισιόν θα αντιδρούσαν αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνείται ακόμη και να συζητήσει πιθανούς τρόπους επιτεύξης συμφωνίας παραδείγματο χάρη στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντα την πρόφαση ότι δεν του αρέσει η πρόταση τη Κομισιόν. Επιπρόσθετα, η στάση αυτή δεν είναι συμβατή με την αρχή τη ειλικρινού συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων που όλοι πρέπει να σεβόμαστε. Εδώ διακυβεύεται ένα θεμελιώδες θέμα σεβασμού για τα προνόμια του Κοινοβουλίου και για την θεσμική ισορροπία. Πρέπει το Συμβούλιο και η Κομισιό να το κατανοήσουν και τελικά δεν έχουμε υποχρέωση να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, αλλά έχουμε το καθήκον να προσπαθήσουμε. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν αντεπεξέλθει στο καθήκον αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Τσιάμπα εξ ονόματος του Συμβουλίου. Αγαπητέ Πρόεδρε, πλησιά στο τέλος της θητείας και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε το σημαντικό θέμα της άσκησης ε, του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Καταρχάς να σας πω ότι συμφωνούμε ως ε, Συμβούλιο ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί το πολιτικό έλεγχο στην Ένωση και αυτό κατοχυρώνεται στο σεβασμό της ε, αρχής της δημοκρατίας ε, του κράτους δικαίου όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Μετά την έκθεση του 2011 εξετάσαμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου διάφορες προτάσεις με πολύ επικοδομητικό ε, πνεύμα και πάντοτε με την ειλικρινή συνεργασία ως βάση. Είναι γνωστό όμως ότι σε αυτή την έκθεση, ε, την έκθεση Μαρτή υπάρχουν σοβαρές θεσμικές επιφυλάξεις ε, και από πλάσκο και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το 226 το άρθρο αυτό της συνθήκης ε, και σε ό,τι αφορά την επέκταση των εξουσιών και δικαιωμάτων ε, των, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρείται ότι αντιβαίνει στο άρθρο 226 παρά τις προτάσεις συμφιλίωσης διαφόρων επιλογών ζητημάτων Παραδείγματο χάρη, οι εμπειρογνώμονε των νομικών υπηρεσιών προσπάθησαν και με πολλέ συναντήσει έχουμε κάνει πρόοδο σε κάποιε μη προβληματικέ διατάξεις, αλλά δεν έχουμε λύσει τα πιο πολύπλοκα ζητήματα νομικού και πολιτικού χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται σε επιστολή που απεστάλλει στην ε, κυρία Χούπνερ πέρυσι τον Οκτώβριο 25 του μήνα συγκεκριμένα από την Προεδρία του Συμβουλίου, καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεσης ε, κυρίου Χαουρέγκη Ορτουόντο ε, για την αναζωγόνηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Είναι ένα non-paper αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένε βελτιώσει σε σχέση με τι προτάσει του 2014 και ορισμένε από τι ανησυχίε του Συμβουλίου διασκεδάζονται και γίνονται κάποιες προτάσεις ε, όπως πρότειναν νομική υπερογνώμηση των τριών θεσμικών οργάνων. Όμως αυτό ήταν επίσημα έγγραφο εξακολουθεί να περιλαμβάνει κάποιε διατάξει. που θα ε, γύρουν σημαντικά πολιτικά και θεσμικά ζητήματα. Το έχουμε πει και ξαναπεί και κατά το παρελθόν. Επί της ουσίας η θέση μας για τα θεμελιώδη ζητήματα δεν έχει αλλάξει μετά την 6 η Μάρτη και για να είμαι πιο συγκεκριμένος θα ήθελα μεταξύ των πλέον προβληματικών ζητημάτων να αναφέρω ότι γίνεται με κάποιου που καλούνται ως μάρτες και δεν είναι ε, υπάλληλοι, ε, οι αξιωματούχοι. Κροάσεις τέτοιων μαρτύρων η εξουσία να ζητηθούν έγγραφα από πρόσωπα που δεν έχουν ρόλο στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου επιβολή σε περίπτωση μη συμμόρφωση. Και τέλο, η διατάξη για τι κυρώσει είναι κάποια θέματα που μας απασχολούν στο ποινικό δίκαιο. Είναι θέματα που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως και ε, στο πλαίσιο του κώδικα ποινική δικονομίας. Δεν θα έλθω, επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι γνωρίζετε πολύ καλά τις ανησυχίες του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται άλλωστε λεπτομέρειες και στην επιστολή που προανέφερα από την αρχή της Προεδρίας μας προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις ε, ε, και σε επίπεδο κομισιών είχαμε πολλές άτυπες επαφές ε, και οι ε, προκάτοχοι μου ε, συνάντησαν τον κύριο Χαουρέγγι και την κυρία Χούμπνερ και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε να είμαστε ανοιχτοί ε, προ οικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να, να στήσουμε ε, μια διέξοδο ε, σε σχέση με το πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει το έργο με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, είμαστε και εμεί έτοιμοι να το κάνουμε με πλήρη σεβασμό στην αρχή τη ειλικρινού συνεργασία. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Να παρακαλέσω την Επίτροπο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτές, ε, Χαίρομαι που με την προφορική ερώτηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα ε, από πλευρά της Κομισιόν να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά το Κοινοβούλιο διατυπώνει πρόταση, αλλά με τη διαδικασία απαιτείται συγκατάθεση Συμβουλίου και Κομισιών. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε συγκεκριμένε προτάσει για μια τέτοια ρύθμιση, ένα τέτοιο κανονισμό και ανεπίσημα είχαμε αυτό το non-paper τελευταία, το οποίο δίθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πέρυσι τον Απρίλιο και διαβιβάστηκε σε Συμβούλιο και Κομισιόν πέρυσι τον Μάιο. Αναγνωρίζουμε πως η μια ανεπίσημη πρόταση ε, έχει καταρτιστεί ε, με πιο συγκεκριμένους όρους και περιλαμβάνει αρκετές βελτιώσεις. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τη συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής, οι διαδικαστικοί κανόνες που έχουν να κάνουν με την έρευνα ή τη δημιουργία ενό κεντρικού ε, συνδέσμου. Είναι θετικέ εξελίξει. Ναι, η επίσημη πρόταση επίση περιλαμβάνει αναφορά ε, σε έναν κανονισμό για την ε, προστασία φυσικών προσώπων, ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και λαμβάνει υπόψη και τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό το ανεπίσημο έγγραφο εξακολουθεί να δημιουργεί κάποιες νομικές και θεσμικέ ανησυχίε, που ήταν και στο επίκεντρο των συζητήσεων ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου από το 2012 και οι πιο βασικές από αυτές τι ανησυχίε είναι οι κυρώσει για τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού ορισμένε πτυχές ε, των ε, εξαστικών μέσων και εργαλείων που θα έχουν στη θέση του αυτέ οι επιτροπέ, επιτόπιε, έρευνε, ακρόαση με επιτρόπους, νυν και με ακρόαση υπαλλήλου νυν και και τα φυσικά πρόσωπα που είπαμε. Επίσης, ε, μισάγεται ένα νέο κανόνα για τα 11 μέσα σε περίπτωση παραβίαση των διατάξεων της συνθήκης από μια εξεταστική επιτροπή, από τα μέλη τη από παλίλου, εξωματούχους ή άλλες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλος υπάρχουν κάποιες διατάξεις που από ό,τι φαίνεται δίνουν διακριτική ευχέρεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την αναστολή των διαδικασιών τη εξεταστική επιτροπή ε, ε, όταν είναι στο δικαστήριο η άλλε υπηρεσίε του ευρωπαικου κοινοβουλιου και τέλο, υπαρχουν κάποιε διατάξει που απο οτι φαινεται δινουν διακριτικη ευχερεια στο ευρωπαικο κοινοβουλιο σε οτι αφορα την αναστολη των διαδικασιων τη εξεταστικη επιτροπης οταν ειναι στο δικαστηριο η διαδικασια παρα ε, και με επιφύλαξη αυτέ τις ανησυχίες θέλω να πω ότι εμεί είμαστε διατεθειμένοι ω Κομισιόν να συνεχίσουμε οικοδομητικέ τριμερίε διμερείς συζητήσεις ε, με στόχο την εξέβρεση των κατάλληλων λύσεων ε, σε ό,τι αφορά τι αποκλήσει που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Μελλοντικό ε, κανονισμό σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκέ εργαλείο που θα σέβεται και τα θεσμικά προνόμια αλλά και των νομικά πλαίσια των κρατών μελών. Αυτό είναι ο στόχο μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε, ο κύριος Βίλαν δεν είναι στην αίθουσα που θα έπρεπε να λάβει το λόγο. Ως εκ τούτου, εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων, η κυρία Γουαρακουτού. Α, η κυρία Ρουΐς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν μας ακούσατε, κυρία Τσιάμπα. Σας είπαμε. Πολάκης. Καθ' όλα αυτά τα έτη και το είπε και ο κύριος Χαουρέγγι, ότι μιλάμε για έλλειψη συνεργασίας. Δεν υπήρξε πιστή συνεργασία. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Σε αυτό το κοινοβούλιο μας έλειπαν ε, ικανότητες κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας για να μπορέσουμε να εργαστούμε καλύτερα στην περίπτωση των Panama Papers και στο Diesel Day και στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία γιατί εσείς θελήσατε να μπλοκάρετε αυτή τη δυνατότητα. Αν ο κύριος Χαουρέγγι έχει στο DNA του τη διαπραγματευτική ικανότητα και μπορεί πολύ εύκολα να φτάνει συμφωνίες και δεν μπόρεσε να το κάνει είναι επειδή δεν υπήρξε συνεργασία από εσά. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους λοιπόν. Εδώ και 25 χρόνια λειτουργούμε με μια απόφαση η οποία είναι μικρή και παροχημένη. Αυτό δεν είναι το Κοινοβούλιο του 1995. Χρειαζόμαστε αυτά τα προνόμια τα οποία εσείς ε, φέροντας διάφορα επιχειρήματα και διάφορους λόγους δεν θέλετε να δώσετε σε αυτό το κοινοβούλιο και κάνετε λάθος γιατί χάνουμε αξιοπιστία γιατί πρέπει να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα εξέτασης πραγμάτων δεν είναι δίκαιο, δεν είναι αξιοπρεπές αδελφά θεσμικά όργανα, όπως είναι το Συμβούλιο και η Κομισιό, να δένουν τα χέρια του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Όταν ε, ασκούμε τα καθήκοντα που μας ε, έχουν δοθεί. Εμείς αυτό το καθήκον έχουμε να υλοποιήσουμε. Δεν είναι δίκαιο ο κύριος Χαουρέγγι να έχει εργαστεί για πέντε χρόνια όπως το έκανε και η πρόεδρος της ε, Κομισιόν τη Επιτροπή Συγγνώμη Συνταγματικών Επιθέσεων, η κυρία Ντανίτα Κνούμπλερ και η γραμματεία τη ΑΦΚΟ. Δεν είναι δίκαιο. Μα κλείσατε την πόρτα στα μούτρα. Έτσι λοιπόν, το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι δεν ε, υπήρξε ε, ιδέους επιμέλεια από την πλευρά σας. Και ευχαριστώ τον κύριο Χαουρέγγι και πάλι ε, για όλο του το έργο του. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα δεν βλέπω τον κύριο Σόλτς, ο οποίος ε, θα έπρεπε να πάρει το λόγο εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Έτσι λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία James εξ του EFDD. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, χρειαζόταν απόδειξη ότι ε, τελικά ε, αποτελεί ένα προπέτυσμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημοκρατία. Το έχουμε εδώ. Αν πρέπει να έχει νόημα η δημοκρατία, τότε οι νόμιμα επλεγμένοι, οι βουλευτέ εδώ, θα πρέπει να επιτρέπεται να αμφισβητούν οτιδήποτε. Ε, αφορά αυτούς που εκπροσωπούν. τα δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων ε, θα έπρεπε να έχει νομική υπόσταση. Διαφορετικά ποιο είναι το νόημα. Δείχνεται ότι απλώς μια μαριονέτα είναι το Κοινοβούλιο ε, για όσους στην Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν έχουν εκλεγεί. Αυτή ε, η νομική υπόσταση, αν δεν αναγνωριστεί, αυτό υπονοείται και με ενοχλεί που το Συμβούλιο και η Κομισιόν λειτουργούν με έναν τρόπο παρακόλλησης όταν μιλάμε για τη διαφάνεια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, αναρωτιέται η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι λαϊκιστέ και οι ευρωσκεπτικιστέ ανθίζουν και ευημερούν. Έχετε την απάντηση ενώπιον σα. Μιλάμε για ε, ένα μεγάλο πλήγμα στη δημοκρατική διαδικασία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ποσπισίλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λυπούμε πολύ με τη θέση του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Διότι με το πρωτογενές δίκαιο έχουμε σαφές, ξεκάθαρο δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων. Και αν αυτό ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί μέσω εκτελεστικού κανονισμού, πραγματικά είναι ντροπή. Με εντυπωσιάζουν δε περισσότερο, θα έλεγα, ε, τα όσα είπε το Συμβούλιο, η συμπεριφορά του Συμβουλίου. Ε, δεν μπορώ να την κατανοήσω. Θα περίμενα από εκπρόσωπο ενός δημοκρατικού κράτους μέλους να κάνει περισσότερα για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε άμεση εκλεγμένοι πρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εξουσίε τι οποίες μας εκχωρεί το βασικό δίκαιο, το πρωτογενέ δίκαιο και δυστυχώ Συμβούλιο και Κομισιόν μειώνουν τι δυνατότητε που έχουμε και την εξουσία μα. Αν αυτό συνέβαινε κάπου αλλού θα το καταλάβαινα, γιατί πολλές φορές ασκούμε κριτική σε τρίτες χώρες και στον τρόπο με τον οποίο παραβιάζεται το δίκαιο όμως εδώ έχουμε ήδη στη δική μας την πίσω αυλή το ίδιο πρόβλημα. Παρακαλώ λοιπόν σκεφτείτε το, προσπαθήστε τουλάχιστον, διότι πρόκειται για ε, κάτι που πραγματικά μας δυσφημεί. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ στη διαδικασία προσέλκυσης ε, της αποσύγησης του κ. Μαριάς ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός κοινοβουλίου η νομοθετική λειτουργία ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και οι εξεταστικές επιτροπές. αυτά κάνουν τα δημοκρατικά κοινοβούλια και το δικαίωμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να προχωρεί στην εξέταση πραγμάτων δηλαδή να κάνει εξεταστική επιτροπή προβλέπεται αυτοτελώς από το πρωτογενές δίκαιο επομένως πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξασκεί αυτά τα καθήκοντά του διότι όταν δεν προχωρά σε εξεταστικές επιτροπές όταν έχουμε σκάνδαλα όπως τα luxleaks τα panama papers το diesel σκάνδαλο και δεν κάνει τίποτε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τότε μειώνεται η αξιοπιστία του δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις του με τους πολίτες αυτό το δικαίωμα θέλουμε να εξασκούμε αυτοτελώς αυτό διεκδικούμε και νομίζω ότι η τοποθέτηση του συμβουλίου δεν συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ήρθε ο κύριο Σόλτ, άρα μπορώ να του δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό εκ μέρου Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να σα πω ότι εγώ είμαι υπέρ ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πλέον, διότι από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μα δικαστικώ. Κατά την άποψή μου, είμαστε και υποχρεωμένοι ω προ αυτό, διότι είμαστε το Κοινοβούλιο των Ευρωπαίων Πολιτών, των Ποτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το δικαίωμα ε, αυτό είναι δικό του. Να έχουν δηλαδή ένα ισχυρό κοινοβούλιο που οι προνομίε του να γίνονται ε, σεβαστέ. Ε, υπάρχει παρελκυστική πολιτική από το Συμβούλιο και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι που ασκούν επιρροή στα μεγάλα πολιτικά κόμματα και οι οποίοι φοβούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δηλαδή καλεί κάποιους, ε, κάποιο μέλη κυβερνήσεων των κρατών μελών ή συγκεκριμένους ε, ε, μάρτυρες. Ε, τι πρόβλημα υπάρχει. Ε, δεν θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες αυτών των εξεταστικών επιτροπών. Και τι γίνεται αν δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ο θεματοφύλακας τελικά των συνθήκων. Είναι στην ίδια πλευρά με το Συμβούλιο. Και δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ε, πώς το ακούν αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή ε, οι επιτροπές, παραδείγματος χάρη εξεταστικές του Κοινοβουλίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους ε, τα έγγραφα τα οποία ζητούν. Τι έχετε να κρύψετε, τι θα σκεφτεί ο κόσμος ε, όταν ακούσει δεν είναι περίεργο να μην έχετε την ευθύνη να δώσετε κατάθεση ε, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπος κυρία Μπιενκόφσκα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τα αξιότιμα μέλη για τις παρατηρήσεις που έκαναν. Θα ήθελα να επαναλάβω το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο που δραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο. Απότερο στόχος είναι τα συμφέροντα και ανησυχίε των πολιτών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου να αντιμετωπίζονται σωστά, να διασφαλίζεται αυτό. Αναγνωρίζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο που έχουν κάνει τα θεσμικά όργανα και αναγνωρίζει ότι το ανεπίσημο έγγραφο αντιστοιχεί σε σαφή πρόοδο σε σχέση με προηγούμενε προτάσει. Από την άλλη, όμω, όπω είπα και νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ανεπίσημη αυτή πρόταση έχει ακόμα κάποια θεσμικά και νομικά κενά, όπω για παράδειγμα οι κυρώσει, τα ε, ένδικα μέσα τα οποία προβλέπονται και το καθεξής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο εργαλείο το οποίο να τηρεί τα βασικά θεσμικά προνόμια των κρατών μελών αλλά και των θεσμικών οργάνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν ε, οι κατάλληλε τριμερεί διαπραγματεύσει προκειμένου να διασκεδαστούν οι ανησυχίε οι οποίοι ακόμα υφίστανται. Ελπίζω ότι στο πολιτικά αυτό αλλά σημαντικό θέμα θα σημειωθεί, ελπίζω θα σημειωθεί πρόοδο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Τσάμπα, ο υπουργό. Παρακαλώ conclude, Κατακλείδη. Να ευχαριστήσω όλους για την ανταλλαγή απόψεων. Ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις μας, εκατέρωθεν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι προηγούμενες προεδρίες έδειξαν ανοιχτό πνεύμα εν ώψη της προσπάθειας εξέβρεσης λύσης. Συζήτησαμε το θέμα σε βάθος στην αρμόδια ομάδα εργασίας. Δυστυχώς, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να κλείσει ο φάκελος στη διάρκεια της παρούσης θητείας του Κοινοβουλίου. Για άλλη μια φορά όμως, το Συμβουλίο σας διαβεβαιώ ενταγμένο στην προσπάθεια συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά τον Μάιο. Είναι προς το συμφέρον όλων, να θεσπίσουμε ενημερωμένους κανόνες, να επερμηθούμε του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εξαίρεση των πραγμάτων. Ευχαριστώ λοιπόν τον κ. Ντόντοφ για τη σπουδαία δουλειά που έκανε ο συγητής. Ξέρω ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βελτιώσει την τελευταία έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για άλλη μια φορά. Είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται η Προεδρία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που είχαμε τους τρεις τελευταίους μήνες. Είχαμε ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για εμάς ήταν ε, χαρά να συνεργαστούμε με την Ρουμανική Προεδρία, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρος συνεχίζει, έλαβα σχέδιο ψηφίσματος στο τέλος της συζήτησης. Το υποβάλλει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια αύριο. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a to jest sprawozdanie pana Fernandesa i pana Guiteliego. Program... Επόμενο σημείο, Φερνάντε Κολθιέρη, έκθεση σχετικά με την πρώτη κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη θέσπιση του προγράμματο InvestEU. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φερνάντε. Κύριε Πρόεδρε, χαιρετώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ όλες και όλους που εργάστηκαν επί του θέματος που αφορά την περίοδο 21-27. Ευχαριστώ και τον ε, Ρομπέρτο Γαλτιέρη, ο οποίο ε, και αυτό εργάστηκε σκληρά. Και να ευχαριστήσω επίση θερμά τους συναδέλφου που εργάστηκαν σκληρά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το σχέδιο Juncker, το ΜΙΟ Juncker. Ευχαριστώ τους και και τους εργάτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και την Γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Την περιοδο 2027 έχουμε μπροστά μας έναν μηχανισμό ο οποίος ε, συγκεράζει και απλουστεύει τη λειτουργία 14 χρηματοδοτικών μηχανισμών. Ενοποιούνται και απλουστεύονται. Χρειάζεται όμω ε, για να γίνει κάτι τέτοιο ένα φιλόδοξο όραμα. Όπως είπα έχουμε σύμπηξη 14 διαφορετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και όλα αυτά με τη μορφή εγγύσεων 40,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιήσουν συνολικά περίπου 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια μικρή διαφορά τα 650 που θέλει το Συμβούλιο. Ε, εν πάση περιπτώσει έχουμε συμφωνήσει όλα με την εξαίρεση αυτού Χαίρομαι, εν πάση περιπτώσει, για αυτήν την προσωρινή συμφωνία. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σύντομα. Πρόκειται λοιπόν για το νέο ταμείο InvestEU, εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε τέσσερις θηρίδες, κατά κάποιο τρόπο, επενδύσεις σε αηφοροανάπτυξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τρίτον έρευνα και καινοτομία και τέταρτον, τέταρτος άξονας, κοινωνική στόχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εξομαλύνει τις διαφορές σε επενδύσει μεταξύ περιφερειών. Πρέπει οι διακρίσεις, οι διαφορές να εξελιχθούν και όλοι να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα τα κρατημέλη πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ένα νέο πεδίο διότι τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και αυτά στις χρηματοδοτήσεις εθελοντικά μπορούν να βοηθήσουν για παράδειγμα επενδυτικές τράπεζες σε κάποιο άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που παρατηρούνται αδυναμίες. Η κάθε χώρα λοιπόν πρέπει να κάνει αυτό που της αναλογεί. Πρέπει επίση οι διάφοροι οργανισμοί χρηματοδότηση αναπτυξιακή μορφή να προετοιμαστούν. Εμεί βλέπουμε το θέμα θετικά. Θέλουμε να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε θέσει εργασία ποιοτικέ. Θέλουμε καλύτερη διακυβέρνηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών. Και πέραν αυτού όσον αφορά το συμβουλευτικό όργανο στην Πορτογαλία κάνει ό,τι μπορεί σε συνεργασία με την ΕΟΚΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εν τέλει θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών, μια Ευρώπη των περιφερειών. Χαίρομαι που κατορθώσαμε να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση όσον αφορά την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Μάλιστα, καταφέραμε να καταργήσουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αυτού του μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μπορούμε να φτάσουμε σε εγγύσεις έως και 100% σε σύγκριση με το 75% της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο συνεισηγητής, ο κύριος Γκουαλτιέρη, ο οποίος απουσιάζει όμως. Επομένως, δίνω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Μπιενκόφσχα. Αξιότιμα μέλη, η σημερινή συζήτηση για το πρόγραμμα Invest EU στην τελευταία αυτή ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια βληματική συζήτηση για την υποστήριξη που δίνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των επενδύσεων. Εξ ονόματο λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Η μερική συμφωνία, στην οποία καταλήξατε πολύ γρήγορα με το Συμβούλιο για το InvestEU, θα επιτρέψει την γρήγορη προπαρασκευαστική εργασία. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος αυτού στο πλαίσιο του επερχόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το πρόγραμμα InvestEU πρόκειται να απλουστεύσει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και με μια ενιαία εγγύηση, με ένα ε, ενιαίο σύνολο κανόνων θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να καλύψουμε επενδυτικά κενά και να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον θέσεις απασχόλησης, ενεργειακή απόδοση, αστικές μεταφορές είναι ορισμένοι από τους τομείς ε, για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις. Η εγγύηση για το πρόγραμμα Invested Youth θα επιτρέψει τις επενδύσεις αυτές και θα κινητοποιήσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για το δημόσιο καλό. Το Ταμείο αυτό θα υποστηριχθεί από το συμβουλευτικό όργανο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμώ επίση το γεγονό ότι οι συνομοθέτε υποστήριξαν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρχει μια εγγύηση από τον ενωσιακό προπολογισμό. Ο στρατηγικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πλέον έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο του κανονισμού και να γνωρίζετε καλύτερα η εμπειρογνωμοσύνη τη τράπεζα αυτή, αλλά υπάρχουν πλέον και άλλοι παράγοντε όπω διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπω η EBRD, η Τράπεζα του Συμβουλίου τη Ευρώπη, οι Εθνικέ Επενδυτικέ Προθετικέ Τράπεζε και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν εταίροι υλοποίηση. Κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε όλη τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη με έναν τρόπο συμπληρωματικό, συνδυαστικό, προκειμένου να έχουμε καλύτερη γεωγραφική κάλυψη και να λάβουμε υπόψη τι τοπικέ ιδιαιτερότητε. Η προετοιμασία του προγράμματος αυτού αλλά και η εφαρμογή του θα φέρει κοντά τους παράγοντες αυτούς, θα τους ε, δώσει τη δυνατότητα να έχουν την κυριότητα του συστήματος αυτού και να διαμορφώσουν το μελλοντικό πρόγραμμα Invest in You. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μακροπρόθεσμου ισχυρού επενδυτέ, οι οποίοι θα υποστηρίζουν του βασικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο, προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη πολιτική καθοδήγηση στο πρόγραμμα InvestEU, η απαραίτητη λογοδεσία, η απαραίτητη διαφάνεια και προκειμένου να αυξηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα αυτά τα σημεία βελτιώνουν την νομοθετική πρόταση. Πρέπει να πω ότι ε, εκτιμούμε πάρα πολύ τις σημαντικότερες προσπάθειες που κατέβαλαν οι δύο συνεισηγητέ, οι σκιώδει εισηγητέ και οι δύο εμπλεκόμενες επιτροπές προκειμένου να καταφέρουμε πάρα πολύ γρήγορα σε ένα πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Δράτω με τι ευκαιρίε προκειμένου να ευχαριστήσω και τη Ρουμανική Προεδρία για τι προσπάθειε που κατέβαλα και αυτή. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιφερειακής ε, ανάπτυξη που είναι η κυρία Τζεντίλε. Αλλά από ό,τι βλέπω, έρχεται ο συνεισηγητή. σω θα σα δώσω λοιπόν το λόγο μετά, κυρία Τζεντίλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε δίνουμε τη δυνατότητα στους ε, Ευρωπαίους πολίτες να δούνε ξεκάθαρα ότι αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε, συχνά, περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο από μια πολιτική λιτότητος προς μια πολιτική επενδύσεων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, όλο και περισσότερο στρεφόμαστε προς την βιωσιμότητα, προς την ε, αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω του προγράμματος You μπορούμε να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, μπορούμε να προωθήσουμε φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές ή την κυκλική οικονομία. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε σχολεία, πανεπιστήμια, καταρτήσεις ε, για νέες θέσεις απασχόλησης. Μπορούμε να ενισχύσουμε επίσης τη δημόσια υγεία, την υγειονομική περίθαλψη. Μπορούμε να προωθήσουμε την κοινωνική οικονομία και να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Το πρόγραμμα InvestEU είναι ένα πρόγραμμα υπέρ των πολιτών και λαμβάνει υπόψη πραγματικά την ευημερία και την καλή διαβίωση όλων των πολιτών σε όλες τις πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ένα πρόγραμμα το οποίο βάλει κατά της φτώχειας. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη, το συνεισηγητή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματική χαρά για μένα να μπορώ να παρουσιάζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πόρισμα μιας ε, άοκνης ε, προσπάθειας που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες και που έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου, Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε, καθώς επίσης και όλους τους και και όλου όσοι συνέβαλαν προκειμένου το κείμενο αυτό να βελτιωθεί. Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε η οικονομική κρίση, είχαμε την πολιτική λιτότητος και κατά αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν πάρα πολύ οι δημόσιε αλλά και οι ιδιωτικέ επενδύσει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία πρωταρχική μα λοιπόν προτεραιότητα ήταν να δώσουμε νέα όθηση στι επενδύσει, περισσότερε επενδύσει ω βασική προπόθεση για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Χάρη σε μία ευέλικτη ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητα και χάρη σε νέε πρωτοβουλίε, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων καταφέραμε να διορθώσουμε την ακολουθούμενη πολιτική οικονομίας. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πολλά επενδυτικά κενά όσον αφορά την καινοτομία, όσον αφορά τις υποδομές, υλικέ και άειλε ε, όσον αφορά τι κοινωνικέ πολιτικέ και όσον αφορά την πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Όλε αυτέ οι προκλήσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ και ελπίζουμε θα τι αντιμετωπίσουμε τώρα με το νέο αυτό πρόγραμμα InvestEU. Ενισχύουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στον τομέα τη έρευνα, στον τομέα τη καινοτομία, τις βιώσιμες υποδομές και θεωρούμε ότι με το πρόγραμμα αυτό, το InvestEU, θα καταφέρουμε να καλύψουμε τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις κοινωνικές υποδομές και θα καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε πολλά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής στέγασης. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Συμβούλιο επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, καταφέραμε να θεσπίσουμε ότι το κόστος της εγγύησης για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνδέεται με το προφίλ του κινδύνου των συγκεκριμένων οικονομικών επενδύσεων και ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε επενδυτικές πλατφόρμες και να προωθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις στις περιοχές εκείνης Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα επενδυτικά κενά. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να επέμβουμε μέσω επενδύσεων στι περιοχέ εκείνε οι οποίε υπολείπονται σε σχέση με τι υπόλοιπε πιο προηγμένε περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι δίδεται μέσω τη νέα αυτή πρόταση ένα πιο κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και στι εθνικέ επενδυτικέ τράπεζε, προκειμένου να μπορούν και αυτέ να συμβάλλουν στο υπηρετικό αυτό πρόγραμμα. Οι εθνικέ αυτέ τράπεζε πρόθεση θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην ενωσιακή εγγύηση και κατά αυτόν τον τρόπο του δίδεται μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερε δυνατότητε χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων που μπορούν να έχουν πολύ θετικέ επιπτώσει για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Τέλο, καταφέραμε να θεσπίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν όχι μόνο τη δυνατότητα να δίνουν μέρος των πόρων τους στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και κατ' επέκταση έπειτα στο πρόγραμμα Invest in You, αλλά θα μπορούν να συνεισφέρουν και με επιπρόσθετους πόρους που κατά προτεραιότητα θα θεωρούνται κατά αποκοπήν ε, συνεισφορέ στο πρόγραμμα και επομένως δεν θα συνυπολογίζονται στον ε, υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματο στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το κείμενο λοιπόν το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο κείμενο και απαιτείται αυτή τη στιγμή ένα 55% των επενδύσεων να συμβάλλουν στους στόχους που προβλέπονται στην Συμφωνία των Παρισίων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το απαραίτητο επενδυτικό θετικό κλίμα, να υπάρχει απαραίτητη προβλεψιμότητα όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό InvestEU να συνάδει περισσότερο με τη χρηματοδότηση η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι ισχυρή στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το πρόγραμμα Invest in You είναι ένα πρόγραμμα καθοριστικό, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί την μόνη πολιτική προτεραιότητα για την επόμενη α, κοινοβουλευτική θητεία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σφαιρικό επενδυτικό πρόγραμμα, προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική βιωσιμότητα, την απασχόληση και την καινοτομία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει εκ μέρους του ΕΛΚΑ ο κύριος Κάρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συγητές Φερνάντες Γκουαλτιέρη. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους ε, ε, και να πω ότι και ο τον Μπούλμαν και εγώ ξεκινήσαμε μαζί με σας αυτόν τον αγώνα για τις επενδύσεις. Σίγουρα ε, δεν είναι ένας ε, αγώνας ε, ταχύτητας, αλλά ένας μαραθώνιος. Ξεκινήσαμε με το σχέδιο Juncker αυτό το μαραθώνιο, που ήταν η πρώτη πρωτοβουλία. Έπειτα είχαμε το FC2 που βελτίωσε τα πράγματα και έχει επιμηκυνθεί η ισχύ του μέχρι το 2020. Θέλουμε επίσης να δούμε και τι γίνεται με τις χώρες γειτονία και για την Αφρική. Και κλείνουμε τώρα αυτή την νομοθετική θητεία με ένα επόμενο κεφάλαιο μέχρι το το 2027 το InvestEU 200 ε, δις ε, ε, ευρώ επενδύσεων προωθήθηκαν 954.000 επιχειρήσεις μπορούν να υποστηριχθούν και μέχρι στιγμής έχουμε κινητοποιήσει 50 δις και θα έχουμε και πολύ περισσότερα ε, κέρδη. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Με το InvestEU Έχουμε ε, επίσης ε, έναν πολύ αποτελεσματικό στόχο, τη μείωση της γραφειοκρατίας, συγχωνεύοντας τα 14 αυτά εργαλεία σε ένα. Και επίσης ενισχύουμε και την εφαρμογή των στόχων για το κλίμα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχουμε αυτό το 25% τουλάχιστον ε, των εγγύσεων που θα πρέπει να συνεισφέρουν προς αυτό το στόχο. Επίσης βελτιώνουμε την παροχή συμβουλών, την υποστήριξη και αυτών ε, που συμμετέχουν σε σχέδια, σε έργα μικρής ε, κλίμακας και έχουμε επίσης την εγγύηση αυτή που την επενδύουμε και σε μικρότερα Ινστιτούτα, σε μικρότερα ιδρύματα. Επίσης βελτιώνεται η διαφάνεια των επενδυτικών αποφάσεων. Το InvestEU όμως δεν είναι το τέλος είναι αν θέλετε το τέταρτο ορόσημο, είναι το τέταρτο στάδιο που θα ενισχύσει ε, τις επενδύσεις από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι και στην επόμενη ε, θητεία θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκλοανέκα Μωρά εκ μέρους Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά και εγώ θέλω να χαιρετήσω το έργο των συνεισηγητών. Η μερική προσωρινή αυτή συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU στο πλαίσιο βεβαίως του ΠΔΕΛΤΑΠΗ 2021-2027 είναι ένα ηχηρό θετικό μήνυμα που ε, είναι υπερήφανο που στέλνει προς ε, το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη και του σε επιτυχία του πρώτου επενδυτικού προγράμματο του σχεδίου Juncker για πολλαπλασιασμό των επενδύσεων με δημιουργία θέσεων απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη από τον Ιανουάριο του 2021. Έτσι, η χρηματοδότηση για τοπικά έργα θα προωθηθεί στον τομέα τη έρευνα, των βιώσιμων υποδομών, ψηφιοποίηση, στήριξη ΜΜΕ, κάτι πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως ε, θεσπίζεται και η εγγύηση που βάζει και έναν ηθικό βιώσιμο χαρακτήρα στην επένδυση. Και αυτό είναι σημαντικό. Μιλάμε για σημαντικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ ε, ΤΕΠ, ε, Κομισιών, και εθνικών και τοπικών επενδυτικών τραπεζών για την πρόθεση περιβαλλοντικών κοινωνικών έργων που επιλέγονται ε, για να σεβαστούμε τους στόχους των Παρισίων και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Εθνών. Μία παρατήρηση έχω ε, που αφορά το τέταρτο σκέλος για το οποίο έκανε λόγο ο κύριος Φερνάντες που λέει ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε κοινωνικές ε, επενδύσει. επενδύσεις στις διάφορες αρμοδιότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους κλάδους των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να σχετιστούν με το θεματολόγιο τον πολιτισμό που δεν μπορεί να μείνει εκτός ε, του διαλόγου. Ε, πρέπει επίσης να στραφούμε ε, εμείς στους πολίτες, γιατί η Ευρώπη έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα απλό χρηματοδοτικό εργαλείο. Το InvestEU πρέπει να είναι φαλτήριο προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ακολουθεί αυτές τις αλλαγές και θα οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή ε, παραδείγματος. Θα πρέπει επίσης να είμαστε προοδευτικοί είναι μια Ευρώπη που θέλουμε να δημιουργήσουμε που θα είναι κοντά στους πολίτες, δίνοντας συγκεκριμένες ελπίδες και φιλοδοξία. Πακέτ, Πρόεδρε, ευχαριστώ Ελβέστιγιου. Θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία. Περίπου 40 δισεκατομμύρια με τη μορφή εγγυήσεων, δεν πρόκειται για επιχορηγήσεις. Πολλές επενδύσεις θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σε πολλούς τομείς. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε θα τύχουν υποστήριξης και θα μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα δεν θα εξαρτώνται από εξωευρωπαίους δωρητές. Θα γίνει μια σύμπηξη λοιπόν των εφισταμένων χρηματοδοτικών επενδυτικών μηχανισμών. Αυτό είναι εξαιρετικό. Τα πάντα πλουστεύονται. Οι εθνικές προθερικές τράπεζες αποκτούν σημαίνοντα ρόλο. Οι φρεμαδικές τράπεζες θα έχουν σημαίνοντα ρόλο και στη δική μου χώρα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα λοιπόν είναι έκτακτο, έξοχο. Η αλλαγή αυτή θα φέρει αποτελέσματα. Πρόκειται για την τελευταία μας ολομέλεια βεβαίω και πιστεύω ότι τελειώνουμε πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της ομάδας Άλντε, κυρία Βίρινγκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είχαμε καταρχά το ΕΦΣΙ και τώρα το InvestEU, το οποίο θα δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και στην επόμενη θητεία. Και δείχνει μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Ένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε από την κρίση του 2008 είναι ότι η σταθερή οικονομία συνιστά ε, μια οικονομία των επενδύσεων. 650 σε, σε παραπάνω επενδύσεις λόγω του προγράμματος. Και αυτό είναι μια υπόσχεση για το μέλλον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 Τιέρες για την επίτευξη ικανοποιητικής συμφωνίας όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του πρόγραμματος InvestEU. Όπως είπε και η Επίτροπος, παρέχουμε ένα κίνητρο, ενθάρρυνση στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με το επόμενο κοινοβούλιο. Έχουμε ξαναμιλήσει για το πρόγραμμα αυτό γιατί όντω πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία όμως θα έχει η μελλοντική εφαρμογή στα κρατημέλη. Θα πετύχει όταν γίνει πιο ορατό, όταν κατορθώσει να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εμπορικές τράπεζες ή από το Ταμείο Συνοχής. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, στις νοφείς επιχειρήσεις. Πρέπει να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν σε μέγεθος. Πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι οποίοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας επενδύσουμε λοιπόν σε έργα τα οποία έχουν μια δυναμική, τα οποία όμως δεν εκτιμάει η αγορά. Χρειάζεται επίσης προσοχή στην γεωγραφική κατανομή των πόρων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αφορούσε κυρίως τις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Ήρθε η ώρα όμως να βοηθήσουμε και τις άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Περέση, παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έγκριση του κειμένου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προκρίθηκε με το σχέδιο Juncker και, την, και χάρη πίεση των σοσιαλιστών. Είναι μερική η νίκη μας εν ώψη της περίοδου 21-27 ε, αλλά χαιρόμαστε έστω και γι' αυτό. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, Σίγουρα έχουμε πετύχει μια καλύτερη ισορροπία, διότι υπάρχει μια διευθύνουσα επιτροπή, μια επιτροπή διακυβέρνηση, όπου συμμετέχει και η Κομισιόν και άλλοι θεσμικοί εταίροι, εθνικές αναπτυξιακέ τράπεζες, καθώς και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις κλειδί με οικολογικό επίσης σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγκαλιάσει το θέμα των αϊφορικών υποδομών, των επενδύσεων στην κοινωνία και στις δεξιότητες καθώς και στον τομέα του πολιτισμού. Προσοχή όμως, το θέμα της καλύτερης στοχοθεσίας. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των δεσμευσεών μας πρέπει το 40% των επενδύσεών μας να πάει προς το πρασίνισμα της οικονομίας. Και να θυμηθούμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλη μια φορά της δίνει προεξέχοντα ρόλο. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για καλή απόφαση όσον αφορά ε, τα δικαιώματα που θα έχει στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέτς, παρακαλώ. Πρόεδρε, το Invest e αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά κάποιες ενστάσεις που έχω και στις οποίες θα αναφερθώ στο τέλος. Το θέμα είναι λοιπόν να εγγυηθούμε τον στόχο της αντιμετώπισης της μεταφορής του κλίματος. Το θέμα είναι καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Λήψη υπόψη της ανάγκης προστασίας του κλίματος Τώρα, ως προς τις ενστάσεις μου, βλέπω ότι εντάσσεται το πρόγραμμα μας και η άμυνα, καθώς και άλλα έργα τα οποία δεν έχουν σχέση με την προστασία του κλίματος. Βλέπω αεροδρόμια, βλέπω επενδύσεις στην ενέργεια μέσω των ορυκτών καυσίμων. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον του πλανήτη ή όχι. Όταν έρθει ο Μάιο λοιπόν και η ώρα των εκλογών σκεφτείτε τις ανάγκες του πλανήτη. Πρόεδρος. Ε, ο κύριος Πασπισίλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συναδελφοί μου ε, με κάλυψαν ήδη λέγοντα πολλά σημαντικά πράγματα όσον αφορά το πρόγραμμα Invest in You, το οποίο προφανώ υποστηρίζω. Θεωρώ ότι το παιδιτικό αυτό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Η εμπειρία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει δείξει ότι οι πρωτοβουλίε αυτέ είναι απόλυτα λογικέ, σκόπιμε και ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μέσω επενδύσεων σε τομεί οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται αρκετά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το πρόγραμμα Invest in Youth επικεντρωθεί στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Χαίρομαι πολύ που θα προωθήσει τους στόχους αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, θα προωθήσει τους περιβαλλοντικούς στόχους και την πολιτική έρευνας και κοινοτομίας. Πιστεύω ότι στο μέλλον το πρόγραμμα InvestEU θα προωθήσει εν γέννη την ευρωπαϊκή οικονομία, ακριβώς επειδή έχει έχει, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παρέχει εγγύησεις για ιδιωτικά δάνεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω λοιπόν το διάδοχο πλέον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θεωρώ ότι έχουμε αντλήσει πολύ θετικά διδάγματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021 με 2027. Ευελπιστώ λοιπόν ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό ώστε να αρχίσει να υλοποιείται από το 2020 και μετά. Κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πριν πέντε χρόνια οι σοσιαλιστές ε, όταν κατεβήκαμε στις ευρωεκλογέ απαιτούσαμε το τέλος ε, της λιτότητας ε, των πολιτικών προσαρμογής και ζητούσαμε να δοθεί μεγαλύτερη τόνωση και όθηση στις επενδύσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Φυσικά και ευχαριστούμε και την Κομισιόν και όλες τις πολιτικές ομάδες που προώθησαν το σχέδιο Juncker γιατί αυτό ήταν σημαντικό για να αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια η κρίση. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το βήμα που γίνεται τώρα για τη δημιουργία ενός μόνιμου εργαλείου. Το νέο αυτό, Invest Europe, Invest EU, που θέλει να συνεχίσει να τονώνει τι επενδύσει ε, και να τη στηρίζει μόνιμα στην Ένωση, είναι κάτι πολύ απαραίτητο αυτή τη στιγμή που βιώνουμε μια μεγάλη περίοδο στασιμότητας και τελμάτωσης. Ε, το σχέδιο Γιούνκερ, ε, όμως ε, εξακολουθεί να χρειάζεται αντικυκλική πολιτική, όπως αυτή που μπορεί να προσφέρουν αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές. Το πρόγραμμα InvestEU είναι μία από τις ε, πιο κεντρικές πλέον πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε θέση να κινητοποιήσει εγγυημένες ιδιωτικές επενδύσεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πολύ πιο φιλικό προβλέψιμο κλίμα για τους επενδυτές. Και βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο μέσω των επενδύσεων αυτών συμβάλλουμε στην ε, ευημερία των πολιτών μέσω καλύτερης οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης, μέσω της έρευνας, της καινοτομία, της ψηφιοποίησης και μέσω της υπεύθυνη χρήση των πόρων. Επί του παρόντος, οι επενδύσεις βλέπουμε ότι επικεντρώνονται σε ορισμένα μόνο κράτη-μέλη. Συνεπώς, Μέσω του προγράμματος αυτό InvestEU και μέσω των επιλέξιμων προγραμμάτων θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε την κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία προκειμένου να μην αυξάνονται περισσότερο ανισότητε μεταξύ των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, α μην στο ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνήθω αντιμετωπίζουν πολύπλοκε διαδικασίε όταν, όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν επενδύσει. Έρχεται λοιπόν τώρα το πρόγραμμα Invest in You για να απλουστεύσει τι διαδικασίε αυτέ και να μειώσει τη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να καταφέρουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, ιδίως σε κάποια μικρά τοπικά προγράμματα, ακριβώ εκεί που μπορεί να επιτευχθεί μόχλευση και εκεί πέρα που μπορούν να συμμετέχουν πολλά κλάστερ ε, επενδυτών. Οι δημόσιε όμως αρχές θα πρέπει και πάλι να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει απαραίτητη δανειοδότηση και το απαραίτητο θετικό ε, κλίμα προκειμένου να προσελκυθούν περισσότερες επενδύσεις. Κύριε Ρούμπιχ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κάρας ε, της, ε, του Intergroup για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ο οποίος στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική στρατηγική απόφαση, γιατί θέλουμε να πετύχουμε την ευημερία τους πολίτες και μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ και 25 χρόνια ξέρω πολύ καλά ε, έχουν πετύχει τα ΔΕΛΤΑΠΗ ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 500 δις ε, διατέθηκαν και από το 2007 στο 2013 που προωθήσαμε το πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με 2 δις. Και βέβαια έχουμε και το Micro ΜΜΕ, 3 δις και το εύση με 500 περίπου ε, δις μαζί με τη μόχλευση. Έτσι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουμε ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 25% τώρα ε, προβλέπεται για επενδύσεις στον τομέα του κλίματος. Ε, και βλέπουμε ότι έχει κάνει έτσι μία στροφή προοδευτική η Ευρωπαϊκή Όνωση για να ε, είμαστε πρωταγωνιστές ε, και θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μπιενκόφσκα γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο ε, να στηρίξει κανείς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δείξαμε όμως ότι αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστώ και καλή τύχη. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία προσέλκυση προσοχή ε, του Προέδρου Κάτς Διάη. Μία, ε, ένας μάλλον ιστισόλογο, Κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα InvestEU πράγματι θα μπορούσε να αποδώσει και θα μπορούσε να συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να στηρίξει την κατάρτιση, να στηρίξει τις δεξιότητες αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν με το σχέδιο juncker διότι η εμπειρία από το ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων ιδίως για την ελλάδα απέδειξε ότι τον των χρημάτων τον πήραν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες στην πράξη χρηματοδοτήθηκαν για να αρπάξουν τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. κλασική περίπτωση η fraport η οποία υποτίθεται ότι θα έκανε επενδύσεις στο πλαίσιο μιας δίθεν αποκρατικοποίησης που επέβαλε η τρόικα και έχουμε μια κρατική γερμανική εταιρεία η οποία παίρνει δάνειο 280 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα τόσα από Ελληνική Τράπεζα και αρπάζει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τέτοιου είδους επενδύσεις δεν νομίζω ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Απλά χρηματοδοτούνται οι δίθεν ιδιωτικοποιήσεις άρα λοιπόν το πρόγραμμα πρέπει να πάει σε μια κατεύθυνση στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αυξημένη προστιθέμενη τοπική αξία. ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπιενκόφσκα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί βουλευτέ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, καθώ και για τα θετικά σα ε, σχόλια για το πρόγραμμα. Και το βασικό συμπέρασμα, το οποίο συνάγω από αυτή τη συζήτηση, είναι ότι υπάρχει συντριπτική υποστήριξη ε, υπέρ του προγράμματος InvestEU. Πάντως σημειώνω βέβαια και τις πολύ ψηλές προσδοκίες σας και τις συστάσεις σας ε, για την ε, εφαρμογή αυτού του προγράμματος και θέλω να σας πω ότι θα τις μεταφέρω και θα τις λάβουμε υπόψη αυτές τις συστάσεις ε, κατά την προπαρασκευή του προγράμματος. Ξανά να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές αλλά και όλους όσοι λάβατε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ και για να ολοκληρώσουμε θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή κύριο Φερνάντης. Οι δημόσιες επενδύσεις ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι ιδιωτικές επενδύσεις εξίσου σημαντικές. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, ε, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφύης επιχειρήσεις, να ενισχύσουμε την ε, παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα αμείβονται καλύτερα, με καλύτερους μισθούς, οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες επενδύσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις ε, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Δυστυχώ στη χώρα με την Πορτογαλία. Με το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση και ιδίω ο Πέδρο Μάρκε, ε, ο αρμόδιο υπουργό, δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ ε, για επενδύσει. Το έργο, το σχέδιο Juncker και το InvestEU θα πρέπει να αξιοποιηθούν για δημόσιες επενδύσεις μεταξύ άλλων, όχι μόνο για ιδιωτικέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να βάλουν το λιθαράκι τους. Ε, στο κοινοβούλιο αυτό εγκρίναμε αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για 700 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κινητοποιούνται πάρα πολύ καλή γεωγραφική κατανομή. Έτσι ε, ενισχύουμε και αυτή την πλατφόρμα, αυτό το συμβουλευτικό κόμβο του InvestEU. Πρέπει να υπάρχουν όμως σε εθνικό επίπεδο τέτοιοι κόμβοι που θα βοηθούν τους επενδυτές. Θα μπορούσαν να είναι και περιφερειακές βέβαια οι πλατφόρμες αυτές ε, με στόχο να βοηθήσουμε να διαρθρωθούν τέτοιου είδους επενδυτικές πλατφόρμες και να ε, κατατίθενται καλές υποψηφιότητε για την αξιοποίηση του Ινβεστιγιού. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε περισσότερη ε, σε επενδύσεις, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Θα πετύχει δηλαδή ε, τους στόχους του αυτό το πρόγραμμα του InvestEU. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και στο πέρα τη συζητήσεω θέλω να ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία. Οι ψηφοφορίες θα λάβουν χώρα αύριο. Θα είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση. Ξεκινούμε στις 8 και μισή έως τις 2. Η μέσα διάταξη είναι ήδη δημοσιευμένη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω τον κύριο Ρουμπίχ όμω που θέλει τον λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, των ε, βουλευτών ε, που είναι παρόντες θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί προεδρεύατε υποδεγματικά πάντοτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και ελπίζω και υπό άλλες συνθήκες να ξανασυναντηθούμε κατηδίαν ίσως και να έχουμε και άλλες τέτοιες συζητήσεις στην ωραία σας τη χώρα. Ευχαριστώ και πάλι ο Πρόεδρος και κλείνει η συνεδρίαση εδώ σε αυτό το σημείο.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 διακοπή σας συνεδρίαση, τα χθεσινά πρακτικά και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Παρατηρήσεις, αν δεν υπάρχουν, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και περνούμε στο πρώτο σημείο της απογευματινής μας ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Μετσόλα, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η κυρία Μετσόλα, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανατέθηκε σε μένα η έκθεση αυτή και κανείς δεν φανταζόταν ότι θα καταφέρναμε έξι μήνες μετά την υποβολή της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Χρειάστηκε λοιπόν να καταβάλουμε πολλέ προσπάθειες, χρειάστηκε να αναλύσουμε όλε τι τεχνικέ πτυχέ και λεπτομέρειε τη πρόταση αυτή, χάρη όμω στην ιδιαίτερη επικοδομητική συνεργασία που είχαμε του συναδέλφου εδώ στο Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί ενό νέου συστήματο για το οποίο μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχαμε κατά νου ότι θα πρέπει να είμαστε Δίκαιοι απέναντι σε αυτού οι οποίοι χρειάζονται προστασία, αυστηρή με όσου είναι παράτυποι μετανάστε και ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και απαιτητικοί με όσους εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τώρα τη νέα αυτή νομοθεσία και σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς αρχικά καταφέραμε να επερκεράσουμε όλα τα προβλήματα και καταλήξαμε τελικά σε μια νέα πρόταση για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θεσπίσουμε συγκεκριμένο αριθμό συνοριοφυλάκων προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να μπορούμε να καταπολεμούμε την διεθνή εγκληματικότητα και προκειμένου να μπορούμε να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα όσων χρειάζονται προστασία και προκειμένου να μπορούμε βέβαια να διαχειριζόμαστε και τη μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να έρθουν στο ύψο των ευθυνών του. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο το νέο αυτό σύστημα το οποίο προτείνουμε αυτή τη στιγμή θα είναι αποτελεσματικό. Βέβαια, η νομοθεσία αυτή δεν είναι η μοναδική λύση που χρειαζόμαστε στον τομέα τη μετανάστευση είναι καθοριστική όμω σημασία προκειμένου να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την νομοθεσία αυτή με τι υπόλοιπε νομοθεσίε. Αν αντιμετωπίσουμε ανάλογη κρίση με αυτή που είχαμε το 2015, τότε τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, όπω η Μάλτα ή πολλέ άλλε χώρε, θα μπορούν πλέον να έχουν επιπλέον προσωπικό και θα μπορούν πλέον να έχουν την απαραίτητη συνδρομή την οποία χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτέ τι καταστάσει κρίση. Η νομοθεσία λοιπόν αυτή που έτυχε διαπραγμάτευση στους τελευταίους μήνες δεν αφορά μόνο τα 10.000 αυτά επιπλέον άτομα. Σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιστροφής για όσους είναι παράτυποι μετανάστες. Μα δίδονται με τη νέα αυτή νομοθεσία περισσότερε δυνατότητε να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη, ιδίω όσον αφορά τον εντοπισμό των παράτυπων μεταναστών και μπορούμε επίσης μέσω της νέας αυτής πρότασης κανονισμού να μπορούμε να δώσουμε, να χορηγήσουμε πιο εύκολα συνδρομή προ του νόμου μετανάστε και να του δώσουμε και τα απαραίτητα εξωτικά έγγραφα. Έχουμε νέε αρμοδιότητες πλέον για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μπορεί πλέον ο οργανισμό αυτό να προασπίζει και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων θα πρέπει να προστατεύονται. Απότερο στόχο μα είναι να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία, το οποίο να συνάδει με τι βασικέ ευρωπαϊκέ αξίε, οι οποίε για μα είναι πάρα πολύ σημαντικέ ιδίω για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Και αυτό διότι βέβαια γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη θα πρέπει να προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ο Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στη γλώσσα σας ε, σας ευχαρίστησα. Πώς ήταν η προφορά μου. Θέλει λίγο ακόμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν σας κρύβω ότι τα σύνορα και η ακτοφυλακή είναι ένα βασικό βήμα για μια συνολική πολιτική μετανάστευσης. Δημιουργήσαμε και εγκαταστήσαμε και ενισχύσαμε σε χρόνο ρεκόρ τον οργανισμό αυτών με κοινέ προσπάθειες. Γνωρίζοντας πολύ καλά τη συνθετότητα των νομοθετικών διαδικασιών συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται περί κατορθώματος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια κυρία Μέτσολα και όλους τους σκιώδεις και τη Ρουμανική Προεδρία που ε, κατέληξαν σε ισορροπημένη συμβιβαστική λύση επί της πρότασης. Η συμφωνία υπογραμμίζει πάλι ότι, και πάλι όταν συνεργαζόμεθα έχουμε καλά αποτελέσματα και δείχνουμε στους πολίτες ότι η Ένωση είναι πρόθυμη και ικανή για δράση. Όταν η κρίση κορυφώθηκε στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015, η Ευρώπη ε, κατελήφθη εξαπίνης και δεν ήταν έτοιμη. Αντιμετωπεί με εισρωή παράτυπων ε, εισόδων από Ανατολάς και Νότο, από τη Μεσόγειο, ε, καταλάβαμε ότι έπρεπε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Δεν υπήρχε ε, ενιαίος οργανισμός για τα σύνορα, ούτε υπήρχε, υπήρχαν επιχειρησιακές ικανότητες επιτόπου. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου δεν ήταν κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Τα συστήματά μας πληροφόρησης δεν μιλούν, συνομιλούν μεταξύ τους και οι προσπάθειές μας ε, για να εντάξουμε τρίτες χώρες ήταν κατακαιρματισμένες. Αναγκαστήκαμε να λάβουμε άμεσα μέτρα και μακροπρόθεσμα μέτρα και να εργαστούμε παράλληλα σε όλα αυτά τα μέτωπα. Τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, Όποιος ε, προσπαθήσει να περάσει παράτυπα τα εξωτερικά μας σύνορα εντοπίζεται, ε, λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και εξετάζεται σε βάθος. Σήμερα έχουμε ένα οργανισμό συνοριοφυλακής ακτοφυλακής ολοκληρωμένο, ε, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και συστήματα πληροφόρηση που γίνονται διαλειτουργικά όλο και περισσότερο. Με τον νέο κανονισμό που συζητούμε σήμερα θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Ένα στοιχείο κλειδί είναι το μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων ακτοφυλάκων που θα δημιουργηθεί γρήγορα και θα αναπτύξει την πλήρη επιχειρησιακή ε, δυνατότητα των 10.000 ατόμων μέχρι το 2027. Όμως θα μπορούμε να παρακολουθούμε ήδη την 1η Ιανουαρίου του 2021 ε, την ε, αύξηση του προσωπικού. Το άλλο στοιχείο κλειδί που αλλάζει τα πράγματα είναι ότι το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού θα έχει εκτελεστικές εξουσίες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει διαχείριση συνόρων, καθήκοντα επιστροφών, αυτοδικαίως. Βέβαια, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής θα παραμείνουν υπεύθυνες και θα διοικούν και θα ε, είναι επικεφαλής στις δραστηριότητες των οριοφυλάκων και ακτοφυλάκων που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος τους ενώ θα είναι ε, υπό το κράτος μέλος υποδοχής κάποια, ε, ε, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνεται έλεγχος σε έγγραφα ταυτοτήτων, να υπάρχει άρνηση της εισόδου, να σφραγίζονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να σταματούνται άτομα που παράτυπα επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα και να υπάρχει και ε, υποστήριξη σε διαδικασίες επιστροφών και από άλλες ε, χώρες, από προσωπικό από άλλες χώρες ε, ή για υπηκόους που επιστρέφουν με αναγκαστικά μέτρα. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζονται και θα γίνονται σεβαστά τα ε, υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και θα υπάρχει σωστή ε, κουλτούρα επιχειρήσεων. Ο οργανισμός θα στηρίζει περισσότερο τα κράτη-μέλη στις επιστροφές για να βελτιώνεται η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ε, εμένουσες προκλήσεις μεταναστευτικές. Χαιρετίζω κι άλλες εξελίξεις που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια αυτού του κανονισμού όπως εξυγχρονισμός του παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της επιχειρησιακής δραστηριότητας του οργανισμού. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι στην καρδιά όλων των πρωτοβουλειών της Κομισιόν και αυτής. Όλες οι δραστηριότητες του οργανισμού και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται στο χάρτη. Ο οργανισμός θα συνεργαστεί στενά με τον μελλοντικό οργανισμό ασύλου για να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες του ασύλου. Ο οργανισμός θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε επίσης ότι εκείνοι που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας θα επιστρέφονται με πλήρη σεβασμό τον, επαναλαμβάνω αυτό, πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι όταν θα συγκροτηθεί το επόμενο κοινοβούλιο, η πρόταση σύστασης ε, του, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου θα εγκριθεί σύντομα. Ελπίζω. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι λυπάμαι διότι η δυνατότητα μηνιαίας διαφορικής πληρωμής στο μόνιμο προσωπικό η πρόταση αυτή δεν διατηρήθηκε στην τελική συμφωνία. Αυτό είχε στόχο να βελτιώσει την ελκυστικότητα του οργανισμού ως εργοδότη, να διασφαλίσει επίσης μόνιμο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται έγκαιρα. Ε, σχετικά με αυτό θα δώσω μια διακήρυξη. Τέλος, πολιτική καθοδήγηση για την ε, ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Αυτό σημαίνει σχεδιασμό ικανοτήτων για τον οργανισμό συνορφυλακής και ακτοφυλακής, ε, αυξημένη ε, συνέπεια με τις υπόλοιπες εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Με αυτό τον καινούριο κανονισμό και ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη θα έχουν εργαλεία για να αντιδρούν και να προβλέπουν μελλοντικέ κρίσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τέλος, θα βοηθήσει αυτό στη διατήρηση της, ε, ε, του χώρου Σέγγεν ελεύθερης διακίνησης. Θα βοηθήσει στη διατήρηση του χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναμφίβολα η νέα εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλάκων Ακτοφυλάκων είναι σημαντικό βήμα ε, ως ευρωπαϊκή αντίδραση για το μεταναστευτικό. Ε, προβλέπεται αύξηση σε 10.000 άτομα, ε, ε, πλοία, αεροσκάφη. Ε, έτσι θα μπορέσει να είναι πιο λειτουργικός οργανισμός και να σώζει και ζωές. Χρειάζονται πόροι. Γι' αυτό αυτό θα λειτουργήσει μόνο αν ε, συμφωνήσουμε σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πολιετές και διευρυμένο. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ε, της Αυστρίας, για παράδειγμα θα ήθελα να πω ότι όποιος θεωρεί σημαντική τη φύλαξη των συνόρων θα πρέπει να πληρώσει και ε, μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Αυτό είναι κομμάτι μόνο μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και σίγουρα είναι και ε, μια πολιτική που εκφράζει ε, αλληλεγγύη επίσης ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοέλιο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και Επίτροπε, κύριε Βραμόπουλε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έγκριση αυτή τη νέα ενισχυμένη ενεργοφυλακή και είναι ένα ιστορικό βήμα για μια κοινή προστασία των εξωτερικών μα συνόρων. Σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία ε, στο χώρο Σέγγεν. Μιλάμε για 10.000 ακτοφυλακέ που μπορούν να μεταφερθούν ε, στις χώρες όπου είναι πιο ευάλωτα τα σύνορα ή όταν προκύπτει κάτι επίγον. Αυτό δεν πρέπει βεβαίως να οδηγεί στα κράτη-μέλη να μην τηρούν τις ε, ε υποχρεώσεις τους. Τα, μισά από τα άτομα αυτά, από τους οκτωφύλακες, θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Η Πορτογαλία θα είναι έτοιμη το 2021 να στείλει 110 ε, συνοριοφύλακες. Ε, όμως, παραδείγματος χάρη, κάνουμε κάτι, κάποιες υποσχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις οποίες ενδεχομένως τα κράτη-μέλη δεν μπορέσουν να τηρήσουν στη συνέχεια. Οι... Θα έχουν επίσης έναν ισχυμένο ρόλο ε, για την επιστροφή ανθρώπων που παραμένουν παράνομα στη χώρα μας. Το ένα τρίτο των αποφάσεων όμως εφαρμόζονται, των αποφάσεων, αποφάσεων επιστροφής. Για την Πορτογαλία δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα των δευτερογενών μεταφορών μεταφορών, μετα, μετα ε, βιβάσεων. Και έχουμε δει ότι τέσσερα κράτη-μέλη, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, κατάργησαν τη Σέγγεν. Ε, και να πω κάτι τελευταίο έκανε για τον εισηγητή που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά ο κύριος Νίντερ Μιούλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε, χωρίς την οποία δεν θα είχαμε καταφέρει να εκπονήσουμε αυτή την νομοθετική πρόταση. Να ευχαριστήσω όμως και τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο και όλο το προσωπικό του γραφείου του για την πολύ στεναρή υποστήριξή του. Το 2015 αυξήθηκε δραματικά ο αριθμό των μεταναστών που φτάναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Κατά συνέπεια, το 2016 είχαμε τη νέα πρόταση για τον Frontex. Η υφιστάμενη πρόταση αποτελεί μια θεωρωμένη πρόταση τη προηγούμενη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ακούσαμε, αυξάνεται το πεδίο εφαρμογή του οργανισμού πλέον και δίδονται περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι, καθώ επίση και περισσότεροι εμπειρογνώμονε και μεγαλύτερο προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων να διασφαλίσουμε ότι ο Frontex θα εξακολουθήσει να σώζει ζωές όσων διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπολοιπόμεθα από την βασική μας αυτή ανθρωπιστική υποχρέωση. Δεν μπορεί ποτέ κυβερνήσεις, υπουργοί να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές για εσωτερικούς καθαρά πολιτικούς λόγους. Παράλληλα τώρα η πρόταση αυτή δίνει στον οργανισμό αυτό περισσότερες αρμοδιότητες στην εφαρμογή των επιστροφών, για όσους δηλαδή δεν έχουν καταφέρει να πάρουν άσυλο. Αυτό όμως θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να δίδεται καμία νομική δυνατότητα στον οργανισμό να συμμετέχει σε επιστροφές από μία τρίτη χώρα προς μία τέταρτη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση αυτή θα ενισχύει τι υποχρεώσει και τι δεσμεύσει του οργανισμού αυτού όσον αφορά τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Τέλο, είναι λυπηρό το ότι ε, ενώ καταβάλαμε προσπάθειες για να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο από την άλλη δεν κατάφερε να καταλήξει μια συμφωνία όσον αφορά το κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου παρεμποδίστηκε τελικά λόγω καθαρά εσωτερικών πολιτικών λόγων και νομίζω ότι ε, και η έγκριση της προκαταρκτικής συμφωνίας ε, όσον αφορά την υπηρεσία αυτή τελικά δεν ευωδόθηκε λόγω εσωτερικών εθνικών εγωισμών. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την έκθεση, ένα ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων και αυτό σαφώς θα απασχολήσει και την επόμενη νομοθετική θητεία. Ο κύριος Βίστησεν τώρα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Τα εξωτερικά σύνορα με έως τώρα, από ό,τι φαίνεται, ποτέ δεν ήταν αντικείμενο ε, πραγματικής ε, προστασίας. Αυτό μας λέτε σήμερα με αυτό το νομοθέτημα. Γι' αυτό το λόγο, 18 χρόνια μετά τη Σέγγεν, ήρθε η ώρα νομίζω να έχουμε μια υπηρεσία συνόρων. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το συμβασμό που προέκυψε από τον Τρίλογο είναι ότι φοβούμαστε ότι είναι πολύ λίγα αυτά που προτείνεται και έρχονται πολύ αργά. Πολλές δικλείδες ασφαλείας ε, δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε την επιστροφή σε τρίτες χώρες. Ε, αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε μία λύση η οποία όμως δεν θα ικανοποιήσει κανέναν, ούτε τους πολίτες, ούτε θα είναι πιο ασφαλές το Σέγγεν. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσπα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Σεπτέμβριο του 2018 ο πρόεδρος Γιούνκερ παρουσίασε μια νέα μεταρρύθμιση της υπηρεσίας Frontex. Και πριν από δύο χρόνια ε, ήμουν εισηγήτρια και είχα χαιρετήσει ε, την το αποτέλεσμα τη πρώτη αναθεώρηση. Στο όνομα τη ομάδα μου σήμερα κάνω πάλι το ίδιο. Σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο ρεκόρ. Λυπάμαι βέβαια ε, για κάποια σημεία. Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένη για το πόσο γρήγορα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση του ζητήματο αυτού με μια ισορροπημένη προσέγγιση, αποτελεσματική για την προστασία των συνόρων μα, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω μα το ζητούσαν οι συμπολίτε μα σημειώνω κυρίω και χαίρομαι γι' αυτό ότι γίνεται ένα πραγματικό βήμα προ τα μπρο σε δημοσιονομικό επίπεδο, σε επίπεδο δυνατοτήτων δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, όπω μόλι αναφέρθηκε. Δύο στοιχεία θα ήθελα όμω να τονίσω. Χαίρομαι που λαμβάνουμε γνώση τη δημιουργία μια μόνιμη δύναμη που θα αποτελείται από 10.000 ακτοφύλακε και νοριοφύλακε και όπου τα κράτη-μέλη θα οφείλουν να συνεισφέρουν είναι πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό, πιο συγκεκριμένο από αυτήν, το, αυτό το απόθεμα των 1500 ανθρώπων που είναι διαθέσιμο υποτίθεται, αλλά με ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Είναι λοιπόν ένα χρήσιμο, ένα απαραίτητο βήμα και συγκεκριμένο. Δεύτερον, ε, ω εισηγήτρια στην αναθεώρηση, είχα ζητήσει στο τελικό κείμενο να γίνει μια αναφορά στη δημιουργία ενό κέντρου κατάρτιση Frontex. Διότι αν θέλουμε να ξεπεράσουμε ε, την εθνική ε, προσέγγιση για την προστασία των συνόρων, διότι τα κράτη-μέλη προφανώ και είναι αρμόδια και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όμω, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερη κυκλοφορία, τη Σέγγεν δηλαδή, εάν θέλουμε να είναι όσο γίνεται λιγότερα τα κενά, πρέπει να είμαστε Ευρωπαίοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ευρωπαϊκό. Και η υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με τι αρχέ των κρατών μελών. Όχι μόνο να τι υποστηρίζει, να συνεργάζεται μαζί του. Για να μπορεί να γίνει όμως αυτό στην πράξη θα πρέπει να αναπτύξουμε μια, μια πραγματική ευρωπαϊκή κουλτούρα σε επίπεδο κατάρτισης. Αυτό ακριβώς ε, ζητεί το κείμενο και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Ρομπέρτα Μετσόλα, την εισηγήτρια, η οποία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έδειξε μεγάλη ενέργεια, αποφασιστικότητα και χάρη σε αυτήν μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Σε λίγες ώρες ε, η ομάδα μου θα υποστηρίξει στην ψηφοφορία αυτήν τη νέα μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αλμπιόλ Γκούθμαν. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Τελειώνει αυτή η θητεία και, και ουσιαστικά όσοι κυβερνούν την Ευρώπη έχουν εγκαταλείψει οποιαδήποτε ανθρωπιά. Πολιτικές που βασίζονται ουσιαστικά στον θάνατο των ανθρώπων στη θάλασσα, ε, στη σκλαβιά τους, ε, τις, ε, τα βασανιστήρια σε κέντρα κράτηση και τον εκτοπισμό του σε χώρε όπου δεν υπάρχουν καμία εγγύηση ότι θα γίνουν σε αυτά τα δικαιώματά του. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ε, ε, τρόποι εισόδου νόμιμοι και ασφαλεί. Ε, δεν υπάρχουν ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Πλέον δεν επιτρέπουμε καν στι μη κυβερνήσει οργανώσει να κάνουν τη δουλειά αυτή, η οποία είναι απαραίτητη. Κάποια στιγμή θα, θα περάσουν από δίκη η, πολιτική θύμητος για τις πάνω από 17.000 νεκρούς των τελευταίων 5 ετών στη Μεσόγειο. Οι πολιτικές τους που κλείνουν τα σύνορα και που ε, ουσιαστικά υποχρεώνουν τους μετανάστες να παίξουν τη ζωή τους γράμματα οδηγούν στο θάνατο 10 ατόμων τη μέρα. Και ο κανονισμός που ε, ψηφίστε σήμερα ουσιαστικά είναι το απάβγασμα αυτής της απάνθρωπης πολιτικής είναι ένα, ε, μια παραστρατιωτική οργάνωση με 10.000 ανθρώπους με 2 δισεκατομμύρια ευρώ προπολογισμό για να ε, κλειδαμπαρώσουν τα σύνορα, για να εκτοπίσουν τους ανθρώπους, για να κλείσουν τους ανθρώπους σε κέντρα ε, ε κράτησης. Είναι ουσιαστικά το ε, ο στρατιωτικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όνειρο της ακροδεξιάς που το κάνουν πραγματικότητα φιλελεύθεροι σοσιαλιστές και συντηρητικοί. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία και την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Νομίζω ότι είχαμε πολύ επικοδομητική θέση ως Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στη διάσωση και την έρευνα. Εμείς ε, φροντίσαμε η Frontex να έχει κατάλληλη εντολή έρευνας διάσωσης λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης που βλέπουμε να ε, λαμβάνει η χώρα στη Μεσόγειο. Η πλειοψηφία ετάχθη υπέρ αυτών. Αλλά τα κράτη-μέλη ψήφισαν διαφορετικά. Ε, μπλοκάρισαν τις προσπάθειες της εισηγήτριας να ενισχύσουν τη διάσωση στο κείμενο του νομοθετήματος. Και αυτό είναι πρόβλημα πραγματικό. Η Frontex μπορεί να διασώζει μόνο ανθρώπους στα πλαίσια και στα, μέσα στα όρια της επιχείρησης διάσωσης και ε, είναι πολύ μικρή περιοχή, λίγο έξω από τη Σικελία. Δεν είναι αυτή η περιοχή όπου υπάρχει το πρόβλημα και πνίγεται κόσμος στη Μεσόγειο. Τώρα που μιλάμε και παρακολουθούμε, ξέρουμε που είναι. Οι δεταγμένες είναι σαφείς. Κανείς δεν πάει όμως να διασώσει αυτούς τους ανθρώπους. Οι ε, κυβερνητικές οργανώσεις ε, ποινικοποιούνται, τους παίρνουν τα πλοία δεν γίνονται επιχειρήσεις και η ε, ε, έρευνα και διάσωση ε, έγινε στη, κοντά στη Λιβύη, αλλά διασώσεις δεν γίνονται, γιατί τώρα ξέσπασε πόλεμος πάλι εκεί. Έτσι παραβιάζεται η υποχρέωση διάσωσης μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρχει στη Μεσόγειο ε, οργάνωση σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, ε, τα κράτη-μέλη δεν, να, δεν είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε με συντονισμένο τρόπο, αλλιώς θα καταρρεύσουν οι αξίες της Ευρώπης μαζί με τους πνιγμένους. Είχεστε μπλε κάρτα, κυρία Κέλλερ. Όχι. Λυπάμαι, προσπάθησα πάντως. Η κυρία Τζέιμις τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μάταιες προσπάθειες να αντιμετωπίσει μια πολιτική μετανάστευση ε, χωρίς νόημα. Ε, 11 δις ευρώ δαπανώνται ε, γι' αυτό. Ο Φρανς Τίμερμανς είπε τον περασμένο μήνα ότι η Ευρώπη δεν βιώνει πια την ε, μεταναστευτική κρίση του 2015 και 2016. Ε, ο Λίβιος Πρωθυπουργό όμως ανακοίνωσε ότι 800.000 τουλάχιστον μετανάστες από τη Λιβύη ε, θα προσπαθήσουν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχουμε 11 δις, έχουμε 10.000 συνοριοφύλακες και οι διακινητές ανθρώπων δεν έχουν καταθέσει τα όπλα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τα δικά του προβλήματα πέραν της μάχης. Τώρα ε, έχουμε ανοιχτή Ευρώπη μετά την πολιτική Μέρκελ η οποία μας δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Ο κύριος έχει λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι φτάνανε όλο και περισσότερα κύματα μεταναστών και προσφύγων που ουσιαστικά επιβάρυναν πάρα πολύ την Ιταλία αλλά και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνιμο αυτό σώμα των 10.000 ατόμων ουσιαστικά θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις εσωτερικές δυνάμεις των κρατών μελών, καθότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συνεισφέρουν στη στελέχωση αυτού του μόνιμου σώματος. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να ανακουφίσει οικονομικά τα κράτη-μέλη. Πέρα από όλο αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, τα οποία δεν δίνανται να συνεισφέρουν σε προσωπικό ή χρηματοοικονομικά, ακριβώ επειδή υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί οικονομικοί περιορισμοί όσον αφορά τον εθνικό μα προπολογισμό. Πώ μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικά. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το μόνιμο σώμα δεν θα είναι αρκετά αποτελεσματικό. Ενδεχομένω να ήταν αποτελεσματικό στα χερσαία μόνο σύνορα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματικό και επιχειρησιακό στα θαλάσσια σύνορα. Σε περιπτώσει όπω αυτέ που αντιμετωπίσουμε στην Ιταλία, που βλέπουμε να φτάνουν εκατοντάδε μετανάστε και πρόσφυγε, οι οποίοι διασχίζουν την θάλασσα που μας χωρίζει από χώρες όπως η Λιβύη. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ανανεωθεί η επιχείρηση Σοφία και να καταφέρουμε τελικά εκ νέου να έχουμε θαλάσσιες αποστολές. Αντίθετα, υπαναχωρούμε, οπισθοδρομούμε με το νέο αυτό κανονισμό. Νομίζω ότι η εθνική κυριαρχία θα μειωθεί εξαιτία του νέου αυτού οργανισμού. Του τελευταίου μήνε η Ιταλία κατάφερε να μειώσει την έλευση των μεταναστών και κατάφερε σε σχέση με το 2017 να μειώσει την έλευση αυτή κατά 80%. Αυτό όμω δεν έγινε χάρη στη μεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χάρη στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση τη χώρα μου. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό οργανισμό. Ο κύριο Συναδεινό έχει το λόγο για ένα λεπτό κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό έπειτα από πέντε έτη ενεργής παρουσίας χαίρομαι που η πολιτική της ένωσης προσαρμόζεται και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και όσα οι πατριωτικές φωνές υπεύθυνα απαρέγκλιτα και πιστά δήλωναν και δηλώνουν για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης για τη διασφάλιση των πολιτών μας και των ζωτικών μας συμφερόντων για την ανάσχεση των λαθρομεταναστευτικών εισρωών απαιτούνται ισχυρά και ασφαλή σύνορα υπό εθνικό έλεγχο και απόλυτη αυτονομία δράσεων από πλευρά των κρατών μελών παρά το όποιο κοινό πεπρωμένο εθνική κυριαρχία που μοιράζεται δεν ισχυροποιείται και δεν πολλαπλασιάζεται. αντιθέτω ασθενεί και απεμπολείται. τα σύνορα δεν ομοσπονδοποιούνται δεν συνδιαχειρίζονται πολύ απλά καταλύονται. επιπλέον η οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση συνόρων είναι ψευδεπίγραφη. τα σύνορα είναι σύνορα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ή παραποίηση. η ένωση ενδιαφέρεται βέβαια μόνο για την εξασφάλιση του συμφερόντων της γερμανίας και των στενών συμμάχων δεν κόπτεται για την προστασία συνόρων αλλά για να παρκάρει τους λαθρομετανάστες στις χώρες της περιφέρειας όπως είναι η ελλάδα και η ιταλία. ευχαριστώ. Λένερς, ε, λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα εξωτερικά σύνορα της Ολλανδίας ε, έχουν πάει στη Λαμπεντούζα πια. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και αυτή την πρόκληση θα την αντιμετωπίσουμε μόνο με τη συνεργασία. Αν στο μέλλον θέλουμε να έχουμε όφελος από το Σέγγεν και να μην έχουμε εσωτερικά σύνορα, όταν θέλουμε να ξέρουμε ποιος έρχεται στην Ευρώπη και γιατί, αν θέλουμε να ελέγξουμε τη μετανάστευση και να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν άσυλο θα επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης, αν τα θέλουμε όλα αυτά, τότε είναι σημαντική η ενίσχυση του Οργανισμού Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής. Αυτοί οι 10.000 χρειάζεται να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα και αυτός είναι και τρόπος οργάνωσης της διαχείρισης των σύνορων μας. Διότι είναι καλό να υπάρχει κάτι όχι ε, μόνο όταν χρειάζεται, αλλά να υπάρχει μια μόνιμη βάση υποστήριξης. Το μόνιμο σώμα θα βοηθήσει εδώ. Θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες η ακτοφυλακή και η συνοριοφυλακή να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και να τις βοηθάει τις τρίτες αυτές χώρες για να σταματάει η παράτυπη μετανάστευση και να διασφαλίζεται η επιστροφή των ανθρώπων αυτών. Είναι σημαντικό και αναγκαίο βήμα αυτό για την βελτιωμένη επιτήρηση των συνόρων να βελτιώσουμε τη διαχείριση των συνόρων. Ευχαριστώ τη Ρομπέρτα Μέτσολα για ε, ε, την ε, αποτελεσματική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση του Οργανισμού Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως μπερδεύουν τα ασφαλή σύνορα με την πλήρη απομόνωση και ε, έτσι καταδιώκουν ανθρώπους ε, και τους στέλνουν στα χέρια των διακινητών. Η, τα, η, η απόρρια αυτής της πολιτικής φαίνεται στη Λιβύη τώρα. Δεν φτάνει ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν αναλαμβάνουν τις χριστιανικές τους ευθύνες, αλλά αν ακολουθούσαμε τους συντηρητικούς θα έπρεπε να ε, αναθέσουν τις επιστροφές σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μεταθέτει δηλαδή ίδιες ευθύνες σε άλλους. Αυτό το απορρίψαμε με επιτυχία. Το Συμβούλιο που λάμπει σήμερα δια της απουσίας του πότε θα ε, ολοκληρώσει ένα πακέτο για το ε, άσυλο που θα είναι ισορροπημένο. Πότε θα υπάρξουν ενιαίοι κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο βιώσιμο και μακροπρόθεσμο τις προκλήσεις στα σύνορα και θα ε, ανταποκριθούμε και ε, όπως πρέπει στις κοινέ μας αξίες. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Σόιντροβα. Οπωσδήποτε όχι, ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ε, Μπέρντ Κέλμελε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση η Frontex και προσωπικό περισσότερο χρειάζεται. Είναι σωστό το μέτρο. Παράλληλα, ε, οι 10.000 ε, δημιουργούν ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα της Ένωσης δεν θα τα λύσουμε ζητώντας μόνο περισσότερα χρήματα αυτό που χρειάζεται για τη μετανάστευση είναι μία ρύθμιση νομοθετική ευρεία που θα δώσει ε, τη δυνατότητα ανάληψης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο έλεγχο στα σύνορα, πρέπει να μπορούμε να αποφασίζουμε ποιος μπορεί να μπαίνει και ποιος δεν μπορεί να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εδώ έχουμε μια πλειοψηφία που αναζητεί απλές λύσεις και νομίζει ότι θα καλύψει τα προβλήματα με λεφτά. Ενώ τα προβλήματα στην πραγματικότητα επιδεινώνονται. Και οι νέοι δεν θα είναι έτοιμοι όταν θα ξεσπάσει νέα κρίση. Και αυτό σίγουρα δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Αν θέλουμε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στους πολίτες, πρέπει τη βούληση των πολιτών να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας στα σοβαρά. Και χρειάζεται να γίνει κάποια στιγμή μια σωστή συζήτηση για αυτό το θέμα. Η κυρία Βίξτρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Ρομπέρτα Μέτσολα για την πολύ καλή δουλειά τη. Σα ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ετών. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την πολύ καλή αυτή πρόταση. Όταν πετάω στην Ευρώπη, εγώ δεν βλέπω σύνορα. Αυτό το είχε πει ο πρώτο πρόεδρο τη ελεύθερη Τσεχοσλοβακία, ο Βάκλαβ Χάβελ η μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής ένταξης, η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, βασίζεται στο να έχουμε ισχυρά εξωτερικά σύνορα. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη οχυρό. Δεν θέλουμε να διώξουμε ανθρώπους. Θέλουμε να ελέγχουμε τις ροές των ανθρώπων που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται ένα σωστός έλεγχος ασφαλείας, υπάρχει μια διέλευση συντεταγμένη για όλου όσου έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντα ε, ε, διεθνή προστασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών, ε, παράνομων ουσιών που δεν θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση που εγκρίνουμε σήμερα δεν πάει προ ένα πλήρε ομοσπονδιακό σύστημα. Για μένα αυτό είναι ο σωστό δρόμο, αλλά έχουμε γίνεται ένα πρώτο βήμα από τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα Κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι εγώ είμαι 10 χρόνια εδώ. Είναι από τις τελευταίες μου ομιλίες ε, στο Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλους όσους με τους οποίους συνεργάστηκα. Ε, όταν τελειώνει η πολιτική, η φιλία μένει. Και είναι μια ευκαιρία και μια νέα αρχή. Ευχαριστώ. You are an optimist. Sometimes politics... Ε, είστε αισιόδοξοι. Καμιά φορά η, η πολιτική καταστρέφει φιλίε, τέλο πάντων. Ελπίζω να ισχύσει αυτό που λέτε στην προηγουμένη περίπτωση. Η κυρία Φορέντζα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 1.311 θάνατοι μόνο και μόνο το 2018. Αυτό είναι ο απολογισμός των θανάτων στη Μεσόγειο. Και εμεί συνεχίζουμε και συζητάμε εδώ πέρα για σύνορα και για ενίσχυση της πολιτικής επιστροφών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Καταρχάς, θα πρέπει να κηρύξει ως μη ασφαλής τους λιμένες της Λιβύης. Το έχει κάνει αυτό επίσημη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχουν κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούν ότι είναι ασφαλεί οι επιστροφέ στη Λιβύη και στι χώρε αυτέ συγκαταλέγεται και η Ιταλία. Αν πραγματικά θέλουμε να μας θυμόμαστε, να μας θυμάται ο κόσμος ως αυτοί που αύξησαν τους θανάτους στην Μεσόγειο, τότε δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό. Το αντίθετο όμως θα έπρεπε να ελπίζουμε. Σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραπέμπουμε στις λιβικές αρχές την όλη αρμοδιότητα και ευθύνη της έρευνας και της διάσωσης. Καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία με την αστευτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης. Ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ακολουθούμε την πολιτική του Σαλβίνη. Πρέπει να είμαστε μια πολιτισμένη ήπειρο. Η κυρία Βαλέρο έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για του πρόσφυγες, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που φεύγουν από τι χώρε του εξαιτία ένοπλων συγκρούσεων και από ό,τι φαίνεται η τάση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Θα έχουμε όλο και μεγαλύτερα μεταστευτικά κύματα εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε εκατομμύρια κλιματικών λεγόμενων προσφύγων. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και του 600.000 πολίτε οι οποίοι θα πληγούν λόγω τη αύξηση τη στάθμη τη θάλασσα σε διάφορε χώρε. Οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να έρθουν προ την Ευρώπη, όχι όλοι βέβαια, αλλά εμεί πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτού οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν προ την Ευρώπη. Επενδύουμε αυτή τη στιγμή τεράστια ποσά προκειμένου να του απομακρύνουμε, προκειμένου να του κρατήσουμε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έπρεπε να τα δίνουμε για την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών, αλλά περισσότερο για τη μείωση τη φτώχεια και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσή του. Ο κύριο Κορά, όχι το λόγο τώρα για μισή λεπτό. Α το πούμε ξεκάθαρα, αγαπητοί συνάδελφοι, απέτυχε η μεταρρύθμιση του κοινού συστήματο ασύλου. Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια τίποτα δεν έγινε προκειμένου να τροποποιηθεί η Συμφωνία του Δουβλίνου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι βυθίζεται σε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο η Λιβύη και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ζωές από τη Λιβύη. Νομίζω ότι η Frontex αυτή τη στιγμή είναι το μόνο εργαλείο το οποίο έχει απομείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικεύει το, το πρόβλημα αυτό, δίνει χρήματα σε τρίτε χώρε για να κάνουν αυτέ τη βρώμικη δουλειά. Και από την άλλη η μεταρρύθμιση του Frontex συνάδει ουσιαστικά με την πολιτική αυτή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, ελπίζουμε μέσω της μεταρρύθμισης αυτής, ελπίζουν ορισμένοι τουλάχιστον, να κερδίσουν περισσότερες ψήφους στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Ανταυτού όμως ε, θα έπρεπε να είχαμε περισσότερη ευρωπαϊκή ελληνική, την οποία όμως δεν θέλουν καν να ακούσουν, ούτε καν ως ιδέα, ως έννοια, ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο οι χώρε εκείνε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίε καλούνται να διαχειριστούν τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω επίσης ότι ε, στις ε, χώρες αυτές θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν ακόμα και εσωτερικούς ελέγχους, τη στιγμή που τους ελέγχους αυτούς δεν μπορεί να κάνει ο οργανισμός, ο Frontex. Κανονικά η αρχή της αλληλεγγύης υποτίθεται ότι προβλέπεται από τις συνθήκες, αλλά στην πράξη δεν ισχύει, δεν λαμβάνει χώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη πως ο Frontex είναι το πλέον ανεπιτυχές πείραμα για να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να τον αναβαθμίσει και να τον μετατρέψει σε οργανισμό ευρωπαϊκής Ακτοφυλακή και συνοριοφυλακής. Ε, το αυξάνει την επιχειρησιακή δύναμη σε δέκα χιλιάδε άτομα και σε περιόδους αγρίας λιτότητας φορολογεί τους ευρωπαίους πολίτες και σπαταλά τα χρήματά τους για να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό άρα και άχρηστο οργανισμό. η αιμονή όμως και η σκοπιμότητα να αφαιρεθούν από τα εθνικά κράτη αρμοδιότητες ζωτικές για την επιβίωσή τους όπως είναι η ασφάλεια των συνόρων οδηγεί την ευρωπαϊκή ένωση να λάβει αποφάσεις που αντίκειται στην κοινή λογική διότι ποιο λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο θα διαφωνήσει με την άποψη ότι η καλύτερη προστασία των συνόρων ενό κράτου επιτυγχάνεται εάν η αποστολή αυτή δοθεί στι ένοπλε δυνάμει και τα σώματα ασφαλεία του κράτου αυτού. η ορθότητα αυτή τη απόψεω έχει αποδειχθεί στην πράξη διότι όλα τα κράτη τα περισσότερα κράτη τη ευρωπαϊκή ενώσεω κλείνουν τα σύνορά του για να αντιμετωπίσουν τα ανεξέλεγκτα κύματα των λαθρομεταναστών και έτσι μεταφέρουν το πρόβλημα στα κράτη εισόδου όπω είναι η ελλάδα η οποία εάν δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει μόνη της να προστατεύσει τα σύνορά της ουδής μαθητευόμενος μάγος της ευρώπης θα τη βοηθήσει υπό οποιαδήποτε μορφή και όνομα και αν εμφανιστεί αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διάς Δεμέρα τώρα έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, θέλω να συγχαρώ τη Ρομπέρτα για την καλή δουλειά της Υπενθυμίζω όμως ότι οι πιο σημαντικέ προτάσεις του πακέτου ασύλου και μετανάστευσης ε, μένουν αυτή τη στιγμή κολλημένες στον τρίλογο. Ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητε ε, σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή στην Οριοφυλακή και θα ψηφίσουμε υπέρ. Είναι σημαντικό να ψηφίσουμε υπέρ αυτού του εργαλείου για να υπάρχουν απαραίτητε δυνατότητε που θα εγγυηθούν μια ολοκληρωμένη διαχείριση τη μετανάστευση με αποτελεσματικότητα και με ένα υψηλό επίπεδο ασφάλεια στο εσωτερικό τη Ένωση Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίω να διαφυλάξουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η δημιουργία ενό σώματο 10.000 ανθρώπων, η υποστήριξη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι επιστροφέ ή η εντετικοποίηση τη συνεργασία με τρίτε χώρε είναι πολύ σημαντικά επιχειρησιακά στοιχεία για να εγγυηθούν μια συνεχή υποστήριξη και για τις χώρες προορισμού και για τις χώρες προέλευσης και για τις χώρες transit. Από κοινού τη Europol αυτή η νέα υπηρεσία θα είναι η λιδία λίθος που θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε το έργο μας για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερε επιχειρησιακέ, να δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερε επιχειρησιακέ και δημοσιονομικέ δυνατότητε σε αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει βεβαίω και μια δικλίδα ασφαλεία, διότι αυτή, αυτό το σώμα υπόκειται στο δίκαιο τη θάλασσα, στο διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο και στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαγιών έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σίγουρα χρειάζεται καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό για την καλύτερη λειτουργία του χώρου Σέγγεν, για την ε, ρύθμιση της μετανάστευσης. Χρειάζονται συμφωνίες ε, για την ε, επέκταση και ενίσχυση του Frontex. Θα ψηφίσω υπέρ. Είναι σημαντικό να έχουμε την αύξηση αυτή ε, στις 10.000 μέχρι το 2027. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την βασική ευθύνη για τη διαχείριση των συνόρων τους και θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατέψουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που θα επιστραφούν από τη Frontex στις τρίτες χώρες. Η συνεργασία με τρίτες χώρες ε, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νέων συμφωνιών που θα λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, προσοχή, οι νέοι κανόνες για τα εξωτερικά σύνορα δεν θα πρέπει να ισχύουν χωρίς να προσαρμοστούν και για τον ε, ευρωπαϊκό εξωτερικό χώρο. Ευχαριστώ. Ο κ. Τσαμπάσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σαφώς θα πρέπει όλα αυτά τα χρήματα να δοθούν στο νέο αυτό οργανισμό. Τα εξωτερικά σύνορα είναι θεμελιώδους σημασίας, προκειμένου πραγματικά να έχουμε ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χαιρετίζω την διευρυμένη αυτή αρμοδιότητα που δίνεται στο νέο αυτό Frontex, και είμαι σαφώ υπέρ τη θέσπιση του μόνιμου αυτού σώματο με επιχειρησιακή δύναμη 10.000 ατόμων. Το έχω πει πολλά και στο παρελθόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού για να σταματήσουμε την έλευση των παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικοί μετανάστε, οι οποίοι δεν δέχονται τι αξίε μα και τον τρόπο ζωή μα, δεν έχουν καμία θέση στι χώρε μα ούτε βέβαια και οι τρομοκράτε, ε, οι οποίοι χρησιμοποιούν πολλέ φορέ τις οδού μετανάστευση. Σα ευχαριστούμε. Ουρτασούν παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η θητεία θα περάσει την ιστορία για την τροπή των 18.000 νεκρών στη Μεσόγειο σύμφωνα με τη Διεθνή ε, Οργανισμό Μεταναστών και το τελειώνουμε τη θητεία με το χειρότερο τρόπο με, τον, με την μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, του κανονισμού του ασύλου που έχουν μπλοκαριστεί και έχουμε τώρα αυτόν τον νέο κανονισμό για μια ακτοφυλακή, συνοριοφυλακή με δισεκατομμύρια που διατίθενται χωρίς να υπάρχει ένας μηχανισμός που να διαφυλάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς μια σαφή εντολή για την διάσωση στη Μεσόγειο όπως είχε ζητήσει αυτό το κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευσή της και στην πραγματική εντολή της το έχουμε ζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν οι κυβερνήσει τελικά ποινικοποιούν τις ΜΚΟ όπως το Open Arms που δεν μπόρεσε, μπόρεσε να ε, φτάσει να, να, να πιάσει λιμάνι στη Βαρκελόνη ε, ποινικοποιούμε λοιπόν τις ΜΚΟ ε, και δεν γίνεται αναφορά σε μια δημόσια προσπάθεια διάσωσης. Είναι πραγματικά μια ντροπή. Στη νέα θητεία θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάλ έχει, δύο, το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η Frontex τη θεωρία ε, θα μπορούσε να προστατεύσει τα σύνορα της Ένωσης όμως είναι ευθύνη των κρατών μελών κυρίως αυτό. Η ενίσχυση λοιπόν της, ε, των αρμοδιοτήτων της Frontex ε, είναι κάτι που θα μπορούσε να διακυβεύσει την ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν πρέπει να παρεμποδιστούν τα κράτη-μέλη από το να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν συνεργασία. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό στην πράξη. Ανησυχούμε, διότι η συμφωνία που επετεύχθη δεν επιτρέπει στην Frontex να έχει την υποστήριξη των αρχών ε, σε τρίτες χώρες όπως τη Μακεδονία και δεν θα μπορεί να βοηθήσει για την επιστροφή των πάνω μεταναστών. Εμείς θα πάντα να υπάρξει μια ενίσχυση ε, των συνόρων και έχουμε καταφέρει εμεί να προστατεύσουμε τα σύνορά μα χωρί την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Η Ουγγαρία όμω δεν είδε ποτέ λεφτά για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Γκυλιόμ. Ίσως να ήταν τελικά απαραίτητο να ενισχυθεί η υπηρεσία Frontex, διότι τα κοινά μα σύνορα πρέπει να τύχουν διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή τη μεταρρύθμιση ε, τη Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή που πρέπει να συνοδεύεται όμω από το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων όσων ελέγχονται στα σύνορα, τα εξωτερικά τη Ένωση. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ και σε δύο παράπονα που έχω στο τέλο τη θητεία αυτή. Λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε μία ε, αποστολή διάσωσης στη γη πάνω από 1.800 ε, άνθρωποι πέθαναν το 2018 άνθρωποι κινδυνεύει η ζωή του, Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί με τέτοια υπηρεσία να το κάνει αυτό. Ε, εδώ και έξι μήνε οι ΜΚΟ το κάνουν αυτό ε, στην θάλασσα. Ε, κλείνουν τα σύνορα, τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν οι μετανάστε να προσπαθούν να περάσουν και βεβαίω υπάρχει δεύτερη μεταρρύθμιση τη Frontex, ε, χωρί να υπάρχει καμία μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά το καθεστώ ασύλου. Και γι' αυτό λυπάμαι και φταίνουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό που μπλοκάρουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, ενώ το Κοινοβούλιο έχει θέσει τη θέση του επιτάπητο εδώ και δύο χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Τόμας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Frontex πρέπει να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αλλά είναι λάθος η κατεύθυνση που του δίνουμε το οργανισμό αντί να εξειδικεύεται σε επίγουσες καταστάσεις και γρήγορη αντίδραση, δημιουργούμε γραφειοκρατικές υπηρεσίες τώρα. Είναι αμφισβητούμενο το πόσο θα αποδώσουν. Πρέπει να λύσουμε άμεσα τα προβλήματα. Η Frontex δεν μπορεί να ε, συμμετέχει σε επιχειρήσεις από τρίτες σε τρίτες χώρες. Δεν θα μπορεί να επιστρέψει ε, από τις, βόρειες Ευρω... Ε, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις χώρες από όπου προέρχονται. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να αντιμετωπίζουμε το οργανωμένο ε, έγκλημα και την παράτυπη μετανάστευση ε, στο κατόφλι των χωρών μας, ε, ενώ θα έπρεπε να γίνεται αυτό όσο γίνεται πιο μακριά. Σας ευχαριστούμε κύριο Ραγχέλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πουσιάζει όμως. Η κυρία Κιέγγε για ένα λεπτό τότε παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προώθησε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού που θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τι εσωτερικέ διχόνοιε, διαπραγματευτήκαμε και καταλήξαμε τελικά σε ένα κείμενο το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξο, αλλά σίγουρα θα συμβάλλει το να παγιώσουμε έναν από τους τέσσερις πυλώνες που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και αναφέρομαι βέβαια στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια στο πλαίσιο του πυλώνα αυτού καλεί την Ευρώπη να ενισχύσει τη δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Θα πρέπει προφανώ να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επομένως, η υποστήριξη της μεταρρύθμισης αυτής θα επιτύχει μόνο αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά και αν εξασφαλίσουμε επίσης τη δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και να κάνω μια έκκληση στο τέλος της θητείας αυτής. Σας παρακαλώ πολύ, εκινήστε εκ νέου την επιχείρηση Σοφία και δώστε τις μεγαλύτερες δυνατότητες έρευνας και διάσωση. Ο κύριος Ράντεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησα την εντολή μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την εποχή εκείνη η όλη ιδέα θέσπιση ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνορεφυλακής και Εκτοφυλακή ήταν ένα πολύ ασαφέ και θεωρητικό σχέδιο. Θεωρούσαμε ότι θα έβλεπε το φω τη ημέρα το νωρίτερο το 2030. Είμαστε όμω πάρα πολύ αφελεί τότε, γιατί μέσα σε ένα χρόνο είδαμε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστε και πρόσφυγε να καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασχίζοντα τα εξωτερικά μα ε, σύνορα και οι τότε συνοριοφύλακες δεν ήταν σε θέση να διχειριστούν ένα τόσο ακραίο φαινόμενο. Έπρεπε λοιπόν επιγόντως να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και συνειδητοποίησαμε ότι ο χώρο Σέγγεν είναι πάρα πολύ σημαντικός και ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Συνειδητοποίησαμε τότε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των εξωτερικών της σύνορων καταρχάς και τέσσερα χρόνια αργότερα να που συζητάμε για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής. Λέμε ότι θα εμπεριέχει και ένα μόνιμο σώμα με δύναμη 10.000 ατόμων. Συζητάμε επίσης για τις νέες αρμοδιότητες του οργανισμού αυτού. Μα νομίζω ότι ο οργανισμός αυτός από μόνος του αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών, αν θέλετε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα άνθρωποι είναι στο κατάλογο για το CatchDI. Θα ήθελα πραγματικά να δώσω σε όλους το λόγο, όμως σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό που θα σας δώσουμε, διότι στις πέντε ψηφίζουμε και έχει υπάρχει άλλο ένα θέμα στη μέση διάταξη πριν. Οπότε σας ζητώ πολύ ευγενικά να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό της παρεμβάσης σας. Η κυρία Σρόιντοβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόταση σχετίζεται με το με πολύ μεγάλο λάθος που έγινε το 2015-2016 όταν τα εξωτερικά σύνορα της Σέγγεν δεν προστατεύθηκαν καταλήλως και υπήρξε διέλευση έως και 2 εκατομμυρίων ανθρώπων μεταναστών και προσφύγων. Κάποιοι από αυτούς ήταν όντως πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις φρικαλαιότητες του. Όμως πολλοί από αυτούς δεν ήταν επιλέξιμοι για άσυλο και θα πρέπει να επιστραφούν. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξωτερικά τη σύνορα για λόγους ασφαλείας. Όταν έχουμε εκατομμύρια ε, μετανάστες οι οποίοι περνούν τα σύνορα, τότε η αίσθηση της ασφάλειας χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, μετά από τρία χρόνια ε, καλής λειτουργίας, η νέα αυτή υπηρεσία, λέει κυρία Πίκουλα, ε, ο κύριο Πίκουλα θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντό της Σέγγεν Καλωσορίζω λοιπόν την θέσπιση αυτής ε, της ε, ε, δύναμης είναι μια αντίδραση στους κινδύνους που υπάρχουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να εξετάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για την ε, χορήγηση ασύλου. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο Σέγγεν, έχει να κάνει και με την έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Είναι καλό ότι θα έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στίβενς, η κυρία Στίβενς. Κυρία, κυρία κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Πάντα είμαστε υπέρ του Frontex. Πρώτη φορά το 2016 ο Frontex ανέλαβε το καθήκον να παρεμβαίνει περισσότερο στις επιστροφές ε, μετά από απόρριψη ασύλου. Και τώρα ξανά υποστηρίζουμε τον Frontex. Γιατί πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Frontex έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. Μπορεί να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο με ισχυρά εξωτερικά σύνορα και εδώ θα μας βοηθήσει ο Frontex. Περισσότερο, περισσότερη πόροι, προσωπικό, θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα έτσι τις προκλήσεις. Ο Frontex θα πρέπει να δραστηριοποιείται και σε μη ε, κράτη-μέλη, ε, χώρες που βρίσκονται μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Frontex θα βοηθάει στις επιστροφές από το Μαρόκο προς μια άλλη χώρα μη μέλος, την Ιγυρία για παράδειγμα, τον Ήγυρα. Αυτό δεν μπορούσαμε, δεν το κάνουμε. Είχαμε χάσει αυτή τη δυνατότητα στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Να ε, πω ότι λυπάμαι ότι σε σημαντικό θέμα που ε, χιλιάδες ζωές εμπλέκονται και εκατομμύρια ε, ευρώ ε, δεν ε, γίνονται τακτές οι ερωτήσεις και δεν γίνεται καλή συζήτηση. Η λύση είναι το κράτος δικαίου. Αν, ο κόσμος, ε, ε, αν κάποιος επιδιώξει να μπει στην Ένωση παράνομα, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός κανόνας που θα λέει «Παρακαλώ, λυπάμαι, πρέπει να πάτε πίσω». Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει και νόμιμη οδός για την ε, αίτηση ασύλου γιατί όλα τα πολιτισμένα κράτη δέχονται το δικαίωμα του ασύλου για αυτούς που διώκονται. Το κράτος δικαίου είναι το βασικό. Τα 11 δις ευρώ και οι έξτρα πόροι και η γραφειοκρατία θα βοηθήσουν ε, ε, να λύσουμε το πρόβλημά μας, ε, ενώ ένας πρακτικός κανόνας θα ήταν καλύτερος. Μπόκοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να έχουμε ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στην Ευρώπη και προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο χώρος Σέγγεν. Δυστυχώ όμω δεν αντιμετωπίσαμε έτσι τα πράγματα του 2015. Επιτέλου όμω, τρία χρόνια μετά, συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την παράτυπη μετανάστευση και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποια βήματα ακόμα. Η εντολή του Frontex θα πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, να μπορεί να περιλαμβάνει και τις επιστροφές από τρίτη χώρα προς τρίτη χώρα. Στη Σλοβενία το 2015 είχαμε σε καθημερινή βάση χιλιάδες διελεύσεις των συνόρων μας και είδαμε ότι η τάση είναι ανωδική και του τελευταίου μήνε και δεν νομίζω ότι πρόκειται να τροποποιηθεί πολύ στο μέλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι έρχονται από τη Βοσνία ή τη Σερβία θα, μπορούν να, θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφονται χάρη στο Frontex. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι Ευρω... Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Ισπανός. Είναι πολύ καλή η στόχη ενός στόχου ελεύθερης, ε, ελευθερίας ε, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ε, ε, έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και σε αυτό θα μας βοηθήσει η ακτοφυλακή, η σνοριοφυλακή ευρωπαϊκή με μια ε, νέα δυνατότητα 15.000 ε, ε, ανθρώπους με σημαντική χρηματοδότηση. Εμείς οι σοσιαλιστές συνεισφέραμε στη βελτίωση του κειμένου με τροπολογίες για να μην υπάρξουν επιστροφές σε τρίτες χώρες και να το συνδέσουμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το χάρτη των Θεμελιών Δικαιωμάτων που ισχύει. Όμως, πρέπει να ξέρετε ότι είναι αρκετά πικρό, πικρή η τελική γεύση, διότι υπάρχει τελικά μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και λιγότερη στον ανθρωπισμό. Στα νότια σύνορα της Ένωσης βρίσκεται η Ισπανία ε, και το πακέτο για το άσυλο ε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το, ο κανονισμό του Δουβλίνου επίση είναι μπλοκαρισμένο στο Συμβούλιο. Αυτά μένουν να γίνουν από το επόμενο Κοινοβούλιο. Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ. για άλλη μια φορά θέλω να μεταφέρω την κραυγή αγωνίας των κατοίκων των νησιών του αιγαίου για τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές και κυρίως το μεγάλο αριθμό παρανόμων μεταναστών οι οποίοι εισραίουν στην ελλάδα. πρόσφατα έγινε και εκδήλωση διαμαρτυρίας στην σάμο γιατί πλέον οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. πιστεύω ότι ο ρόλος της frontex πρέπει να βελτιωθεί να μπορέσει πραγματικά να κάνει σοβαρή δουλειά στα θέματα που αφορούν την φύλαξη των συνόρων όχι μόνο στα θαλάσσια σύνορα γιατί βλέπουμε πλέον μεγάλη έλευση και από την μεριά των χερσαίων συνόρων την περιοχή του εύρου. επομένως εδώ πρέπει να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη βελτίωση της δουλειάς που κάνει η ίδια η frontex αλλά και στην περιοχή της Υπήρου, που υποτίθεται υπάρχει η frontex στα σύνορα ελλάδος αλβανίας και από εκεί έχουμε εισρωή κακοποιών